Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί τέος συνάδελφοι. Θα ήθελα επίσης ε, να καλωσορίσω και τους υπόλοιπους συναδέλφους που σιγά σιγά καταφθάνουν Ίσως το γεγονός ότι ήρθε πλέον ο χειμώνα να ευθύνεται για το γεγονός ότι δεν είμαστε πολύ στην αίθουσα αυτή τη στιγμή. Πάντως θα έπρεπε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας γιατί δεν έχουμε και απεριόριστο χρόνο στη διάθεσή μας. Εάν έχετε παρακολουθήσει το πρόγραμμά μας, θα γνωρίζετε ότι για τη δεύτερη ημερίδα της ακροασής μας σήμερα Έχουμε το πάνελ καταρχάς παριθμών 3 με συντονιστή τον Χέντρικ Κάφζακ από την Frankfurter Allgemeine Zeitung. Δεν είναι εδώ ο συντονιστής διότι χθες ένα τέταρτο πριν ξεκινήσει η χθεσινή μας συνεδρίαση μας είπε ότι δυστυχώς ε, υποφέρει και δεν μπορεί να μεταβεί στη συνεδρίαση. Είναι ασθενής. Εγώ βέβαια αντιλαμβάνομαι διαφορετικά τα πράγματα Νομίζω ότι το συγκεκριμένο άτομο δεν θέλει να είναι στο κοινοβούλιο γιατί έγραψε ένα άρθρο στο, ε, στη Frankfurt Allgemeine Zeitung που ήταν εχθρικό απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν νομίζω ότι θα το ήθελε και ιδιαίτερα να έρθει εδώ ε, έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι θέλει δηλαδή να εμφανιστεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά από όσα έγραψε. Τέλος πάντων δεν έγινε και κάτι. Έχουμε πάρα πολύ σημαντικούς προσκεκλημένους Έχουμε τον κύριο Όλμπριχτ, ο οποίος ε, θα αναλάβει ευχαρίστω το συντονισμό του πρώτου πάνελ. Το πάνελ το οποίο απαρτίζουν οι ε, Mercedes Μπρέσο, πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών, ο Φαμπρίτσιο Μπάρκα, που είναι Γενικός Διευθυντής στο Ιταλικό Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, και ο Εμίλ Ντίγκα, που είναι αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Ρωμανικού Ινστιτούτου Τραπεζών. Σας καλωσορίζω όλους και δίνω το λόγο στον Γιάνν ευθύ αμέσω ε, για να αναλάβει τον συντονισμό του πάνελ. Όπως και χθες θα ακούσουμε καταρχάς για πέντε λεπτά το συντονιστή, ο οποίος ε, θα κηρύξει την άρξη της συζήτησης. Ε, εν συνεχεία θα ακούσουμε για πέντε λεπτά ο καθέ, τον καθένα από τους ε, τρεις ομιλητές του πάνελ και στη συνέχεια οι συνάδελφοι βουλευτές θα έχουν τη δυνατότητα να θέσουν ερωτήσεις. Θα υπάρξει ένα ή δύο γύροι ερωτήσεων. Ξεκινάμε λοιπόν. Δεν κρύβω ότι ο συντονισμός ε, του πάνελ για μένα αποτελεί μεγάλη τιμή. Ακριβώς λόγω του ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά τα μέλη που απαρτίζουν το πάνελ σε ό,τι αφορά τη συνεργασία μας ε, για τις μελλοντικέ δημοσιονομικές προοπτικές στην πολιτική συνοχή που πρέπει να επεξεργαστούμε. Νομίζω ότι είμαστε η Επιτροπή η οποία επεξεργάζεται τις ε, προτεραιότητες για τη δημοσιονομική προοπτική. Δεν είμαστε δηλαδή μια Επιτροπή η οποία εξεργάζεται τα πάντα. Δηλαδή δεν ε, εξετάζουμε την πολιτική συνοχή ε, αυτή καθεαυτή, δηλαδή τι θα πρέπει να γίνει στο μέλλον. Έχουμε δύο ώρες στη διάθεσή μας. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα της Επιτροπής μας. Το πρόβλημα της Επιτροπής μας είναι που θα πρέπει να τεθούν οι προτεραιότητες. Και δεύτερον, ποιοι είναι, ποιος είναι ο αντίκτυπος, ποιες είναι οι επιπτώσεις για τον προϋπολογισμό τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο βέβαια και, των εθνικών ε, και στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Η Επιτροπή νομίζω ότι αντιμετωπίζει μια νέα πρόκληση διότι έχουμε σήμερα διαφορετικά έγγραφα τα οποία αποτελούν τη βάση των εργασιών μας σχετικά με τις προτεραιότητες. Πρώτα απ' όλα έχουμε το έγγραφο στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 αν δει κανεί αυτό το έγγραφο θα δει ότι υπάρχει ένας ε, κατάλογος προτεραιοτήτων που περιγράφεται. Σε αυτόν τον κατάλογο προτεραιοτήτων βλέπουμε ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση το σημαντικότερο στο μέλλον είναι η ανάπτυξη. Βέβαια αυτό το έγγραφο, η Στρατηγική 2020, θεσπίζει, εισάγει τρεις διαστάσεις ανάπτυξης. Ευφυή, βιώσιμη και ανάπτυξη για όλους. Και τα τρία αφορούν την ανάπτυξη. Δείχνει επίσης αυτό το έγγραφο ότι η πολιτική του χρόνου και από του χρόνου και μετά βέβαια θα πρέπει να βασίζεται στους τρεις αυτούς άξονες. Δεύτερον, αναθεώρηση του προπολογισμού. Αυτό το έγγραφο δεν αφορά μόνο τις προτεραιότητες, υπερβαίνει το πεδίο αυτό, αλλά μεταφράζει το έγγραφο αυτό σε προπολογισμό και ξέρετε ότι μετά την αναθεώρηση του προπολογισμού υπάρχει και πρόταση αλλαγής τη ίδια της δομή του προπολογισμού και προτείνεται οι προτεραιότητες τη στρατηγική 2020 να χρησιμοποιηθούν ως υποκατηγορίες, subheadings για τον προπολογισμό. Έχουμε λοιπόν αυτή την προσωρινή στρατηγική, η οποία θα αλλάξει ενδεχομένω τη δομή του προπολογισμού. Άρα, ίσω στην προσεχή στρατηγική να έχουμε ακόμη μια αλλαγή του προπολογισμού, τη δομή του, κάτι το οποίο είναι ενδιαφέρον. Καθιστά όμω τον προπολογισμό ιδιαίτερα ευέλικτο και ιδιαίτερα πολιτικό στη φύση του. Βλέποντα λοιπόν τα συμπεράσματα από την αναθεώρηση του προπολογισμού, είναι ξεκάθαρο ότι η πρόταση είναι οι φυστάμενες πολιτικές, της συνθήκης, όπως τις αποκαλούμε, να μπουν σε κάποια κουτιά, σε κουτιά προτεραιοτήτων. Πρώτο κουτί, καινοτομία. Διευρωπαϊκά δίκτυα. Κοινή γεωρική πολιτική και κλιματική αλλαγή, δεύτερο κουτί. Τρίτο κουτί, πολιτική συνοχής. Το για όλους δηλαδή. Άρα η πολιτική συνοχή θα είναι, πλέ, θα στο ένα τμήμα της ανάπτυξης για όλους. Και αυτό πρέπει να το πω ευθύ εξ αρχή Δεν συνάδει απόλυτα με τη στρατηγική 2020, διότι μιλάμε για ανάπτυξη για όλους στην στρατηγική 2020, αλλά είναι κοινωνικό πιο πολύ. Ενώ στην άλλη περίπτωση ε, αυτός ο όρος μπορεί να περιλαμβάνει τα πάντα και όχι μόνο την κοινωνική πολιτική. Επομένως, Ποιο είναι το συμπέρασμα, τι θα πρέπει να κάνουμε στο μέλλον με τι δημοσιονομικέ προοπτικές, πώ θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τι προτεραιότητε, πώ θα πρέπει να αντιληφθούμε ε, την κατάρτιση του προπολογισμού. Αυτό θα ήθελα να ακούσω από το πάνελ. Μεταξύ άλλων, θέλω να ρωτήσω το εξή στου ομιλητέ μα. Πώ εννοείται την ανάπτυξη για όλου, Τι θα πει, πώ εννοεί η συνθήκη τον όρο ανάπτυξη για όλου και πώ αυτό ο όρος μπορεί να μεταφραστεί σε συγκεκριμένα στοιχεία του προπολογισμού. Διότι αν αυτό δεν το εξηγήσουμε αυτής εξ αρχής, ενδέχεται να προβαίνουμε από εδώ και πέρα σε επανερμηνίες της στρατηγικής 2020, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε έναν προϋπολογισμό. Είναι ενδιαφέρον το εγχείρημα, αλλά πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Αυτό το οποίο προτείνω είναι στο τέλος να απαντηθεί το εξής ερώτημα. Θα πρέπει η πολιτική συνοχής να θεωρείται κάτι το οποίο απλά βάζουμε στο κουτί της ανάπτυξης για όλους. Αυτό το αφήνω έτσι ως ανοιχτό ερώτημα. Ξεκινήσουμε λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν με τους ομιλητές μας. Πρώτη ομιλήτρια είναι η πρόεδρος Επιτροπής των Περιφερειών, η κυρία Μερσέδες Μπρέσο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ε, ε, ευχαριστώ. Ε, καταρχήν επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω ε, τον, την Πρόεδρο που μας ε, προσκάλεσε σε αυτήν την ακρόαση για την ε, στρατηγική της Ευρώπης για το 2020 και το μελλοντικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτήν την ειδική επιτροπή για τις πολιτικές προκλήσεις. Και εμείς ως Επιτροπή έχουμε συστήσει μια ειδική επιτροπή για τον προϋπολογισμό της Ένωσης και κατεργαζόμαστε μία πρόταση. Το 2011 θα εξετάσουμε και το πολιετές δημοσιονομικό ε, πρόγραμμα για αυτό το ζήτημα των πόρων, που είναι ζήτημα ουσίας. Θα ήθελα να υπάρχει ένας μόνιμος διάλογος με τη δική σας Επιτροπή από εδώ και στο εξής, και να διαμορφώσουμε κάποιους ε, τρόπους κοινή εργασίας, ανταλλαγής εγγράφων, ανταλλαγής ε, απόψεων. Μπορούμε, πιστεύω, να συνεργαστούμε και να επεξεργαστούμε και να δούμε τις προτάσεις που έρχονται στο τραπέζι. Τώρα, για το θέμα της ε, διάρκειας του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, η Επιτροπή πρότεινε ήδη το 2008 ένα μοντέλο 5 συν 5, το οποίο καλά λειτουργεί από ό,τι βλέπουμε και επιτρέπει να έχουμε έναν πιο μακροχρόνιο προγραμματισμό και να προσαρμοζόμαστε σε αυτές τις πολύ πλατιές, ευρείες στρατηγικές όπως η στρατηγική της Ευρώπης το 2020 αλλά μας επιτρέπει επίσης η εργασία αυτή να προσεγγίζουμε και πιο πλατιά θέματα για τη στρατηγική 2020, για το δημοσιονομικό μηχανισμό και τους νέους μηχανισμούς, νομίζω τα τρία αυτά θέματα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ενός κοινού ε, προγραμματισμού. Ως φορολογικές αρχές, πολλές κοινότητες και δήμοι καλούνται να συμμετέχουν στη μεταρρύθμιση των ε, πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα καταρχήν να εκφράσω την πλήρη υποστήριξη της Επιτροπής μας στον αγώνα που έχει ξεκινήσει το Κοινοβούλιο για να προάγει τις νέες στρατηγικές του και προτεραιότητές του στο πλαίσιο της συνθήκης της Λισαβόνας. Τώρα, για τη στρατηγική του 2000, για το 2020, θα ήθελα, μάλλον όπως το θύμισε η προλαλή σας, θέλουμε μια ανάπτυξη η οποία να καθορίσει με σαφήνεια τους δεσμούς της με τις άλλες πολιτικές, να ενταχθεί στις άλλες πολιτικές. Κατά την άποψή μας, αυτό το θέμα της ε, ανάπτυξη σε τρία επίπεδα μπορεί να θεμελιωθεί και σε μια διακυβέρνηση σε πολλά επίπεδα, στην ε, κοινότητα, στα κράτη-μέλη και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πριν να επισέλθω στα ειδικότερα θέματα, θα ήθελα να σας εκφράσω ορισμένα βασικά πολιτικά ζητήματα. Καταρχήν να υπενθυμίσω ότι η, κοινή, η τοπική αυτοδιοίκηση ε, υλοποιούν και απορροφούν το 60% των πόρων της κοινότητας. Πρόκειται για, για δημόσιες δαπάνες ποιότητας σε στενή σύνδεση με τις ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις που γίνονται ε, στις περιφέρειες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική το 2020 δεν θα μπορέσει να υλοποιηθεί αν δεν αποκτήσει και δικούς της πόρους, αν η τοπική αυτοδίκηση και τα κράτη-μέλη δεν έχουν και δικούς τους πόρους και αν δεν είναι μια στρατηγική που να τη συμμερίζονται όλα τα επίπεδα αλλά και όλοι, όλοι οι προϋπολογισμοί. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ε, προσανατολισμός στρατηγική η πρόταση που έκανε, που γίνεται μέσα από την ε, συνεργασία για την σωστή ανάπτυξη πρέπει να ανοίξει σε τοπικές συμφωνίες μεταξύ αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης, δομών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το κράτος θα πρέπει να καθορίσει μια σύμβαση, μια συμφωνία, αλλά θα πρέπει η συμφωνία αυτή, η σύμβαση αυτή να υλοποιείται σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Επιτροπής και κρατών μελών δεν αρκούν, γιατί επαναλαμβάνω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι εκείνη που υλοποιεί το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων. Τρίτον, ο προϋπολογισμός του 1% του εκαθάριστου εγχώριου προϊόντος δεν μπορεί να υπηρετήσει όλες τις λειτουργίες. Διαρθρωτικές επενδύσεις για την ανάπτυξη, ε, μάχη κατά της συγκυρίας, μηχανισμός ευελιξίας για την ανταπόκριση στις έκτατες καταστάσεις. Μου φαίνεται αδύνατο οι νέες λύσεις απέναντι στις δαπάνες και στην οικονομική διακυβέρνηση είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να προωθήσουμε. Πρέπει επίσης να έχουμε το ευρωομόλογο για να μπορούμε να χρηματοδοτούμε μεγάλης κλίμακας έργα που να αποφέρουν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Χωρίς αυτή τη δυνατότητα θα συμβεί αυτό που συμβαίνει μέχρι τώρα. Τα μεγάλα δίκτυα των μεταφορών προγραμματίζονται και διακηρύσσονται αλλά ποτέ δεν υλοποιούνται γιατί δεν έχουν στα μέσα, τα μέσα που χρειάζεται δεν έχουν στα χέρια τους τα κράτη-μέλη τα μέσα που χρειάζονται. Χρειάζονται και πολλές άλλες επενδύσεις και πρέπει οι επενδύσεις αυτές να μπορούν να έχουν και αποδόσεις, αποδόσεις ίσως πιο μακροπρόθεσμες. Έτσι λοιπόν αυτά τα ευρωπαϊκά ομόλογα που θα μπορούν να υπηρετούν αυτή τη μακροπρόθεσμη απόδοση των επενδύσεων μας φαίνεται ένας πολύ σημαντικός μηχανισμός. Το θέμα των ίδιων πόρων είναι ένα θεμελιώδες ζήτημα. Η Επιτροπή δεν έχει κάποιες προκαθορισμένες ιδέες στο μυαλό της σε σχέση με τους έξι μεγάλους προσανατολισμούς. Μου έρχεται στο νου και η επίπτωση των, ε, η μελέτη των επιπτώσεων. Ε, πρέπει να προχωρήσουμε και στην πράσινη ανάπτυξη, αρκεί οι πόροι που θα συγκεντρωθούν θα μπορούν να διοχετευθούν κατευθείαν στην τοπική αυτοδιοίκηση έτσι ώστε να επιτύχουμε την πρόληψη και την παρέμβαση σε, σε, περίπτωση σημαντικών καταστροφών. Υπάρχουν όλα τα προγράμματα που έχουν να κάνουν με την πράσινη διάσταση, αλλά ε, ε, οι επενδύσεις αυτές έχουν ε, εξαρτώνται έντονα και από τις πολιτικές επιλογές. Παράδειγμα, η περίφημη ενίσχυση των δημοσιονομικών μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Ταμείου αλληλεγγύης. Αυτό μας δείχνει πως οι αποφάσεις για τον προϋπολογισμό που θα λάβουμε θα έχουν τεράστιο αντίκτυπο για τη ζωή των πολιτών μας, αλλά και για το πώς βλέπουν την, προσ... την, την προστιθέμενη οικονομική αξία που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκβαση αυτών των πολιτικών θα μας δείξουν κατά πόσο θα είμαστε ικανοί να υλοποιήσουμε τις στρατηγικές της Λισαβόνας, δηλαδή πολιτικές που να έχουν ρίζες στο ε, έδαφος των κρατών μελών, που να έχουν σημασία για τον Ευρωπαίο πολίτη, που να είναι ευρύτερη ανάπτυξης κτλ. Αυτές ήταν κάποιες πρώτες δηλώσεις που είχα να κάνω και θα προσπαθήσω στη συνέχεια να υπησέλθω στο θέμα ε, που μου έθεσε η συντονίστρια αυτό που με έθεσε ο συντονιστή. με συγχωρείτε, για τις τρεις διαστάσεις της ανάπτυξης που προτείνει η στρατηγική της Ευρώπης για το 2020 και τις διάφορες πολιτικές. Ε, νομίζω ότι είναι δυνατό αυτό, αλλά είναι δυνατόν μόνο μέσω των, του συστήματος των συμβωνιών, των συμβάσεων. Αρκεί αυτές να έχουν ως αφετηρία μία δέσμευση σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης της Υπήρου μας. Αν όλοι μαζί από κοινού επικεντρωθούμε στις τρεις διαστάσεις της ανάπτυξης, που έχουν διαφορετικές πτυχές και διαφορετικά εργαλεία βέβαια, αλλά που ασφαλώς μπορεί, μπορούν να τη συμμεριστούν όλοι, τότε θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε να ε, υλοποιήσουμε ταυτόχρονα να πραγματοποιήσουμε ένα άλμα προς τα εμπρός στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Υπήρου, αλλά και να το κάνουμε λαμβάνοντας υπόψη και άλλους στόχους. Ε, τη συμπερίληψη όλων, την ένταξη όλων, την σύγκληση όλων των ε, περιφερειών και περιοχών μας προς αποδεκτά επίπεδα εισοδήματος και ποιότητας ζωής. Μια έντονη αύξηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, αειφορίας, ασφαλώς είναι ένα ζήτημα που επιτρέπει ανάπτυξη και μεγέθυνση ε, που να είναι βιώσιμες για τις περιοχές και τις περιφέρειες και που να την χάνουν και σωστής διαχείρισης. Και σίγουρα η έξυπνη ανάπτυξη που θα βασίζεται στην τεχνολογία των πληροφοριών παρέχει μεγάλες δυνατότητες και ανάπτυξης και παραγωγής και μεγέθυνσης. Έτσι λοιπόν ευθύς εξ αρχής ε, διαφαίνεται ένα ζήτημα, ε, ένα θέμα διακυβέρνησης εν τη πράξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Βέβαια εγώ ε, το ερώτημα που έκανα δεν αφορούσε τίτλους ή ονόματα αλλά τις συνέπειες, επιπτώσεις. Δηλαδή όταν κάτι το συμπεριλαμβάνουμε στον προϋπολογισμό έχουμε τις επιπτώσεις του είδους των επενδύσεων που μπορεί να γίνουν με τον τάδε τον δίνω προπολογισμό. Δηλαδή δεν είναι θεωρητικό το εγχείρημα γιατί μιλάμε για τις επιπτώσεις. Χθες, στο πρώτο πάνελ, ένας από τους ομιλητές είπε ότι δεν θα πρέπει να συγχέουμε την ανταγωνιστικότητα με τη συνοχή. Και ότι ευφυής ανάπτυξη ουσιαστικά σημαίνει αριστεία και ανάπτυξη της καινοτομίας. Ήταν ξεκάθαρο λοιπόν ε, και ήταν και παραδοσιακό τρόπο σκέψη για την ε, συνοχή. Πάντω το είπαν χθε οι του πάνελ. Τώρα λοιπόν προχωρούμε. Και από την πλευρά των εφιών ε, ομιλητών, αν μπορώ να του χαρακτήσω έτσι, του πάνελ, είχαμε μία, ένα διχασμό. Τώρα να περάσουμε στον επόμενο ομιλητή, τον Φαμπρίτσιο Μπάρτσα, να απαντήσει. Ευχαριστώ. Διάβασα το πολύ ενδιαφέρον εγγραφό σα και όντω θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη πρόκληση. Θα προσπαθήσω να απαντήσω. Θα κάνω έτσι μια γενική ε, παρουσίαση και θα κάνω και κάποια σχόλια. Το πώ έχουν τα πράγματα είναι απλό. Οι προκλήσει ζητούν καλύτερη χρήση του προπολογισμού και πιο ισχυρή αναπτυξιακή πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πολιτική συνοχή ω έχει ε, και όπω την ορίζει η ε, συνθήκη, η εδαφική, η πολιτική, η οικονομική, μπορεί να μας πάει μπροστά, εφόσον βεβαίως αυτή μεταρρυθμιστεί για να μπορέσει να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά της. Η Κομισιόν ε, έχει υποβάλει μια μεγάλη μεταρρύθμιση για την πολιτική συνοχή με βάση τρεις πτυχές. Θα τις ε, αναφέρω, ε, συγκέντρωση, αιρεσιμότητα και μετρήσιμη στόχη. Μπορώ αν θέλετε να σας πω ποια είναι η άποψή μου, αλλά δεν θέλω να, τα, να πω σε λεπτομέρειες. Αυτό έχουμε τώρα επιτάπητος. Αυτά είναι τώρα τα τρία μηνύματα. Πρώτο μήνυμα. Η πολιτική συνοχή και οι στόχοι της θα πρέπει, αντίθετα με αυτά που άκουσα μόλι, να ε, διευρυνθεί και πέρα από την ανάπτυξη και να ε, καλύψει και τους πέντε στόχους. Πέντε στόχους. Οι πέντε στόχοι οι τρεις βασικοί στόχοι της ε, πολιτικής του 2020 θα πρέπει να προωθηθούν. Τι είναι η πολιτική του 2020? Πρέπει να είναι πλήρως συνεκτική και ανεξάρτητη από την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού που βασίζεται στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων για το 2020. Όλα αυτά καλά ισχύουν, αλλά θα ήμουν ε, προθύστερο εάν δεν έλεγα ότι αυτή η πολιτική, αυτή μεταρρύθμιση πρέπει να προχωρήσει. Η πολιτική συνοχή ε, δεν είναι όπω είναι σήμερα. Μιλούμε για την πολιτική συνοχή όπω αυτή θα μεταρρυθμιστεί. Ξε, ξεχάστε το ότι πρέπει να είναι έξυπνη και περιληπτική κτλ. Δεν θέλουμε να ακούμε τέτοια σλόγγαν. Ε, δεν θέλουμε όμως να ακούμε και για τον προπολογισμό. Ο προπολογισμός είναι κάτι ε, σημαντικό. Αυτοί οι πέντε λοιπόν στόχοι που έχει, θώσει, που έχει θέσει το Συμβούλιο είναι πολύ συγκεκριμένοι. Ε, δεν θα τους επαναλάβω, τους ξέρετε. Πέντε συγκεκριμένοι στόχοι που υπάρχουν. Για, κάποια, για, κάθε από αυτή, για, κάθε, για κάθε έναν από αυτούς τους στόχους η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμφωνήσει για κάποιες βασικές, κάποιους βασικούς ε, στόχους με τα κράτη-μέλη που λένε να ότι θέλουν να δημιουργήσουν δικού τους, δικούς τους ε, εθνικούς στόχους. Όλοι αυτοί οι στόχοι όμως πρέπει και μπορούν να προωθηθούν από την πολιτική συνοχή. Η πολιτική συνοχή θεωρείται και κοινωνική ε, συμπερίληψη και ανταγωνιστικότητα. Γιατί η πολιτική συνοχή θέλει να εξασφαλίσει ότι όλε οι περιφέρειε μπορούν να έχουν την ευκαιρία να αναπτυχθούν. Αυτό σημαίνει ότι θα, είναι, ότι θα συμπεριλαμβάνουν όλου του πολίτε με ένα συγκεκριμένο επίπεδο διαβίωση και θα έχουν την μέγιστη δυνατή ανάπτυξη. Η πολιτική συνοχή λοιπόν θα πρέπει να διατηρήσει τον ξεχωριστό τίτλο τη στον προπολογισμό. Δεν υπάρχει αμφιβολία περί αυτού. Το να μην υπάρχει θεματική προτεραιότητα σχετική με την ανάπτυξη θα πρέπει να αποκλειστεί. Ούτε καν για τις βασικές υποδομές. Οι βασικές υποδομές αφορούν την, ε, την απάλληψη των αδιεξόδων που έχουμε βρεθεί. Χρειαζόμαστε λοιπόν με ένα τέτοιο διευρωπαϊκό δίκτυο για παράδειγμα γιατί μειώνει την τιμή αναμονάδα για τις, και για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις. Είναι λοιπόν σημαντικό κομμάτι της πολιτικής 2020 η πολιτική για το 2020 θα καταφέρει να τα συγκεράσει όλα αυτά. Αυτό που μας δίνει η Κομισιόν ως απάντηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Η συγκέντρωση δεν είναι κάτι που σημαίνει ότι κάποιος της Βρυξέλλες αποφασίζει για την άλλη άκρη της Ευρώπης ποιος θα κάνει κάτι. Είναι ότι μια περιφέρεια της Ευρώπης μπορεί να αποφασίσει για τον εαυτό της. Αν θέλετε να τα συμπεριλάβετε όλα, τα συμπεριλαμβάνετε όλα. Αν θέλετε να επικεντρωθείτε στην ανταγωνιστικότητα, επικεντρώνεστε στην ανταγωνιστικότητα. Δεύτερον, η προστιθέμενη αξία της πολιτικής συνοχής η πολιτική συνοχή έχει ένα πλεονέκτημα έναντι τη ανοιχτή μεθόδου συντονισμού. Μάλιστα έχει τέσσερα πλεονεκτήματα. Πρώτον, μπορεί να συμπεριλάβει και στην Κομισιόν και στα κρατη μεταξύ διάφορων ε, πολιτικών τομεακών ε, όλα τα στοιχεία, καθώς και όλα τα στοιχεία μεταξύ διαφόρων, ε, πολιτικών, διαφόρων ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, οι διαρθρωτικές αλλαγέ και οι θεσμικές προσαρμογές που χρειάζονται σε κάθε κράτο μέλο και περιφέρεια για δράσεις πολιτική και για να είναι αυτές αποτελεσματικέ. Στην περίπτωση της πολιτικής συνοχής, δεν είναι απλώς ρητορικές πολιτικές δεσμεύσεις. Μπορούν μαζί με τις μεταρρυθμίσεις, εάν γίνουν οι μεταρρυθμίσεις, να γίνουν δεσμευτικές ε, Εσεί θα, θα το ε, αποφασίζετε, Εσεί τα κρατημέλη, όχι οι Βρυξέλλε. Αν δεν γίνουν αυτέ οι προσαρμογέ, τότε εμεί δεν θα σα δώσουμε τα χρήματα για το συγκεκριμένο ε, project, γιατί δεν έχετε τις ε, προποθέσει που πρέπει να πληρούνται. Τρίτο, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βασιστεί ε, στου ανθρώπινου ανθρώπινους πόρους που είναι βασικοί, και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βασιστεί σε έναν συντονισμό ε, εδαφικών αρμοδιοτήτων, Γενική Διεύθυνση αλληλεία, Περιφερειών κτλ. Όλοι αυτοί λοιπόν μπορούν να συνεργαστούν όπως προτείνει η Κομισιόν και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί έτσι μπορούμε να ενώσουμε και τις τομεακές γενικές ε, και τέλος ε, στη μεταρρύθμιση ένα σύστημα δικτών και στόχων υπάρχει και δεν επιβάλλεται από πάνω προς τα κάτω, αλλά ε, ορίζεται όπως το χρειάζονται οι περιφέρειες και ε, καθοδηγείται από μια ενισχυμένη κομισιόν που θα εξασφαλίσει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι πολίτες, τα ΜΜΕ ε, θα λαμβάνουν τα συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία, θα λαμβάνουν τα αποτελέσματα ε, που είναι σημαντικά για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε λοιπόν και έναν πίνακα, δεν θα τον ε, αναφέρω τώρα έτσι λεπτομερώς, αν θέλετε μπορούμε να επανέλθουμε, αλλά κατά την άποψή μου, εδώ μιλούμε για τη σχέση μεταξύ των διαδικασιών εθνικών προγραμμάτων και της πολιτικής συνοχής είναι μια σχέση συνεκτική και όχι εξάρτησης του ενός από το άλλο. Ένα λεπτό αν έχω πρόεδρε. Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Στην ε, προηγούμενη διαπραγμάτευση έγιναν κάποιες ε, προσπάθειες για να μεταρρυθμιστεί η πολιτική συνοχή, οι οποίες όμως δεν πέρασαν ακόμη και από τα μεγάλα κρατημέλη που συνέβαλαν προτίμησαν τελικά να αρνηθούν τις μεγάλες εγγύησεις που θα ήθελαν τα υπόλοιπα κρατημέλη, όχι η μόνιμη σύνηθεση υποπτή, οι νότιες χώρες, ανατολικές κλπ. Αλλά αρνήθηκαν να δώσουν τις ε, εγγύησεις αυτά τα ίδια τα κρατημέλη, τα μεγάλα και έτσι ε, δεν πέρασαν οι μεταρρυθμίσεις. Κάποιοι κρατημέλοι έλεγαν και τότε και λένε και σήμερα ότι ξέρουν πολύ καλύτερα πώς ε, εκπονείται η, ε, η πολιτική συνοχή. Δεν χρειάζονται ούτε ιδέες, ούτε καθοδήγηση από τις ε, Βρυξέλλες και μετά έρχονται εκλογέ. Αλλάζουν οι ε, κυβερνήσεις, κοιτάμε την ίδια χώρα, η, την επόμενη μέρα η πολιτική συνοχή τη ίδια χώρα έχει αλλάξει τελείω. Ναι, αλλά μήπω αν είχατε συζητήσει αυτή την πολιτική με τι Βρυξέλλε να, να ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Τέλο λοιπόν, Πρόεδρε, για τρίτη φορά, ε, νομίζω ότι Τώρα πια είναι, ο, είναι η χρονική στιγμή σωστή για να περάσει η μεταρρύθμιση και όλα αυτά τα πράγματα που έχω πει για την πολιτική συνοχή θα μπορούσα να τα, τα αποσύρω αμέσω εάν ε, ε, η πολιτική συνοχή δεν περνούσε όπως ε, θα έπρεπε. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το βήμα που μπορεί να ελέγξει καλύτερα την εφαρμογή και το σχεδιασμό της μεταρρύθμισης, έτσι ώστε να ξέρουμε ότι αυτό που, θα, που λέμε τώρα θεωρητικά θα γίνει κάποια στιγμή και πράξη. Θέλω να ρωτήσω το εξή. Τι γίνεται με τις τράπεζες, πώς αντιλαμβάνονται την όλη διαδικασία οι τραπεζίτες. Ας δώσω όμως το λόγο στον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του Ρωμανικού Ινστιτούτου Τραπεζών, Εμίλ Ντίγκα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Για να δώσω ένα πιο σαφές μήνυμα, θα με επιτρέψετε να μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα, τα ρουμανικά. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το ερώτημα που έθεσε ο κύριος Όλμπριχτ, ο συντονιστής, Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα και η ομιλία μου την οποία έχετε και μπροστά σας αλλά η οποία και θα ακουστεί μέσω του διαδικτύου θα επικεντρωθεί ακριβώς αυτό το ζήτημα. Κατά την άποψή μου η συνοχή είναι ένα κοινωνικό θέμα, κοινωνικό ζήτημα και έτσι θα πρέπει να παραμείνει. το μέσο επίτευξης του στόχου της συνοχής είναι οικονομικού χαρακτήρα. Και για να είμαστε βέβαιοι ότι θα επιτευχθούν οι κοινωνικοί στόχοι, πρέπει να έχουμε οικονομικούς πόρους, οικονομικά μέσα. Και κατά την άποψή μου το μέσο είναι η βιωσιμότητα της ανάπτυξης, η διάρκεια της ανάπτυξης. Θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η στρατηγική για την Ευρώπη 2020 εξασφαλίζει την ανάπτυξη σε διάφορους στόχους, αλλά χωρίς να κάνει συγκεκριμένα λόγο για την βιωσιμότητα, τη διάρκεια των στόχων αυτών. Και θα ήθελα να ξεκινήσω μιλώντας για την αρχή flexicurity, ευελιξία με ασφάλεια. Εγώ θα αντικαθιστούσα τον όρο αυτό με τον όρο sus cohesion, sustainability and cohesion, δηλαδή βιωσιμότητα και συνοχή, βιωσιμοσυνοχή. Τι μπορεί να εξασφαλίσει τον όρο αυτό, η συνοχή θα πρέπει να τροφοδοτεί τη βιωσιμότητα. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεύτερο, αναφέρθηκε ένα άλλο πρόβλημα οι τρεις στόχοι της πολιτικής συνοχής όσοι έχει τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διατηρηθούν. Πρέπει ή δεν πρέπει. Η σύγκληση, η ανταγωνιστικότητα, η απασχόληση αλλά και η εδαφική συνεργασία. Στόχοι που κατά την άποψή μου δεν είναι ομοιογενείς. Η σύγκληση ουσιαστικά συνεπάγεται τους άλλους δύο τους άλλους δύο άξονες θα έλεγα. Με συνέπεια, οι στόχοι της πολιτικής συνοχής να πρέπει να είναι ανεξαρτητή ο ένας από τον άλλον, να μην αντιφάσκει ο ένας με τον άλλο, αλλά και να αλληλοσυμπληρώνονται, ανά δύο. Άρα, οι τρεις στόχοι της πολιτικής συνοχής κατ' εμέ, θα έπρεπε να είναι η εξή. Πρώτα απ' όλα, σύγκληση, οικονομική, εδαφική και κοινωνική, φυσικά. Παραγωγικότητα, που δεν προβλέπεται στη Στρατηγική Ευρώπη 2020 και η οποία όμως εξασφαλίζει την διάρκεια για την οποία έκανα λόγο προηγουμένως και βέβαια διάρκεια βιωσιμότητα. Από αυτήν την έννοια και σε συνάρτηση και σχέση με όλα αυτά πιστεύω ότι θα μπορούσε στο μέλλον να γίνει μια αλλαγή σε σχέση με την πολιτική συνοχής. Τι εννοώ. Η πολιτική συνοχής θα έπρεπε να επικεντρωθεί, θα έλεγα, στην παραγωγικότητα. Και γιατί το λέγω αυτό. Διότι από μόνη της η απασχόληση, ο στόχος απασχόληση της στρατηγικής 2020 από μόνος του δεν αρκεί. Μπορούμε να έχουμε ψηλά ποσοστά απασχόλησης, αλλά μειωμένη παραγωγικότητα. Εγώ νομίζω ότι η πολιτική στον πληθυντικό θα πρέπει να έχουν στατιστικά στοιχεία ή δείκτες που θα δείχνουν και την απασχόληση και την παραγωγικότητα. Και έχω μία υπόδειξη να διατυπώσω. Θα μπορούσε αυτό να είναι ο λόγος, η αναλογία ΑΕΠ προς τον πληθυσμό 25 με 64. Πρόκειται για ένα δίκτυ που ουσιαστικά είναι ποσοστό απασχόλησης, ποσοστό παραγωγικότητας. Σύνθετος δείκτης. Έτσι θα μπορούσε η πολιτική της ανάπτυξης ή της απασχόλησης μάλλον να γίνει και ουσιαστικά πολιτική συνοχής. Τώρα, ένα άλλο θέμα το οποίο έχει να κάνει με τον προπολογισμό, με τη δομή του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Όλοι γνωρίζουμε την έκθεση Λαμασού. Γνωρίζουμε επίσης ότι αυτή τη στιγμή γίνονται συζητήσεις σε σχέση με το σύστημα των ιδίων πόρων. Ίσως θα μπορούσε να συγκροτηθεί μια ομάδα εργασίας που θα καθορίσει ένα κοινό, μια κοινή φορολογική βάση ε, που δεν θα έχει διακυμάνσεις από κράτος σε κράτος, που θα είναι παρατηρήσιμη, μετρήσιμη και που θα είναι σε συνάρτηση του βαθμού με τον οποίο ένα κράτος μέλος ωφελείται από την ολοκλήρωση. Και αυτό το ποσοστό, αυτός ο βαθμός θα πρέπει να ε, να καθορίζει και τα ποσοστά του κάθε κράτου στον προϋπολογισμό. Στην πρόταση που έχουμε λάβει γίνεται λόγος επίσης για τις συνέργειες μεταξύ της στρατηγικής 2020 και των εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων. Έχω μια πρόταση. Θα μπορούσαμε ίσως να υπολογίσουμε τη συμμετοχή των κρατών μελών τη συμμετοχή τους στην εκπλήρωση των στόχων 2020, προσαρμόζοντας την ισοδύναμη αυτή αντίστοιχη συμμετοχή με τους εθνικούς στόχους. Οπότε θα μπορούσαν να υπάρχουν περισσότερα κίνητρα για τα κράτη-μέλη να λάβουν μέρος σε στρατηγική 2020. Και τέλος θα ήθελα να αναφέρω κάτι το οποίο προβλέπεται και στη στρατηγική 2020. Καμιά ευρωπαϊκή πολιτική δεν θα πρέπει να υλοποιείται αν δεν λαμβάνει υπόψη του στόχου της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Θα πρέπει να είναι δηλαδή ένα master plan, ένα γενικό σχέδιο η στρατηγική 2020. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα. αν θα πρέπει ο προπολογισμό κατά 100% να αφοσιωθεί στους στόχους της στρατηγική 2020. Ε, ε, και η απάντησή μου είναι ναι, είναι καταφατική η απάντησή μου. Και θα πρέπει να δούμε ίσως και το επίπεδο ΝΑΤΣ που θα έπρεπε να αποδώσουμε για κάποιες μακροπεριφέρειες. ίσως το επίπεδο νάτς 0 για τις μακροπεριφέρειες. Δηλαδή κάποιες υπερεθνικές περιφέρειες που είναι μοχλή της διαδικασίας συνοχής. Και βέβαια όποιος θέλει λεπτομέρειες ευχαριστώ να δώσω περισσότερα στοιχεία στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Ο συντονιστής. Βλέπουμε μετά και τους τρεις ομιλητές που ακούσαμε ότι έχουμε διαφορετικά επίπεδα στη συζήτηση. Το ένα επίπεδο αφορά τη θέση της ε, ούτω λεγόμενης πολιτικής συνοχής στις ευρωπαϊκές πολιτικές και πώς θα πρέπει αυτή να αντικατοπτρίζεται στον προπολογισμό. Και βέβαια το θέμα είναι ε, ποια θα είναι η σχέση και με τη στρατηγική 2020. Δεύτερος άξονας, μέθοδος. Μπορούμε να τη διαχωρίσουμε βέβαια, αλλά όταν λέμε μέθοδο εννοούμε μεταρρύθμιση. Αυτό που ο κύριος Μπάρκα είπε ότι η μέθοδος ε, ίσως είναι η αλλαγή, ε, μάλλον η αλλαγή της πολιτικής βασίζεται ε, στη μέθοδο. Ότι θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή στη μεθοδολογία. Τώρα λοιπόν μπορούμε να κάνουμε τις ερωτήσεις μας. Έχουμε λίγο πολύ 20 λεπτά για τη συζήτηση και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. ich schon eine Liste. Έχω έναν σύντομο κατάλογο. Ευχαριστώ. Δύο ερωτήματα και μία παρατήρηση. Να ευχαριστήσω τον Φαμπρίτσιο Μπάρκα που έτσι σαφέστατα μας ανέφερε την ανάπτυξη που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και θα πρέπει να, συμμετέχει, να συμμετέχουν όλοι που συνδέεται με την πολιτική συνοχή. Εγώ είμαι εισηγήτρια για την Επιτροπή Περιφερειών για, την, για το θέμα αυτό και θα ήθελα να μου δώσει μια σύσταση για το πώς μπορώ εγώ να καταστήσω σαφές ότι αυτές, αυτά τα τρία σλόγγαν είναι τελείως ανόητα για να τα χρησιμοποιούμε γιατί πραγματικά προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν μέσω αυτών των ε, σλόγγαν να ε, ανεξαρτητοποιήσουν ας πούμε τον ε, ε για την ε, πολιτική συνοχή, να τον αυξήσουν, κάτι που αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει. Επίσης, ε, για την κυρία Μπρέσο. Έχουμε την εντύπωση ότι θα υπάρξει, θα πρέπει να υπάρξει τουλάχιστον μια εφταετία για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές και για τις περιφέρειες και έχοντα υπόψη αυτό και έχοντα υπόψη ότι έχουμε τη στρατηγική τη Λισαβόνα την οποία θεωρήσαμε κάποια στιγμή και ως ε, τελείως ε, ε, αποτυχημένη και το 2014 θα έχουμε νέα πολιτική συνοχής και έχουμε και την στρατηγική 2020 αν θέλουμε να, το, ε, να χωρίσουμε μόνο τις, ε, το, την περίοδο αυτή μόνο σε δύο πενταετίες, τότε ε, το πρόγραμμα θα είναι, θα είναι δύσκολο να προχωρήσει. Ίσως λοιπόν αυτά τα δύο, τα, οι δύο πενταετίες να μην είναι η απόλυτη, απόλυτα σωστή περίοδος. Και επίσης, βιωσιμότητα για την πολιτική συνοχής και ανταγωνιστικότητα. Νομίζω ότι αυτό το θέμα είναι πολύ ευρύ και δεν μπορούμε να το συζητήσουμε εντελεχώ σήμερα. Ευχαριστώ. Η Χέλγκα, παρακαλώ. Ε, um, Ευχαριστώ, Γιούτα. Θα επανέλθω στο έγγραφο που μας έδωσε ο κύριος Μπάρκα, γιατί είπε ότι Ίσως ε, το έξυπνο, ε, βιώσιμο και συμπεριληπτικό ε, θα πρέπει να, δούμε, να το δούμε μέσα από τους πέντε βασικούς στόχους που ήδη έχουν ξεκινήσει και συμφωνηθεί. Ο πρώτος είναι η βελτίωση των συνθηκών για την καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη και βελτίωση της, ε, των επιπέδων εκπαίδευσης. Τρίτον, συμφω... Ε, ε, ε τους στόχους για την ενέργεια και την στρατηγική της και την κλιματική αλλαγή. Υπάρχει όμως μεγάλη σύνδεση εδώ μεταξύ καινοτομία και ε, χαμηλής, οικονομία χαμηλού άνθρακα ή οικονομία χωρίς καθόλου άνθρακα γιατί αυτό είναι κομμάτι ε, των όλων των προγραμμάτων μας. Οπότε, κατά την άποψή μου, είναι σημαντικό εδώ να συνδέσουμε τη βιωσιμότητα με την κλιματική αλλαγή και την καινοτομία. Γιατί αν πάμε σε, ένα άλλο είδους, σε μια άλλου είδους καινοτομία, χωρίς να έχει πτυχή ε, κλιματική, τότε θα έχουμε πρόβλημα. Γιατί ε, στην στρατηγική της Λισαβόνας δεν υπάρχουν σαφείς σύνδεσμοι και εν τω μεταξύ θεωρώ ότι έχουμε προχωρήσει. Φυσικά λοιπόν πρέπει να συνδέσουμε τους στόχους για το κλίμα με, τα, με, τα δικά μας, με, το, με, τις, με τους δικούς μας στόχους και το τι ακριβώς καινοτομία θέλουμε να έχουμε. Μείωση του διοξιδίου του άνθρακα, μείωση άλλων τοξικών ουσιών. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό να είναι απολύτως σαφές εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η στρατηγία του 2020 θα έχει ως στόχο αυτούς ακριβώς, αυτός, αυτές ακριβώς τις πτυχές ε, και την ένωση των, της καινοτομίας με την κλιματική αλλαγή. Γιατί νομίζω ότι θα επανέλθουμε στην κατάσταση που επικρατούσε ε, όταν συζητούσαμε τη στρατηγική τη Λισαβόνα. Και επανέρχομαι στο βασικό. Ποιο είναι ο βασικός ε, συνδυασμό μεταξύ των στόχων της πολιτικής 2020 και των κρατών μελών και των στόχων των κρατών μελών. Αν δηλαδή τα κράτη-μέλη δεν είναι έτοιμα να παρακολουθήσουν, δεν είναι έτοιμα να μας ακολουθήσουν και να προχωρήσουν ε, με ε, προγράμματα μέσα των ε, διαφορετικών ταμείων και, του Ταμείου συνοχή, τότε θα αποτυχούμε και πάλι. Οπότε πρέπει να καταστήσουμε σαφέ το ποιο θα αναλάβει α πούμε την ε, ηγεσία όλων αυτών, ποια είναι η αιρεσιμότητα εδώ για τα κράτη-μέλη και πώς ακριβώς θα μετρήσουμε την επιτυχία, δηλαδή τι θεωρούμε επιτυχία ουσιαστικά και πώς τη μετρούμε. Ίσως θα μπορούσατε να επανέλθετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Χέλγα. Η Κίνγκα. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι συζητούμε το, την πλέον ε, σημαντική πτυχή της ε, στρατηγικής 2020, γιατί το συνδέουμε και με τον ε, προπολογισμό. Νομίζω ότι αυτό ήταν το πιο σημαντικό και της ε, στρατηγικής της Λισαβόνα, ότι ναι, υπάρχουν πολύ ωραία σλόγγαν κτλ, αλλά χωρίς να έχουν καμία εφαρμόσιμη αξία. Χάρηκα που άκουσα ότι η πολιτική συνοχή θα πρέπει να καλύπτει και τους πέντε στόχους. Νομίζω ότι το χειρότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να ε, κατακριματίσουμε τον, ε, ε, τον προπολογισμό. Έχουμε ξεχωριστό προπολογισμό για κάθε στόχο κτλ. Δεν πρόκειται να πετύχουμε τίποτα έτσι. Το γνωρίζουμε καλά όλοι. Το βασικό ερώτημα και το είπανε και οι υπόλοιποι συνάδελφοι είναι πώς θα ε, τα εφαρμόσουμε όλα αυτά. Είπατε κι εσείς ότι έχουμε τομεακούς στόχους, έχουμε εδαφικά προγράμματα, ε, συγκεκριμένες προτεραιότητες και, προτεραιότητες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε και τις ομάδες κρούσης τις Task Force. Ε, είναι σημαντικό, είναι πολύ χρήσιμο ε, εργαλείο ώστε να μην χρειαστεί να κατακαιρματίσουμε τον ε, τον ε, προπολογισμό. Νομίζω ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τις ομάδες αυτές, συνδέοντας όλους αυτούς τους στόχους. Και άλλο ένα πολύ σημαντικό είναι πώς θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε με τα διάφορα επίπεδα κυβερνήσεων, τοπικών, ε, περιφερειακών, εθνικών, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί δεν έχουμε παρόμοιε δομέ, εναρμονισμένε δομέ, ώστε να μπορέσουμε να εναρμονίσουμε και του στόχου. Και ακόμη εξακολουθούμε να διατρέχουμε τον κίνδυνο αυτά τα project να σχετιστούν ε, με συγκεκριμένα επίπεδα ε, διακυβέρνησης. Οπότε πριν πάρουμε όλες αυτές τις αποφάσεις, νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε περισσότερο τις δομές των ε, διαφόρων επιπέδων διοίκησης. Και επίσης θα πρέπει να να δούμε και το ευρωπαϊκό εξάμεινο ε, και εκεί ίσως θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την εναρμόνιση εθνικού και ευρωπαϊκού επίπεδου, αλλά νομίζω ότι αυτές οι διαδικασίες θα πρέπει να τις δούμε πολύ καλύτερα για το μέλλον, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ελίζα. Thank you very much. I think this is Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είναι πολύ κρίσιμο το ζήτημα που συζητούμε εδώ. Και η ερώτησή μου αφορά τη συμβατότητα ανάμεσα στο πακέτο ε, για την οικονομική διακυβέρνηση, το οποίο επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή και το οποίο απαιτεί πολύ έντονο συντονισμό μεταξύ των χωρών έτσι ώστε οι πιο περιφερειακές χώρες να μπορέσουν να μπουν σε ένα δρόμο περικοπών των κυβερνητικών δαπανών για να ενταχθούν σε μία ονομαστική σύγκληση των οικονομικών δικτών τους και να αποφύγουν ε, τις κυρώσεις σε περίπτωση παράβαση αυτών των στόχων. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι επαρκής προστασία ούτε των εθνικών συνεισφορών για τους στόχους του 2020, γιατί μερικές από τις χώρες αυτές όταν μειώνουν τις δαπάνες τους, αναπόφευκτα περικόπτουν ό,τι έχει να κάνει με την παιδεία, την κατάρτιση, την επιστήμη, την τεχνολογία ε, και χάνουν τη σχετική προστασία αυτών των τομέων και από την άλλη πλευρά υπάρχει ένα άλλο φαινόμενο. Η περικοπή ε, των ε, εθνικών συμβολών συνεισφορών στα διαρθρωτικά ταμεία. Ε, οι Financial Times σήμερα αναφέρουν ότι μόνο 10% από τα 347 δισεκατομμύρια για την ε, ανάπτυξη έχουν καταβληθεί γιατί οι χώρες που πραγματικά έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για την ανάπτυξη δεν οργανώνονται έτσι ώστε να πληρώσουν τη συμβολή τους στα όργανα και τα εργαλεία της συνοχής. Αυτή δεν είναι μια καλή λύση γιατί έτσι οι αποκλήσεις θα πολλαπλασιαστούν και η ικανότητα χρήσης των διαθροτικών ταμείων θα μείνει ε, να εωρείται. Νομίζω ότι χρειάζεται να σημειωθεί μια πιο οριζόντια πρόοδος για τις ε, για την εξισορρόπηση αυτών των διαρθρωτικών ανισοτήτων, έτσι ώστε οι χώρες ε, να δουν, ιδίως αυτές που είναι εντός της Ευρωζώνης, πώς θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στην ατζέντα για το 2020. Και αυτό νομίζω ότι δημιουργεί άλλη μια πρόσθετη πίεση στο, για το ρόλο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας γι' αυτό. Ευχαριστώ. Τελευταίος ο Ζωζέ Μανουέλ και μετά να περάσουμε στις απαντήσεις. Ευχαριστώ. Θα ήθελα το πάνελ να μας βοηθήσει να καταλάβουμε Ποια πρέπει να είναι η δομή του επόμενου προϋπολογισμού. Μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτά. Ε, πώς το βλέπετε. Πιστεύετε ότι κάθε κατηγορία πρέπει να αντιστοιχεί σε κάποια προτεραιότητα, ε, ανάπτυξη για όλους, βιώσιμη. Εν τέλει, ποια είναι η δομή που προτιμάτε εσείς για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να έχει διάρκεια 10 ετών με υποχρεωτική αναθεώρηση κάθε 5 χρόνια. Έτσι θα έχουμε ε, το θεσμικό μας ρόλο, αλλά ταυτόχρονα και τα κράτη-μέλη θα υποχρεωθούν να ε, προβαίνουν στις αναγκαίες αναθεωρήσεις των ποσών. Ε, η στρατηγική για το 2020 έχει έντονη συμβολική αξία βέβαια, αλλά δεν θα ήθελα να θεωρούμε ε, ότι θα μπορούσαμε να κινηθούμε σε ένα επταετές πλαίσιο όπως το προηγούμενο. Μιλάμε για το 2020, θα πρέπει να έχουμε ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο πέντε ετών. Θα πρέπει πιστεύω λοιπόν η διάρκεια να είναι 10 χρόνια. Άλλο σημαντικό ζήτημα. αν σκεφτεί κανείς και το ισχύον πλαίσιο και το μελλοντικό πλαίσιο, είναι να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή όλων των πλευρών. Επίσης, σκέφτομαι την διαφάνεια. Συχνά δεν ξέρουμε, δεν έχουμε εικόνα του ποιοι καταλήγουν τα χρήματα αυτά και για ποια προγράμματα προορίζονται. Είναι λοιπόν σημαντικό να ξέρουμε ποια προγράμματα έχουν εγκριθεί, και πώς ε, έχει η κατάσταση. Η συζήτηση αυτή θα πρέπει να αρχίσει ήδη από χαμηλότερο επίπεδο. Μετά, το ζήτημα ε, του μηδέν η εδαφική συνεργασία κτλ. Και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Στη συνέχεια, ποια μεθοδολογία πρέπει να υιοθετήσουμε για αυτό το χρηματοδοτικό πλαίσιο, το πολιετές. πρώτα συμφωνείτε το ποσό και μετά διαιρείτε το ποσό ανάλογα με τις πολιτικές προτεραιότητες και τη μεθοδολογία ή πρώτα θα, θα θέτουμε τις προτεραιότητες και στη συνέχεια για κάθε προτεραιότητα, για κάθε δράση θα καθορίζουμε ένα ποσό και στο τέλος θα κάνουμε την πρόσθεση και θα ξέρουμε ποιο θα είναι το συνολικό και οριστικό ποσό. Δηλαδή, με λίγα λόγια, θα είναι μια μεθοδολογία από κάτω προς τα επάνω. Ποια είναι η μεθοδολογία που κατά την άποψή σας πρέπει να ακολουθήσουμε. Ο κύριος Γιώργος Σταυρακάκης. Και μετά να κλείσουμε τον κατάλογο των ομιλιών. Πολύ πολύ σύντομος. Έχω μία ερώτηση στον κύριο Ντίνκα. Αν κατάλαβα καλά, ο στόχος απασχόληση ε, προτείνεται να αντικατασταθεί με τον στόχο παραγωγικότητα. Και επειδή τουλάχιστον εγώ στο μυαλό μου έχω ότι αυτοί οι δύο στόχοι βρίσκονται σε σχέση καθρέφτη ενώ ειδόλου αντικειμένου, θα παρακαλούσα τον κύριο Ντίνκα να μας πει ε, κάτι παραπάνω έτσι ώστε να κατανοήσουμε ακριβώς τη διαφορά μεταξύ αυτών των δύο νόρων. Ευχαριστώ πολύ. Yes, uh, before giving the floor to the panelists in the opposite direction. Πριν δώσω το λόγο στο πάνελ από το τέλος προς την αρχή, να πω κάτι. Ας κάνουμε ένα έτσι πείραμα στο μυαλό μας. Η πρώτη, το πρώτο ερώτημα είναι η 2020 η πολιτική για τη δεκα, η δεκαετής πολιτική ή η πενταετής πολιτική. Αν μιλούμε για τη δεκαετή πολιτική ξεκινούμε τώρα με τον προπολογισμό που έχουμε. Ή είναι η πολιτική που θα ξεκινήσει με τον νέο προπολογισμό. Οπότε προετοιμάζουμε τον προπολογισμό αντίστοιχα για την νέα πολιτική. Εγώ νομίζω ότι η πολιτική 2020 είναι μια δεκαετής πολιτική και ξεκινά τώρα. Και τώρα θέτουμε τους στόχους και τις προτεραιότητες και πρέπει να ξεκινήσουμε τώρα. Βέβαια το θέμα είναι πώς θα αλλάξουμε τις, ε, ε, τις ε, προτεραιότητες μας για, τον, για να γίνει πιο αποτελεσματική η πολιτική μας μέσω και του προϋπολογισμού. Αν θέλει κανείς να αλλάξει τη διάρθρωση του προϋπολογισμού, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από ό,τι φαίνεται την ε, στρατηγική για το 2020 το 2014. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τον κύριο Ντίγκα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να μιλήσω για συγκεκριμένα τέσσερα ζητήματα ε, και άλλωστε τρία ερωτήματα απευθύνθηκαν σε μένα προσωπικά. Το τέταρτο είναι γενικότερο. Σε ό,τι αφορά την αμφιβολία για την ε, διασύνδεση παραγωγικότητας συνοχής, η κοινωνική ένταξη που είναι στόχος της πολιτικής συνοχής, φυσικά και συνεπάγεται την ποιότητα ζωής Και η ποιότητα ζωή βέβαια περιλαμβάνει την αναψυχή, τον ελεύθερο χρόνο, γιατί η προσωπικότητα αναπτύσσεται κυρίω στη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου. Και αυτό σχετίζεται και με την παραγωγικότητα. Δεν θέλω να αναφερθώ στην αμυγό οικονομική έννοια τη παραγωγικότητα, αλλά στην έννοια τη αποτελεσματικότητα, τη οικονομική δραστηριότητα. Και όταν πρότεινα η παραγωγικότητα να συσχετιστεί με την απασχόληση, αυτό το οποίο σκεφτόμουν είναι ότι αν υπάρχει μεν απασχόληση αλλά μειωμένη παραγωγικότητα, δεν θα εξασφαλιστεί κοινωνική συνοχή, ποιότητα ζωή, έλεγχο χρόνο κτλ. Ούτε και το αντίστροφο όμω ισχύει. Δηλαδή, μεγάλη παραγωγικότητα που όμω δεν οδηγεί σε απασχόληση, ε, με το ίδιο ποσοστό τουλάχιστον, επίση οδηγεί σε κοινωνικό αποκλεισμό. Είναι στατιστικό ο δείκτη αλλά όχι ποσοτικός, δεν είναι δείκτη ποσοτικοποίηση, είναι μία έννοια, είναι ενιολογική προσέγγιση που, που κάνω. Πρέπει να το δούμε λοιπόν ε, ως ένα σύνολο αυτό το δίπτυχο παραγωγικότητα συνοχή. Τώρα για το επίπεδο 0 ε, ήταν ε, πιο πολύ μια παρομοίωση αν θέλετε ή μια μεταφορά. Έχουμε τις ευρωπεριφέρειες στο πλαίσιο της εδαφικής συνοχής. Θα μπορούσαμε, λέω, να δημιουργήσουμε και κάποιες οικονομικές ή κοινωνικές περιφέρειες που έχουν ισχυρή οικονομική ανάπτυξη και θα μπορούσαν να είναι μοχλή οικονομικής ανάπτυξης αλλά και κοινωνικής συνοχής. Βλέποντας ε, βέβαια τα πράγματα έτσι με κάποιο χρονικό ορίζοντα, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να σκεφτούμε το ενδεχόμενο αυτής της περιφερειακής διάρθρωσης, ιδίως γιατί τα αναπτυξιακά προγράμματα είναι εθνικά και δεν υπάρχουν ομοιογενή κριτήρια σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σημαντικότερο ερώτημα το οποίο ετέθε εδώ, κατά την άποψή μου, έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο θα είναι διαρθρωμένος ο προϋπολογισμός λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους ε, της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Εγώ συμφωνώ με αυτό το οποίο είπε η κυρία Γκίνκα Γκέντς. Δηλαδή, ότι ο προϋπολογισμός είναι ένα μέσο. Αυτό είναι προφανές. Αυτό το οποίο εγώ ως εμπειρογνώμων θα έκανα θα ήταν πέραν του ευρωπαϊκού προπολογισμού να έχω και μια δημοσιονομική στρατηγική ευρωπαϊκή με οικονομικούς, κοινωνικούς, εδαφικούς στόχους και στον προπολογισμό αυτό θα έφτιαχνα μία δομή δαπανών βάση των μέσων. Ένα μέσο, είπε η κυρία ε, Γκέντς, δεν πάει μόνο σε ένα στόχο, μπορεί να ε, έχει επιπτώσεις σε διάφορους στόχους, περισσότερους του ενός. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια δομη δαπανων βάσει των μεσων ενα μεσο ειπε η κυρια γκεντς δεν παει μονο σε ενα στοχο μπορει να εχει επιπτωσεις σε διαφορους στοχους περισσοτερους του ενος πρεπει λοιπον να εχουμε μια στρατηγικη με κάποιους τελικούς στόχους και έναν προϋπολογισμό με κεφάλαια δαπανών που δεν απευθύνονται κατά περίπτωση σε συγκεκριμένους στόχους. Και θα πρέπει να έχουμε και μία μήτρα για να μπορούμε να τα επαληθεύουμε όλα αυτά. Of, uh, Barca. Αυτό που λέει ο Φαμπρίτσιο όντως είναι, είναι σωστό. Για να δούμε. που θα έβαζα εγώ την ε, πολιτική συνοχή. Εκεί που είναι, ως ξεχωριστό τίτλο. Απλώς θα προσέθετα τη λέξη ανάπτυξη. Νομίζω ότι θα ήταν λάθο να μην το κάνουμε. Γιατί γι' αυτό, ε, περί αυτού πρόκειται. Αν όλα τα θεσμικά οργανά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι έτοιμα να περάσουν από το 2020 στο 2024, τότε θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ένα 5 συν 5, δύο πενταετίες. Ε, αλλά το 5 5 θα πρέπει να πληρεί και τις 5 προϋποθέσεις. Ότι θα γίνει η μεταρρύθμιση της ε, πολιτικής συνοχής, που τη συζητούμε τώρα και που θα είναι τόσο αποτελεσματική ώστε να μην χρειάζεται άλλη αλλαγή από το 2014 μέχρι το 2024. Δεύτερον, ότι οι δημοσιονομικοί πόροι θα καθοριστούν με βεβαιότητα για τουλάχιστον 7 χρόνια, ακόμη και αν μιλήσουμε για 5 5, γιατί τα 5 χρόνια είναι λίγα για πολλά προγράμματα. Τρίτον, ότι ο πρόεδρος του των τελευταίων, μάλλον το ε, μερίδιο συγγνώμη, των τελευταίων τριών χρόνων θα συνδέεται με τα προηγούμενα και ότι η σύμβαση που θα γίνει μεταξύ κρατών μελών, κομισιών και περιφερειών θα καταγραφεί μέχρι το τέλος του πέμπτου έτους. Ε, εντάξει, αυτό, αυτές είναι οι δικές μου απόψεις, εν πάση για να μπορέσουμε να περάσουμε από το 2020 το 2024, τέλος δηλαδή της προγραμματικής περίοδου και του οράματος που έχουμε. Τρία επιχειρήματα υπάρχουν. Ένα είναι ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε το περί τίνος πρόκειται όταν μιλούμε για ε, ανάπτυξη. Μιλούμε ανάπτυξη στην, ε, στο χώρο εργασία, στους ακαδημαϊκούς, στις πολιτικές που καλύπτουν ε, και το θέμα της ε, επάρκειας, της αποτελεσματικότητας, μιλούμε για μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα, μιλούμε για κοινωνική συνοχή, κοινωνική ισότητα, αυτά δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Αυτά, αυτά είναι η ανάπτυξη, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα από αυτά, ακόμη και αν θέλαμε. Δεύτερον, η καινοτομία της πολιτικής είναι ότι πρέπει να έχει σαφείς στόχους, σαφείς δείκτες και σαφή αποτελέσματα. Ακόμη δεν έχουμε ε, δείκτες για τα τρία σλόγγαν, έχουμε δείκτες για τους πέντε στόχους που έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο. Και τρίτον, έχουμε, οι πολιτικές είναι περίπλοκες. Έχουμε πρόβλημα λοιπόν. Έχουμε Τρει ή πέντε τέλο πάντων διαφορετικούς στόχου που συνδέονται μεταξύ του. Όπω είπαμε, βιωσιμότητα και καινοτομία για παράδειγμα. Μόνο μία πολιτική που θα τα καλύπτει όλους μπορεί να, καταλήξει στο εξή αποτέλεσμα. αν έχουμε, ε, στην επιτυχία δηλαδή, αν έχουμε συγκεκριμένε ε, ξεχωριστές μιλούμε για παρέμβαση. που θα είναι στοχευμένη είτε προς ε, την ε, κλιματική αλλαγή, είτε προς την ισότητα κτλ. Αλλά κάθε φορά που κάνουμε ένα project, πρακτικά έχουμε ένα ε, στόχο και έχουμε και κάποιους περιορισμούς. Μόνο αν τα ενώσουμε όλα αυτά κάτω από την ίδια πολιτική θα μπορέσουμε να έχουμε τους στόχους χωρίς να ξεχνούμε όμως και τους μεμονωμένους τομείς για τους οποίους πρέπει να επιτύχουμε τους στόχους. Τρίτον, πώς θα εξασφαλίσουμε ότι τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Η μετρησιμότητα και η αιρεσιμότητα είναι δύο βασικά στοιχεία. Η μετρησιμότητα των στόχων και η αιρεσιμότητα. Αν δείτε τον πίνακα που έχω εδώ στην ε, παρουσίασή μου. Αν δείτε τη διαδικασία της πολιτικής συνοχής στα αριστερά, υπάρχουν ε, δύο βασικά σημεία. Ένα με την γενική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εκεί θα καθοριστεί και η αρχή της αιρεσιμότητας. Μιλούμε δηλαδή για αρχές που θα διατηρηθούν και θα ισχύουν για όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης ώστε, και πρέπει να είναι αρκετά γενικόλογες, ώστε να μην αντικατοπτρίζουν οποιοδήποτε πολιτισμό ή οποιοδήποτε ειδικό εθνικό πλαίσιο και θα πρέπει να συνάδουν και με τις ε, ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές. Ούτε να εξαρτώνται ε, από αυτές, αλλά θα πρέπει να είναι συνεκτικές. Η ομάδα της, διαπραγματευτική ομάδα της Κομισιόν έφτιαξε αυτές τις ομάδες ε, της Task Force. Βεβαίως αυτές θα πρέπει να συνεργαστούν και με τις ε, ε περιφέρειες γιατί τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να συμφωνηθούν ταυτόχρονα. Υπάρχουν ε, ομοσπονδιακά κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου δεν υπάρχει σύμβαση ε, ανάπτυξη χωρί να έχει δώσει τη σύμφωνη γνώμη τη η περιφέρεια. Είναι δηλαδή νόμο αυτό. Οπότε σε αυτή τη ε, διαπραγμάτευση ε, αυτές οι βασικές αρχές που έχουν τεθεί για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνονται δεσμευτικέ. Οπότε δεν θα σα δώσω ε, τα λεφτά ή δεν θα δεχτώ εγώ τα λεφτά εάν μπορώ να εγγυηθώ ότι θα υπάρξουν θεσμικές προσαρμογές. Και κλείνω λέγοντας ότι θα πρέπει να δούμε τους ε, ε, δείκτες για το αποτελέσματος. Έχουμε το, το, τους δείκτες αποτελέσματος για την Ευρώπη στο σύνολό τη. Έχουμε τους στόχους για τα κεφάλαια και έχουμε και κάποιους δείκτες οι οποίοι θα τεθούν για τον, ε, για τον Ευρώπη στο σύνολό της. Μετά θα δούμε τα προγράμματα που θα τα αποφασίσουν τα κράτη-μέλη μαζί με την Κομισιόν. Και επίση, ε, οι δείκτε αποτελεσμάτων για τα project, τα οποία τα έχουμε, τους οποίους έχουμε ξεχάσει συχνά στο παρελθόν. Οι κοινοτικοί δείκτε είναι καινοτόμοι, αναπτύσσονται σε πολλά κράτη-μέλη και μετά τα πράγματα είναι απλά. Απλώ θα ζητούμε, θα βάζουμε κάποια απέτηση. Α πούμε, όποιο χρησιμοποιεί ε, τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων θα πρέπει να, έχουν, να έχει ένα συγκεκριμένο στόχο στο project του. Και θα πρέπει να μα πει ποιο είναι, ποιο είναι ο μετρήσιμος δείκτης βάσει του οποίου θα μετρήσει τι συνέπειε, όχι το πόσα χιλιόμετρα ταξίδια έκανε ή πόσους ανθρώπους ε, ε, χρησιμοποίησε, αλλά πώς χρησιμοποίησε, αν βρήκε καλύτερο ανθρώπινο δυναμικό, με καλύτερες δεξιότητες, με περισσότερα προσόντα κτλ. 30 δευτερόλεπτα, πρόεδρε μου, δίνετε για να πω ένα τελευταίο για, το, για τα μάκρο θέματα. Στην Ευρώπη δεν μπορείς να αποφύγεις ε, το αντιστάθμισμα που πρέπει να δώσεις, αλλά όλα αυτά πρέπει να γίνονται σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο, ώστε όλα αυτά να είναι υπόλογα, να μπορούν να είναι συζητήσιμα. Ένα είναι η αναθεώρηση της ε, αρχής της, ε, ε, του, της επιπλέον ε, ε, της προσθέμενης αξίας το, την οποία μπορούν να μετρήσουν όσοι ασχολούνται με τα μακροοικονομικά θέματα έτσι ώστε να μπορέσουμε όλοι να δούμε αν υπάρχει κάποια αντίθεση, αντίφαση κάπου και να απαλάβουμε την αντίστοιχη πολιτική απόφαση. Αλλά τουλάχιστον θα είναι όλα αυτά διαφανή. Δεν σας πειράζει ε, για την ερώτηση του κυρίου Φερνάντες να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ορολογία του να μην μετατρέπουμε τα σλόγγαν σε επικεφαλίδες. Σωστά το είπα? Μάλιστα, σωστά το είπατε. Yes, but but... Ναι, αλλά η ερώτησή σας είναι πώς να οργανώσουμε τις δημοσιονομικές προοπτικές, σε τι είδους διάγραμμα, σε τι είδους διάταξη. Τέλος πάντων, παρακαλώ, απαντήστε. Συγγνώμη, δεν ήθελα να επισέλθω σε αυτό γιατί είχα πολλά πράγματα να πω και δεν, δεν είμαι έτοιμος αυτή τη στιγμή να παρουσιάσω αναλυτικά ένα σχέδιο ή ένα διάγραμμα ή μια διάταξη. Εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω την ανάπτυξη σαν μια γενική επικεφαλίδα και κάτω από την ανάπτυξη θέλω να απαριθμούνται όλες οι πολιτικές. Για παράδειγμα, ένα α, προγράμματα συμβάλλουν στην ανάπτυξη αλλά μόνο στην καινοτομία. Ανήκουν λοιπόν στην ανάπτυξη. Ενώ η ανάπτυξη περί είναι κάτι που πιάνει και τις τρεις πτυχές. Αυτού του τύπου το σχήμα έχω στο μυαλό μου. Ο τελευταίος μας ομιλητής θα είναι η κυρία Μερσέντες Μπράσο, πρόεδρος της ε, Επιτροπής Περιφερειών. Ευχαριστώ. Καταρχήν το ζήτημα 5 συν 5. θεωρούμε ότι ένα, μια διάρκεια 10 ετών για την οργάνωση πολύ περίπλοκων προγραμμάτων είναι μια καλή διάρκεια. Αυτή η διάρκεια επιτρέπει την επιδίωξη μιας στρατηγικής για μια επαρκώς μακρά περίοδο και ταυτόχρονα ε, η δυνατότητα μια σημαντικής αναθεώρησης στην πενταετία επιτρέπει την προσαρμογή, την πιο ταχεία προσαρμογή ή τροποποίηση. Ε, ώστε να ανταποκριθούμε στις αλλαγές ε, των οποίων διέρχονται οι κοινωνίες μας. Επίσης ανταποκρίνεται και στον ρυθμό εναλλαγής ε, των ευρωπαϊκών οργάνων. Ξέρετε ότι έχουμε μια καινούργια επιτροπή κάθε πέντε χρόνια και έτσι μπορεί να ληφθεί σωστά υπόψη αυτή η εναλλαγή στο επίπεδο της πενταετίας. Ε, η άλλη ερώτηση ήταν αν ξεκινούμε τώρα αμέσως ή το 2014-2015. Πότε ξεκινάει η στρατηγική για την Ευρώπη του 2002. Εγώ νομίζω ότι ξεκινάει ευθύς αμέσως. Νομίζω ότι είναι δυνατόν ήδη να στρέψουμε την προηγούμενο προγραμματισμό προ τους στόχους μας. Είναι κάτι που μπορεί να γίνει, αλλά προφανώς πρέπει ε, να πούμε ότι ε, πότε καθίσταται πραγματικά η στρατηγική για το 2020, κοινή στρατηγική όχι μόνο των κοινοτικών οργάνων αλλά και των κρατών, των περιφερειών, των πόλεων, των δήμων, ώστε να επηρεάζεται ολόκληρη η πολιτική και όχι μόνο η πολιτική των Ευρωπαϊκών Ταμείων. Ε, για να έχουμε αποτελέσματα και εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως ε, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στην ε, Επιτροπή Περιφερειών, να δημιουργήσουμε μια πραγματική ε, προσήλωση στο ευρωπαϊκό σχέδιο, έτσι να, να δημιουργήσουμε αν θέλετε την ε, νοητική, τη σωστή νοητική προσέγγιση προς την στρατηγική της Ευρώπης για το 2020 που πρέπει να είναι πράσινη, ίσως κοινωνική και ταυτόχρονα καινοτόμα και το πράσινο και κοινωνική και τα δύο είναι καινοτόμα πράγματα. Δεν είναι παραθετική η σύνταξη, πράσινη, κοινωνική, καινοτόμα. Πρέπει να είναι και τα τρία ταυτόχρονα. Το ζήτημα των προϋποθέσεων και της μετρησιμότητας. Νομίζω ότι το ζήτημα των προϋποθέσεων ε, συνδέεται ε, με τους δείκτες, οι οποίοι πρέπει να είναι απλοί και μετρήσιμοι. Συμφωνώ με τον κύριο Μπάρκα. Αντίθετα, ε, είμαστε εντελώς αντίθετοι με την ιδέα των μακροοικονομικών προϋποθέσεων που θα, που θα σήμαινε ότι αν τα κράτη-μέλη δεν σεβαστούν το σύμφωνο σταθερότητας, τότε οι περιφέρειες θα χρησιμοποιήσουν ιδίως το, ταμείο, το Γεωργικό Ταμείο, το Ταμείο Ανάπτυξης της Υπέθρου, ε, ε, όλα αυτά θα υποστούν τις συνέπειες ε, της μη του Συμφώνου Σταθερότητας από τα κράτη-μέλη. όχι, αυτό θα ήταν λάθος. Θα ήταν μια καθαρή παραβίαση της αρχής της επικουρικότητας και θα μπορούσε κανείς να καταφύγει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. νομίζω ότι η αρχή των προϋποθέσεων σημαίνει να θέσουμε πόρους στη διάθεση εκείνων που με μεγαλύτερη επιτυχία υπηρετούν τους στόχους της Ευρώπης για το 2020 και σε αυτούς να διοχετευθούν οι πόροι των διαρθρωτικών ταμείων. Τώρα, πώς να εξασφαλίσουμε μια πολιτική συνοχής ολοκληρωμένη ε, που να περιέχει όλους τους στόχους και τα πέντε σημεία τα οποία παρουσίασε ο κύριος Μπάρκα. Νομίζω ότι η ιδέα ενός ενιαίου κειμένου προγραμματισμού το οποίο να περιέχει να εμπεριέχει όλους τους πόρους, όχι μόνο το Ταμείο Συνοχής, το Κοινωνικό Ταμείο, ε, το το Ταμείο της Ανάπτυξης της Υπέθρου, την κοινή γεωργική πολιτική. Ε, νομίζω ότι είναι ένας σωστός τρόπος για να έχουμε ένα γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ο καθένας εντάσσει τις προτεραιότητές του λαμβάνοντας υπόψη τους κοινού στόχους. Ο καθένας επιλέγει από το μενού που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιλέγει ο καθένας λοιπόν τις προτεραιότητές του και τις εντάσεις σε ένα συνολικό πλαίσιο. Στη συνέχεια φυσικά κάθε πολιτική θα έχει το δικό της ειδικότερο πλαίσιο, το οποίο θα επιδιώκει και θα υπηρετεί τους συγκεκριμένους στόχους αυτής της πολιτικής. Για παράδειγμα, η γεωργική πολιτική να, να δει κανείς τη γεωργική πολιτική υπό το πρίσμα της ε, βιωσιμότητας, υπό το πρίσμα της ικανοποίησης των στόχων της κλιματικής αλλαγής. Είναι θεμελιώδου σημασίες. Το κοινό πλαίσιο προγραμματισμού λοιπόν θα πρέπει να πλαισιώνει όλες τις πολιτικές σύμφωνα με τη στρατηγική της Ευρώπης το 2020 και σύμφωνα με τους ε, στόχους που κάθε εδαφική υποκατηγορία έχει ε, επιλέξει. Στη συνέχεια, προφανώς, επί τη βάση αυτών των γενικών κατευθυντήριων στρατηγικών κατευθύνσεων, θα πρέπει να διαμορφωθεί ειδικότερα η κάθε πολιτική. Νομίζω ότι έτσι πρέπει έτσι δείχνει κανείς ταυτόχρονα και ότι είναι υπεύθυνο για μια κοινή στρατηγική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και ότι την υλοποιεί ο καθένας και την εξειδικεύει με βάση τις ιδιαιτερότητές του και με βάση τις ειδικότερε ανάγκες του. Τέλο, τελευταίο ζήτημα, ο προϋπολογισμός. Είναι αλήθεια ότι τα κράτη, οι περιφέρειες και η τοπική αυτοδιοίκηση υφίστανται μια τέτοια αυστηρή κατανομή πόρων που πολλές φορές δεν καταφέρνουν να ανταποκριθούν στις ε, στρατηγικές επενδύσεις που απαιτεί η στρατηγική για την Ευρώπη του 2020. Ποιος μπορεί να κάνει αυτές τις επενδύσεις. Νομίζω ότι το 1% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ προφανώς δεν επαρκεί για τον προσανατολισμό των πολιτικών. Ταυτόχρονα οι αυστηρότητες και οι ακαμψίες των εθνικών προϋπολογισμών επίσης δεν επιτρέπουν ε, δεν ανοίγουν και μεγάλα περιθώρια επενδύσεων. Είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Νομίζω ότι οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από δημοσιονομικής άποψης πρέπει να γίνουν λίγο περισσότερο φιλόδοξες και πρέπει να βρεθούν πόροι. Πόροι καταρχήν να βρεθούν δυνατότητες αύξησης των πόρων, να εξεταστεί η δυνατότητα έκδοσης ευρωπαϊκών ομολόγων, τουλάχιστον για τις μεγάλες επενδύσεις και για τις μακροπρόθεσμες ε, στρατηγικές και νομίζω ότι αυτά πρέπει να ε, συνυπολογιστούν, γιατί δεν μπορεί δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι θα επιδιώξουμε τέτοιες ευρείες στρατηγικές, φιλόδοξες στρατηγικές με έναν ελάχιστο προϋπολογισμό και με κράτη-μέλη που θα είναι υποχρεωμένα να υφίστανται σε αυτούς τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, τους τρομακτικούς μερικές φορές. Ποια θα είναι η πραγματικότητα τελικά πίσω από τις λέξεις πίσω από τις λέξεις πρέπει να υπάρχουν πόροι, γιατί χωρίς πόρους κανένας δεν θα καταφέρει να επηρεάσει την πολιτική του και να αλλάξει την κατάσταση της επικράτειας της εκάστοτε επικράτειας. Νομίζω ότι εδώ ε, με το Κοινοβούλιο ε, με το Κοινοβούλιο μπορεί να συμφωνούμε ως προς αυτό, αλλά πολύ λιγότερο δυστυχώς συμφωνούμε με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ακούσαμε εξαιρετικά συμπεράσματα από τους ομιλητές ε, του πάνελ. Και σε ό,τι αφορά τους στόχους μας και δει τους στόχους στρατηγικής 2020, για να προχωρήσουμε θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με όλα αυτά τα επίπεδα. Είναι προφανές ότι όπως και για την ε, στρατηγική της Λισαβόνας ε, θα οδηγηθούμε σε αποτυχία. Όπως είπα και χθες ε, όταν μιλάω στον πληθυντικό, δεν μιλάω για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε κάμια περίπτωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντοτε υποστήριζε και υποστηρίζει την κοινοτική προσέγγιση για να την αποκαλέσω έτσι. Και πάντοτε εκφράζουμε την ευχή να συμφωνήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με το τι πρέπει να υλοποιηθεί σε επίπεδο κρατών μελών. Αυτοί οι οποίοι σε τακτά διαστήματα μπλοκάρουν τα πράγματα είναι τα κράτη-μέλη. Και δεν θα πω το Συμβούλιο, γιατί νομίζω ότι μεμονωμένα τα κράτη-μέλη πολλές φορές δημιουργούν τα προβλήματα και όχι σαν συλλογικό όργανο το Συμβούλιο. Θέλω να ευχαριστήσω τους ομιλητές του πάνελ που μας ε, βοήθησαν να, μορφώσουμε άποψη και να καταλήξουμε σε μία θέση την οποία τον Ιούνιο του 2011 θα πρέπει να εγκρίνουμε ως θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις μελλοντικές δημοσιονομικές προοπτικές. Και συγκεκριμένα θα ψηφίσουμε τον Ιούνιο σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για τη διάθεσή σας και θα καλέσω στο βήμα το επόμενο πάνελ. Δεν πάμε άσχημα όσο ό,τι αφορά το χρόνο που τη βλέπω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 Liebe Kollegen, if you want to continue your conversation, then please outside. Liebe Kollegen, wir sind jetzt... Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαστε στο τέταρτο πάνελ. Να καλωσορίσω όλους όσους είναι εδώ στο πόντιου, Ο συντονιστής μας, ο Φάβιαν Τσούλεκ, είναι οικονομολόγος του ε, Κέντρου για την Ευρωπαϊκή Πολιτική. Μετά, είναι μαζί μας ο Διευθυντής της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ο Ντομινίκ Ντε Χαγενκούρ, η Αμελή Μπαρμπιέ Γκοσά, επιστημονική σύμβουλος στο κέντρο για στρατηγική, για στρατηγική ανάλυση. Η Κέρστη Κάλγιουλα εδώ στα αριστερά μου, μέλος του ελεκτικού συνεδρίου και τον Άντρα Βέρτες, ο οποίος είναι πρόεδρος του GKI για την οικονομική έρευνα. Κύριε Τσούλεκ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ που με καλέσατε σήμερα να πω έτσι κάποια εισαγωγικά για το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Ε, για όσους δεν μας ξέρετε, είμαστε ένας, ε, ένα think tank, ένα, μια δεξαμενή σκέψης ε, που λειτουργούμε στα πλαίσια του, με, με τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό εδώ και κάποια χρόνια. Βλέπουμε τα θέματα διακυβέρνησης και τις επιπλοκές που έχει, τις συνέπειες που έχει η νέα συνθήκη της Λισαβόνας. Νομίζω λοιπόν ότι είναι καλή η παρουσία μας σήμερα εδώ. Θα επικεντρωθούμε σήμερα στις ευρωπαϊκές ε, αρχές και τις πολιτικές. Θα δούμε πώς ο ευρωπαϊκός προπολογισμό μπορεί να ενισχύσει τις επενδύσεις, πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τη συμπληρωματικότητα με τους εθνικού ε, προπολογισμού. Το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε την αποτελεσματικότητα του ε, ευρωπαϊκού προπολογισμού και πώς μπορούμε να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα ανεξαρτήτω του μεγέθου του προπολογισμού. Υπάρχουν πολλά δύσκολα ερωτήματα τα οποία συνδέονται με το θέμα αυτό και είναι ένα κινούμενος στόχο ε, το θέμα, η συζήτηση συνεχίζεται. Θα πρέπει να δούμε πώς έχουν διεξαχθεί οι συζητήσεις για την ευελιξία του ευρωπαϊκού προπολογισμού και στα πλαίσια του προπολογισμού για το 2011. Πρέπει να δούμε τι γίνεται με τη συζήτηση για την οικονομική διακυβέρνηση και το ρόλο που πρέπει να παίξει ο προπολογισμό σε αυτό. Νομίζω ότι ε, θα πρέπει να απαντήσουμε σε κάποια ερωτήματα. Τέσσερα είναι τα βασικά που έχω διαπιστώσει εγώ. Καταρχήν, ποιο, ποιος, ε, ποιος τρόπος δαπανών θα πρέπει να είναι αυτός που θα χρησιμοποιήσει καλύτερα τους πόρους του προπολογισμού και θα φέρει καλύτερα αποτελέσματα. Για τα... Επίσης, είναι αποτελεσματικός ο, ο για τις μεταφορές, για τη διανομή των αγαθών. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε κυρίως στην ε, πολιτική 2020 στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Είναι αυτό, είναι αυτό συμβατό με το τι συμβαίνει σήμερα σε σχέση και με τους, το, με, με που έχουμε ε, τις μεγαλύτερες δαπάνες όπως πούμε τη Γεωργία. Δεύτερο μεγάλο ερώτημα, πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερη προστιθέμενη αξία. Εδώ τίθενται ερωτήματα απλούστευσης, ε, ε, προστιθέμενης αξίας, ευελιξίας, ε, επίσης ελέγχου, γραφειοκρατίας, ευθύνε, ποιε ευθύνε βρίσκονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τι ευθύνη έχουν τα κρατημέλη, το περιφερειακό επίπεδο. Επίσης, ένα τρίτο ερώτημα, τι γίνεται με του Εθνικού και τον ευρωπαϊκό προπολογισμό και τη γενικότερη συζήτηση που γίνεται για την ε, ε, διακυβέρνηση πώς ας πούμε γίνεται η συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και πώς αυτό ε, μπορεί να εξασφαλίσει την συμπληρωματικότητα με τους εθνικούς προπολογισμούς. Και εδώ τίθενται διάφορα, διάφορα δύσκολα ερωτήματα. Υπάρχει προστιθέμενη αξία ε, σε ένα τομέα, ας πούμε, αν ας πούμε, ο προπολογισμό χρησιμοποιηθεί ως μηχανισμός κύρωσης για να ε, ε συγκερασμό των δημοσίων κονδυλίων. Μπορεί αυτός, αυτή η επιτυχία στον ένα τομέα να υπονομεύσει την επιτυχία ενός άλλου τομέα. Και ένας τέταρτος τομέας γενικώ είναι το τι άλλο μπορεί να γίνει στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προπολογισμού και των ε, συνδεόμενων ε, ε, μέσων, ας πούμε, δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και πώς μπορούμε να ισχύσουμε τις επενδύσεις. Και εδώ μιλούμε γενικώ για επενδύσεις και δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σε διάφορους τομείς, όχι μόνο ε, οικονομικές δηλαδή επενδύσεις. Και όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και στα πλαίσια και της δημοσιονομικής κρίσης που περνούμε, οι δημόσιες επενδύσεις θα περιοριστούν δραματικά στις περισσότερες χώρες μέλη στα επόμενα χρόνια. Και επίσης σημαντικό είναι να ξέρουμε ότι έχουμε περίεργες εμπειρίες από την ε, συμπερίληψη του ιδιωτικού τομέα στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλουμε λοιπόν αυτό να γίνει στο μέλλον, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα ενσωματώσουμε τον ιδιωτικό τομέα καλύτερα από ό,τι το έχουμε πράξει στο παρελθόν. Και πολύ πιο σημαντικό είναι να δούμε πώς γίνεται να εξασφαλίσουμε ότι θα επενδύσουμε στις οικονομίες των ε, οικονομικώς αδύναμων χωρών και λόγω της κρίσης ε, με το ευρώ, λόγω και της κρίσης του δημοσιονομικής σε πολλές χώρες. Νομίζω ότι θα είναι αδύνατο να, λύσουμε την, ε, να ξεπεράσουμε τη λύση αυτή εάν δεν επιστρέψουμε στην ανάπτυξη, αν αυτές οι χώρες μέλη δεν, συνεχί, δεν προχωρήσουν στο δρόμο της ανάπτυξης. Αν δεν γίνει αυτό, αποκλείεται να βγουν από την κρίση. Οπότε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εμείς έχουμε ε, την ευθύνη ώστε να χρησιμοποιήσουμε χρηστά τον ευρωπαϊκό προπολογισμό για να μπορέσουμε να ε, εξαλείψουμε τις διάφορες μακροοικονομικές ανισορροπίες που υπάρχουν. Αυτά λοιπόν είναι τα τέσσερα έτσι ευρεία ερωτήματα που θα χρειαστεί να απαντήσουμε. Να δώσουμε τώρα το λόγο στους ομιλητές και θα ήθελα να σας ζητήσω να περιοριστείτε σε πέντε λεπτά έκαστος είναι μεγάλο το θέμα, αλήθεια είναι αυτό, αλλά καλό θα ήταν να έχουμε και κάποιο χρόνο για συζήτηση αργότερα. Ξεκινούμε λοιπόν με τον ε, κύριο Ντε Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, που μας ε, καλέσατε. Ευχαριστώ και τους άλλους, ε, τα λαμέλη του πάνελ να, ξε... αρχίσω από αυτά που είπατε για την αρχή του προβλήματος και συγκεκριμένα. Οι σημερινές δυσκολίες όλων των προϋπολογισμών, είτε είναι κοινοτική είτε είναι εθνική, ε, για την επιβίωση την επαύριο της κρίσης, είναι καθεαυτές ένας κίνδυνος για τις επενδύσεις, για ότι συνήθως προτιμά κανείς να αφιερώσει δαπάνες κρατικές για τη μακροπρόθεσμη, ε, μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Αυτή είναι η μία πλευρά της ιστορίας. Από την άλλη και οι τράπεζες έχουν μεγάλες δυσκολίες, ενοποίησης ε, και Προσαρμογή προσαρμογής στην οδηγία της Βασιλείας για την κεφαλιακή επάρκεια. πρέπει, ε, έχουμε λοιπόν τους προϋπολογισμούς με τους περιορισμούς τους, έχουμε και τις τράπεζες με τους ε, περιορισμούς τους. Από πού να αντλήσουν κεφάλαια με ασφάλεια. Υπάρχουν τόσοι κίνδυνοι. Πρέπει να γίνεται λοιπόν η καλύτερη δυνατή χρήση των πόρων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των Ταμείων της Ευρώπης. Τα βάζω ως δύο φάρους ε, δημοσιονομικών πόρων για τη στήριξη των κοινοτικών πολιτικών. Έχουμε τα κονδύλια από τον ε, κοινοτικό προϋπολογισμό και μετά έχουμε τις μετοχές και τις ε, εκδόσεις γενικώ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Και το ερώτημα είναι πώς να συνδυάσουμε επιτυχώς τα δύο εργαλεία. Ε, καταρχήν, ε, γιατί να χρησιμοποιήσει κανείς μετοχικά δάνεια αντί για κονδύλια. Δεύτερον, ε, ποιο είναι το πλεονέκτημα της χρήσης αμφωτέρων, ενός είδους μείγματος δηλαδή. Και τρίτον, αν επιλέξει κανείς το μείγμα, ποια είναι τα σημαντικά χαρακτηριστικά που πρέπει να παρακολουθεί κανείς για να παρακολουθεί ότι τα δύο αυτά εργαλεία εκπληρώνουν τους στόχους τους και χρησιμοποιούνται σωστά. Λοιπόν, γιατί να, γιατί να χρησιμοποιηθούν κονδύλια για, γιατί δάνεια και όχι κονδύλια. Ε, νομίζω ότι είναι αρκετά απλή η απάντηση εδώ. Η χρηματοδότηση επενδύσεων οι οποίες απαιτούν ε, αποδόσεις, η χρηματοδότησή τους με... Ε, ε, Investment has a low risk and has a very high return. Δεν είναι δυνατόν να επιδοτεί κανείς με, να επιδοτεί κονδύλια επενδύσεις οι οποίες απαιτούν να έχουν αποδόσεις. Έχουμε λοιπόν αναπτύξει ένα ενοιολογικό πλαίσιο ε, για να δούμε πότε να χρησιμοποιούμε τη μία μορφή, πότε την άλλη και πότε ένα μείγμα και τον δύο. Τα, τα πλεονεκτήματα της χρήσης και των δύο είναι τα εξή. Καταρχήν υπάρχει έντονο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα επιτύχαμε με το περίφημο εργαλείο RFFF, δηλαδή το χρηματοδοτικό μέσο ελάφρυσης των κινδύνων για την έρευνα. Ε, για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε ένα εκατομμύριο από τον Ευρωπαϊκό από τον κοινοτικό προϋπολογισμό για να, με μία πρόβλεψη για την τράπεζα που λέει ότι η τράπεζα πρέπει να διαθέσει μέχρι 10 εκατομμύρια για επικίνδυνα ερευνητικά προγράμματα. Και τι συνέβη, αντί να χρηματοδοτηθεί ένα πρόγραμμα ενό εκατομμυρίου που είτε επιτυχάνει οπότε σωστό χρησιμοποιήθηκαν οι πόροι, είτε αποτυγχάνει οπότε κακώς χρησιμοποιήθηκαν οι πόροι, τότε διατίθενται δάνεια ύψου 10 εκατομμυρίων, οπότε αν αποτύχει ένα πρόγραμμα υπάρχουν 9 που μπορούν να επιτύχουν. Αυτό σε πολύ αδρέ γραμμέ είναι το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα τη χρήση ενό μείγματο κονδυλίων ή επιδοτήσεων και δανείων. Δεύτερον, ε, έχουμε την, ε, επιτυγχάνεται η ευελιξία. Η ευελιξία βέβαια εξαρτάται από το τι προσπαθείς να βοηθήσεις. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις. Μπορεί κανείς να βρει ένα σωρό μετοχικά προϊόντα. Τρίτον, ε, δημοσιονομική πειθαρχία και έλεγχος. Όταν πρέπει κανείς να επιστρέψει τα χρήματα, υπάρχει σε μεγάλο βαθμό παρακολούθηση και ανάλυση τόσο της αξίας του ίδιου του προγράμματος όσο και της δυνατότητάς του να επιστρέψει τα χρήματα. Υπάρχει εδώ και ένα θέμα διανεμητικής ε, επάρκειας ε, και ε, αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας που εξασφαλίζει ότι έχει ξοδέψει τα λεφτά σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τα καλύτερα δυνατά προγράμματα. Επίση, τα τελευταία τρία με πέντε χρόνια δόθηκαν χρήματα για έρευνα, για μεταφορές, για μικρομεσαίες επιχειρήσει μέσω των διαρθρωτικών ταμείων. Θα επανέλθω σε αυτά τα διάφορα παραδείγματα, εάν το επιθυμείτε κι εσείς. Τρίτον, ποια είναι τα κυρία χαρακτηριστικά που πρέπει κανείς να παρακολουθεί και να διασφαλίζει όταν χρησιμοποιεί ένα μείγμα εργαλείων, ε, καταρχήν επιδοτήσεων ή κονδυλίων από τον προϋπολογισμό και δανείων ή μετοχικών προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Υπάρχουν τρία βασικά χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει κανείς να διασφαλίζει. Απλότητα, μάλλον να τα εξηγήσω. Απλότητα. Είναι ίσως το πιο ζωτικό. Γιατί τα εργαλεία που είναι αδιαφανή Όλοι ξέρουμε τι έχει γίνει στο παρελθόν. Δεν θέλουμε κάτι πολύ περίπλοκο. Θέλουμε κάτι διαφανές, απλό που να ελαχιστοποιεί το κόστος, που να μπορεί να επαναληφθεί, να αναπαραχθεί σε διάφορες τομείς πολιτικής και που να είναι εύκολο να ελεγχθεί από τους χαράκτες αποφάσεων, πολιτικών αποφάσεων. Το revolving. Το revolving είναι επίσης μια σημαντική πτυχή. Όταν δίνεις χρήματα με χρηματοδοτικά μέσα, θα πρέπει να δοθούν πίσω τα χρήματα αυτά με τον με τον άλλο τρόπο. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να χρησιμοποιηθεί αυτή η ροή επιστροφής για την επαναχρηματοδότηση παρόμοιων προγραμμάτων σε πολλούς επαναληπτικούς γύρους, αν θέλετε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να αυξάνεται έτσι το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα ενός περιορισμένου πολίτη, προϋπολογισμού. Επίσης ενισχύεται ο μηχανισμός ελέγχου με την έννοια ότι είναι οι ίδιοι παράμετροι και τα ίδια κριτήρια ε, τα οποία πρέπει να ελεγχθούν σε κάθε γύρο. Τέλος πρέπει να είναι να δρά ως το μείγμα αυτό. Είναι σημαντικό λοιπόν να ε, προσελκύσουμε και τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα και να προσελκύσουμε πολλούς διαφορετικούς πόρους. Να μην περιορίζεται αυτό στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση παράδειγμα από το πρόσφατο ε, παρελθόν και πιθαν... που μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλαπλασιαστικά. Τα ομόλογα των έργων είναι κάτι το οποίο θα ανέπτυσα αν είχα το χρόνο, γιατί είναι ένα καλό παράδειγμα. Ίσως να το αφήσω για τις ερωτήσεις αργότερα. Να πω απλώς ότι τα ομόλογα των έργων είναι ένα απλό παράδειγμα τέτοιων εργαλείων. Αλλά δεν πρέπει να υπάρχει σύγχυση με τα ευρωπαϊκά ομόλογα. Δεν είναι ευρωομόλογα για την, για επιμήκυνση του προϋπολογισμού, ούτε για να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη. Είναι ομόλογα έργων τα οποία δεν επιβαρύνουν τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Θα το αναπτύξω αργότερα αυτό. Εν κατακλείδη, σε αυτή την εισαγωγική παρέμβαση, να πω ότι για μας είναι πολύ σημαντικό να συνεργαζόμαστε στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να θέσουμε το πλαίσιο της χρήσης αυτών των εργαλείων στο μέλλον με το πολλαπλασιαστικό τους αποτέλεσμα για τις επενδύσεις, για τους πόρους και από την άλλη πλευρά είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει και αυτή η συνεργασία με άλλους διεθνείς, με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς ε, φορείς, πρωταγωνιστές και νομίζω ότι θα σταματήσω εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να πω τα λίγα αυτά λόγια. Um, ευχαριστώ πολύ. Φυσικά και θα σας δώσω τη δυνατότητα ε, να μιλήσετε στη συνέχεια για κάποια ακόμη λεπτά. Ένα ερώτημα, κοιτώντας το μέλλον, τη μελλοντική δημοσιονομική προοπτική, τι νομίζετε ότι είναι το βασικό που θα πρέπει να γίνει διαφορετικά από πλευράς ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Απάντηση. Νομίζω ότι το ερώτημά σας είναι πάρα πολύ δύσκολο και μου το υποβάλλατε έτσι εντελώς ξαφνικά. Ε, αν αυτό σχεδιάσω θα πω ότι ίσως το σημαντικότερο που θα πρέπει να εξασφαλίσουμε είναι να σταθεροποιήσουμε, να παγιώσουμε την παρελθούσα εμπειρία Κάποιες φορές ε, ευτυχώς ή ατυχώς έχουμε επανεφεύρει τον τροχό πάρα πολλές φορές σε πολλούς τομείς ε, με διαφορετικά προϊόντα είτε από κοινού με την Κομισιόν είτε όχι. Θα πρέπει λοιπόν την εμπειρία μας αυτή να την παγιώσουμε και να την συγκεντρώσουμε σε μικρά, σε μικρά τον αριθμό, ε, ολιγάριθμα τέλος πάντων ε, και σημαντικά εργαλεία στους ε, βασικούς τομείς προτεραιότητας ε, που θα είναι καταλήτες. Και έτσι και θα υποστηριχθούν οι πολιτικές αλλά και θα είναι ορατά αυτά τα εργαλεία για τους Ευρωπαίους πολίτες. Θα βλέπουν ότι αυτό το οποίο ουσιαστικά κάνουμε είναι ότι ως ε, τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχουμε μακροπρόθεσμες επενδύσεις μέσω του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού. Η Αμελή Μπαρβιέγκο Σάρ τώρα έχει το λόγο. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι σήμερα εδώ για να σας μιλήσω για την προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής, των ευρωπαϊκών δημόσιων δαπανών και επικεντρωνόμαστε στη συγκέντρωση πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Σε ένα πλαίσιο δημοσιονομικής εξυγίανσης το θέμα ε, των καλύτερων, της καλύτερης δαπάνης των δημόσιων πόρων είναι πάρα πολύ επίκαιρο, διότι η αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών καθίσταται ιδιαίτερα αναγκαία. Η συζήτηση λοιπόν που γίνεται σήμερα για το μέλλον του ευρωπαϊκού προπολογισμού δείχνει ότι το επίκεντρο πλέον είναι πώς μπορούμε μαζί να δαπανούμε καλύτερα, αλλά όχι περισσότερο. Και υπ' αυτήν την προοπτική θα πρέπει να ενισχυθεί η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση των οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που θα έδινε τη δυνατότητα να έχουμε πιο αποτελεσματικές δημόσιες δαπάνες. Αν βλέπει κανείς λοιπόν τις ε, δημόσιες υπηρεσίες, τα δημόσια αγαθά, νομίζω ότι είναι καλό ε, να συγκεντρωθούν οι πόροι γιατί αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πιο αποτελεσματική κατανομή ε, των δημόσιων πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να επιμείνω στην ανάγκη τα ευρωπαϊκά δημόσια οικονομικά να τα δούμε κάπως ομαδοποιημένα, κάπως συνολικά. Αυτό θα πει ότι θα πρέπει να τα δούμε σε κοινοτικό επίπεδο αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Να έχουμε δηλαδή μια ακριβή γνώση της κατάστασης αυτής της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης των οικονομικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να δούμε επίσης τις εθνικές πρακτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό τα ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά και υπηρεσίε μπορούν να θεωρηθούν ω δημόσια αγαθά και υπηρεσίε που παρέχονται σε κοινοτικό επίπεδο. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντε οι οποίοι επηρεάζουν ε, τη συνάφεια τη ε, συγκέντρωση, όπω είναι οι προτιμήσει ε, των πολιτών, τα spillover effects όπως λέγονται ή ακόμη δυνατότητα υλοποιηση οικονομιών κλίμακας. Από οικονομικής πλευράς, οι οικονομίες κλίμακας είναι τα πλεονεκτήματα αύξηση τη κλίμακα παραγωγή προ το κόστο, δηλαδή κόστο αναμονάδα. Τι θα πει τώρα pooling resources, η συγκέντρωση πόρων. Θα πει ότι χρηματοδοτούμε από κοινού το σύνολο ή μέρος μια συγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης. Σε αυτό το πλαίσιο η συγκέντρωση πόρων θα μπορούσε να οδηγήσει στην ε, αποκόμιση πλεονεκτημάτων από τις οικονομίες κλίμακος. Είναι ένα μέσο που θα επιτρέψει την αποτελεσματικότερη χρήση των δημόσιων πόρων. Σε ποιου τώρα τομεί πολιτική θα μπορούσαμε να σα κάνουμε αυτή τη συγκέντρωση πόρων. Θα μπορούσε να είναι οι τομεί αυτοί έρευνα και ανάπτυξη, μεταφορές, ενέργεια, ασφάλεια και άμυνα. Γιατί να επιλέξουμε αυτούς τους τομείς πολιτικής. Πρώτα απ' όλα, γιατί σημαντικές οικονομίες κλίμακας μπορούν να βρεθούν ακριβώς στην ένταση κεφαλαίου, όπως παραδείγματο χάρη, μεταφορές, ενέργεια, υποδομές. Δεύτερον, γιατί αυτοί οι τομείς πολιτικής ενθαρρύνονται και στο πλαίσιο της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020 εκτός βέβαια από την ε, ασφάλεια και άμυνα. Τρίτον, διότι για αυτούς τους τομείς πολιτικής, για ορισμένους από αυτούς, υπάρχει ήδη μη κοινοτική ευρωπαϊκή δαπάνη, ιδίως στην έρευνα και ανάπτυξη, με το Γιουρίκα και το ΕΖΟ, αλλά και στην ασφάλεια και την άμυνα με το ΟΚΑΡ. Και τέταρτον, επειδή φαίνεται ότι είναι συγκεντρωμένη, κεντρικοποιημένη η τομή αυτής για άλλα παραδείγματα στον κόσμο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης των δημόσιων οικονομικών Καναδάς, Ελβετία, μεταξύ άλλων. Τώρα, πώς έχει η κατάσταση σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των ε, ωφελών από τη συγκέντρωση πόρων. Υπάρχουν ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αρκετά παραδείγματα συγκέντρωσης πόρων. Για παράδειγμα, το ΟΚΑΡ, European Armament Organization, Ευρωπαϊκό, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εξοπλισμών, για την ε, υλοποίηση οικονομιών κλίμακας. Συνολικό κόστος ενός project όπως το Α400M είναι 4 δις ευρώ. 10 με 25% του κόστους αυτού είναι πάγια τέλη, πάγιο κόστος. αλυσίδα παραγωγής κτλ. Πάγει ο κόστος λοιπόν ανεξαρτήτως της εκάστοτε εθνικής συμμετοχής. Κατά αναλογίαν επίσης ε, είναι το κόστος αυτός ανάλογα ε, με τις συμμετέχουσες χώρες. Εάν επομιστεί αυτό το κόστος μόνο μία χώρα θα μπορούσε να φτάσει μέχρι τα 5 δις. Αλλά αν 5 χώρες συμμετέχουν ε, στο project αυτό το πάγιο κόστος μπορεί να μειωθεί στα 4 δις αναχώρα. Επίσης ε, βλέπουμε αυτή τη στιγμή τι μπορεί να γίνει σε ό,τι αφορά την ε, προσθέμενη αξία με την Notre Europe. Εγώ ε, συντονίζω μια έκθεση η οποία θα δημοσιευθεί την επόμενη άνοιξη για αυτό το θέμα και επίσης έχουμε υποβάλει μια πρόταση για ένα ερευνητικό πρόγραμμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ερευνών ώστε να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε ακριβώς ποια θα είναι τα ωφέλη από τη συγκέντρωση πόρων σε διάφορους ε, τομείς πολιτικής και για τα δημόσια οικονομικά, αλλά και για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Um, για αυτέ τι οικονομίε τις οικονομίες κλίμακα πρέπει να είμαστε και αποτελεσματικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βέβαια, για να τι επιτύχουμε. Πάμε τώρα να ακούσουμε το ελεγκτικό συνέδριο. Θα σας θέσω και εσά το ίδιο ερώτημα. Αν δηλαδή υπάρχουν ε, αλλαγές στον ε, ρόλο του ελεκτικού συνεδρίου που να θεωρείται απαραίτητες να γίνουν ε, την, στο προσεχές μέλλον. Ε, Κυρίε και κύριοι Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσω τι σκέψει μου για το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τι δαπάνε του. Καταρχήν πρέπει να πω ότι εδώ μιλώ ε, εξ ονόματο ε, δικού μου μόνο και όχι εξ ονόματο όλου του ελεγκτικού συνεδρίου. Βεβαίω, οι σκέψει μου επηρεάζονται πάντα από την εμπειρία που έχω από το ελεγκτικό συνέδριο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έναν προπολογισμό που είναι περίπου 1% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 140 ε, δισεκατομμύρια το χρόνο είναι ένα τεράστιο ποσό ε, και σε απόλυτους όρους και είναι μικρό σε σχέση με την ευρωπαϊκή οικονομία στο σύνολό της. Βέβαια πρέπει να ε, δαπανηθεί χρηστά, αλλά παρόλα αυτά η σύγκριση με άλλου προπολογισμού δίνει ένα σαφέ μήνυμα. Τα κράτη-μέλη δαπανούν 35% και άνω του ΑΕΠ ε, σε δημόσιε δραστηριότητε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δαπανίσει μόλι 1%. Το μήνυμα από, του, από τα αριθμητικά στοιχεία λοιπόν είναι ότι πρέπει να σκεφτούμε πολύ προσεκτικά το πώ θα δαπανίσουμε τα ποσά αυτά ώστε να ε, γίνει κάτι παραπάνω από μια σταγόνα στον ωκεανό. το μερίδιο που αναλογεί στην Γεωργία, δηλαδή του ΑΕΠ, έχει το στόχο να ενισχύσει την τεχνολογία, να διευκολύνει τον τομέα, να καλύψει τις ε, ε, αναταράξεις στην ε, ζήτηση που, υπάρχουν για τα αγροτικά προϊόντα, που υπάρχει για τα αγροτικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίνεται σε κατακαιρματισμένο επίπεδο προς το παρόν για να, υπάρξουν, να, μείωση, να υπάρξει μείωση των διαφοροποιήσεων από την παρέμβαση και τα κράτη-μέλη αποφασίζουν από μόνα του πώ θα δραστηριοποιηθούν με το δικό τους προπολογισμό. Βεβαίω, αυτό ε, αποτελεί έτσι μια κακοφωνία των ανταγωνιστικών εθνικών γεωργικών πολιτικών ε, και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δει κατά πόσο μπορεί να εγγυηθεί μια ισονομία. Μετά την μείωση της γεωργίας έχουμε παραμείνει με 80 δισεκατομμύρια ανά χρόνο στις δημοσιονομικές προοπτικές. Αυτό το τμήμα του προπολογισμού πρέπει να θεωρηθεί ότι δαπανήθηκε σωστά εάν μπορέσει να πάει σε γενικούς στόχους κοινού για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν μπορούμε να το διχειριστούμε σε υπερεθνικό επίπεδο. Ε, αυτό δαπανάται με τέτοιο τρόπο στο, παρα, στο παρόν δημοσιονομικό πλαίσιο. Νομίζω όχι. Γιατί ε, αρκεί να υποθέσουμε ότι αν έχουμε μόνο 1% του ΑΕΠ για να δραστηριοποιηθούμε δεν θα προσπαθήσουμε να δραστηριοποιηθούμε σε όλες τις ε, ε, δραστηριότητες ε, δημοσίων δραστηριοτήτων, όπως αν θα είχαμε πολύ μεγαλύτερο προπολογισμό υποστηρίζοντας ε, δραστηριότητε προστασία των ε, καταναλωτών ε, και προσπαθώντας να κρατήσουμε ας πούμε, τα παιδιά στο σχολείο. Από τον υποστηρίζουμε τις περιφερειακές κυβερνήσει, τα κράτη-μέλη για τις προσπάθειες που κάνουν για την ψηφιακή επικοινωνία, μέχρι να οργανώσουμε εξαρτίε κατά της υπερκατανάλωση αλκοόλ. Εγώ είμαι υπέρ όλων όσων θέλουν να έχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Επίση, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε του κανόνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχουμε ένα κοινό πεδίο για να μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε όλοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται σαφεί κανόνε για να σα δώσω ένα παράδειγμα για το πώ οι καταναλωτέ θα πρέπει να προστατεύονται. Αυτό είναι ένα θέμα που το διαπραγματεύεται καλύτερα, ε, που μάλλον είναι εύκολο να το διαπραγματευτούμε και από πλευρά οικονομική αλλά και διοικητική. Ε, τι σημαίνει αυτό Πρέπει να ε, μπούμε σε διαδικασία να το συμπληρώσουμε όλο αυτό με υποβολές προτάσεων για να μετάσχουμε σε ε, χρήματα τα οποία ούτως ή άλλως θα δίνονται. Ε, δεν, δεν νομίζω. Πολύ συχνά ε, καταλήγουμε να καταβάλουμε, καταλήγουν τα κράτη-μέλη να δαπανούν χρήματα για ε, προγράμματα τα οποία δεν είχαν θεωρήσει ότι ήταν άξια για χρηματοδότηση από το δικό τους ε, προπολογισμό. Έχουμε δύο αρχές. Να, να κάνουμε αυτά που δεν μπορούν να κάνουν τα κράτη-μέλη σε ένα υπεραθνικό επίπεδο, ε, επικουρικότητα, και να μην δαπανίσουμε τα ε, χρήματα σε ε, πολλές και μικρές δόσεις. Δηλαδή αρχή της συγκέντρωσης. Η εφαρμογή τώρα των ε, αρχών αυτών, εγώ θα ήθελα να διαχωρίσω την συνοχή ε, σε χρήματα που πάνε σε φτωχότερα κρατημέλη και σε ε, υποδομές. Το τελευταίο θα μπορούσαμε να το διαχειριστούμε καλύτερα με τις δραστηριότητες για τα διευρωπαϊκά δίκτυα που υπάρχουν. Εγώ θα έθετα ε, στόχους και θα έδινα τα, τα κονδύλια ώστε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να τα διαχειριστούν ε, μέσω των εθνικών του θερμοστικών συστημάτων και όχι το πολύ ακριβό δαπανηρό σύστημα που υπάρχει τώρα. Επίση, πέρα από τη γεωργία και την ε, συνοχή, θα είχα και ε, χρηματοδότηση της έρευνας. Ε, και γιατί είναι διεθνή από τη χρήση τη και επειδή είναι ο βασικό στόχο για την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη Λισαβόνα και την πολιτική του 2020 η Κομισιόν ε, μπορεί να ε, ε, λογοδοτήσει για πολύ λιγότερα σε ό,τι αφορά την διαχείριση και ίσως το θέμα της λογοδοσίας να, ήταν, να μπορούσαμε να το λύσουμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο βλέποντας και την εφαρμογή και την ανάλυση και τον συντονισμό των πολιτικών. Η τελευταία φράση μου τα λέει όλα νομίζω. Αν ήταν λιγότερο κατακριματισμένος ο προπολογισμός τότε και η διαχείρισή του θα ήταν σαφέστερη, θα ήταν διαφανέστερη και θα ήταν και πολύ πιο εύκολο για έναν ελεγκτή να μειώσει τους σπόρους που δαπανώνται λόγω του ότι υπάρχει, δεν υπάρχει σωστή α, διαχείριση του προπολογισμού. Η εφαρμογή λοιπόν ήταν ε, ανεπιτυχής, γι' αυτό θα πρέπει να δούμε και την ανάλυση του, α, του πώς εφαρμόζεται, πώς ε, δαπανάται ο και να την ε, βελτιώσουμε. Ευχαριστώ. Thank Κυρίες και κύριοι, καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την ευγενή ε, πρόσκληση και την εξαιρετική εισαγωγή του Φαβιάνα Τσιλέγκ. Εγώ θα μιλήσω για πέντε πράγματα. Πρώτον, η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία είναι μία από τις θεωρητικές οικονομικές βάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό να μην είναι μόνο προϋπόθεση για την τήρηση του προϋπολογισμού, αλλά να έχει κάποια ισχύ για το συντονισμό και την νομοθεσία επίσης. Τα νέα παραδείγματα είναι η ενιαία αγορά, ή η εισαγωγή του οικονομικού εξαμήνου. Δεύτερον, η... τα χρήματα που ξοδεύονται είναι πιο καλό να ξοδεύονται σε τοπικό και κρατικό επίπεδο. Ε, η δυσκολία εκπλήρωσης τώρα. Γιατί δυσκολία εκπλήρωσης. Θα αναφέρω κάποιους λόγους. Πρώτον, δεν είναι δυνατόν να διευκρινιστεί η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία χρειάζεται να αποκτήσει κάποιο πρόσωπο, ε, όπως συχνά συμβαίνει στην οικονομία βέβαια. Δεύτερον, διαφορετικοί εμπειρογνώμονες, διαφορετικά κράτη-μέλη έχουν διαφορετικές ιδέες για το ποια είναι η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και για το τι δεν συνιστά ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και τρίτον. Είναι πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς στην, στο στάδιο του προγραμματισμού την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία γιατί τα χρήματα που δαπανώνται στις επενδύσεις και στα έργα, στα προγράμματα έχουν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και είναι πολύ δύσκολη η απόδειξη και η τεκμηρίωση των μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων. Ε, ενώ στο μικροεπίπεδο είναι πολύτιμη η προστιθέμενη αξία, μακροπρόθεσμα υπάρχει πολύ θόρυβος αν θέλετε, υπάρχει ε, πολλά πράγματα αλλάζουν. Η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία λοιπόν είναι πολύ καλή στη θεωρία αλλά πολύ δύσκολη να εφαρμοστεί πρακτικά. Τι πρέπει να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Εγώ είμαι υπέρ των πρακτικών προσεγγίσεων αρκετά παρόμοιον υπό αυτή την έννοια με αυτά που ανέφερε η Αμελή Μπαγβιέ Γκοσάχ. Από την βιβλιογραφία έχω πάρει μια τυπολογία των πιθανών θεωρητικών δραστηριοτήτων που παράγονται με βάση την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Ένα. Έργα με πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα ή που έχουν ως αποτέλεσμα οικονομίες κλίμακας ή που έχουν διακρατικά αποτελέσματα ε, επενδύσεις στην ενέργεια, στη συνοχή, δίκτυα, κλιματική αλλαγή, μεταφορές κτλ. Δεύτερη πιθανότητα. έντονη δεσμή προς τα πρόσω ή προς τα πίσω, για παράδειγμα ασφάλεια των τροφίων, προστασία του περιβάλλοντος των φυσικών πόρων. Τρίτη δυνατότητα, συνέργειες για την εσωτερική αγορά. Παράδειγμα, κοινή αγροτική πολιτική, συνοχή, αριστεία στην έρευνα και άλλα. Καταλητικά αποτελέσματα ή αποτελέσματα επέκτασης, spillover, για παράδειγμα, για την ποιότητα και κινητικότητα της εργατικής δύναμης, τη διάρθρωση της αγοράς εργασίας, την εκπαίδευση, την επαιδεία κτλ. Οι εξωτερικές οικονομίες, οι πλεονάσματα, ε, μεταναστευτική πολιτική κτλ. Αυτά είναι πιθανές πηγές δημιουργίας ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας στη θεωρία. Πρέπει βέβαια να εξασφαλίσουμε ότι και στην πράξη γίνονται αυτά. Καταρχήν πρέπει να τα διασφαλίσουμε αυτά, όπως λέει και το όνομά μας. Ε, Βεβαίω οι οικονομολόγοι δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Δεν είναι βέβαιοι πώς να χρησιμοποιήσουν τη θεωρία αυτή στην πράξη. Υποθέτω ότι το ίδιο ισχύει πάνω κάτι που ανέφερε και ο κύριος Κράιενκουρ. να, να κρατάμε τα πράγματα απλά. Αυτή είναι η προσέγγιση μου. Ε, χθες κάποιος ανέφερε ότι η μόνη δυνατότητα είναι να, το κάνουμε, να καταστήσουμε τη στρατηγική της Ευρώπης το 2020 αξιόπιστη. Ε, έτσι λοιπόν το ίδιο πρέπει να κάνουμε και για την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Αν αναλύσουμε το πρόβλημα της επικουρικότητας, θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα. Πιστεύετε ότι ο κόσμος έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στους κρατικούς προϋπολογισμούς σε σχέση με τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Όχι, συνήθως ε, ο κόσμος δεν συγκρίνει τους προπολογισμού, δεν συγκρίνει τον κοινοτικό με τον εθνικό προπολογισμό. Ο κόσμος είναι ικανοποιημένος εάν κάτι βελτιωθεί ε, με βάση τη χρήση των ευρωπαϊκών πόρων. Αυτό είναι το κύριο μέλημα του απλού κόσμου και αυτό είναι και το κεντρικό μου μήνυμα. Εγώ υποστηρίζω την θέση του κυρίου Μπάρκα σήμερα το πρωί. Η τελειότητα είναι αδύνατη κατά την διάρκεια του προγραμματισμού. Αν θέλουμε να είμαστε προ... τέλειοι δεν το καταφέρουμε ποτέ. Ε, το, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα θα πρέπει να αποδεικνύεται στην πράξη, όχι στη θεωρία. Θα πρέπει να είναι μετρήσιμο. Όλα τα αποτελέσματα θα πρέπει να είναι μετρήσιμα. Γι' αυτό προτείνω να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στη μέτρηση των αποτελεσμάτων. Οι κρατικοί προϋπολογισμοί είναι πιο μεγάλοι, ο κοινοτικός προϋπολογισμός είναι πιο μικρός συγκριτικά. Εάν λοιπόν οι δαπάνες μας είναι καλά στοχευμένες μέσω και των κρατικών προϋπολογισμών, υπάρχουν, περιορίζονται οι πιθανότητες να κάνουμε μεγάλα λάθη. Και το τελευταίο σημείο, έχουμε μάθει πολλά, έχουμε πρακτική εμπειρία, πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε. Η θεωρία δεν θα μας φέρει και πολύ μακριά. Η μέτρηση των αποτελεσμάτων, η μάθηση μέσω αυτών που κάνουμε είναι τα καλύτερα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Τώρα έχουμε χρόνο για ερωτήσεις και για συζήτηση μόνο θα ήθελα να προσθέσω κάτι. Νομίζω ότι μιλήσαμε για την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και φαίνεται να έχουμε εστιάσει την προσοχή μας κυρίως στα πράγματα που θα πρέπει να κάνουμε. Αυτό που δεν έχουμε συζητήσει είναι πώς συνδέεται αυτό με την πραγματικότητα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού αυτήν τη στιγμή και ποια είναι τα πράγματα που πρέπει να περιορίσουμε στο μέλλον. Είναι μια επανερχόμενη συζήτηση αυτή για τη γεωργία, για τις δαπάνες, για τις περιφέρειες, για τις φτωχότερες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση για το κατά πόσο αυτές οι δραστηριότητες επιφέρουν όντως ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Νομίζω λοιπόν ότι τώρα μπορούμε να, έχουμε, να δεχθούμε ερωτήσεις. Ωραία. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους. Η Χέλγα Τρούπελ είναι πρώτη και μετά η Μέρη Μαγκίνες. Να ξεκινήσω με ένα πολιτικό σχόλιο και μετά θα επανέλθω στα ερωτήματά μου. Πολύ απογοητευτικό, απογοητευτικό χτες. Στο πάνελ ακούσαμε δύο μιλητές που είπαν ότι καλύτερο θα ήταν να επενδύσουμε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ειδικά σε μικρές επιχειρήσεις, γιατί αυτές είναι οι πιο καινοτόμες και βρίσκουν νέες ιδέες, νέες παραγωγές, νέες γραμμές παραγωγής, νέα προϊόντα κτλ. Το σχόλιο μου είναι ότι με τον επόμενο προπολογισμό νομίζω ότι κάνουμε το ακριβώς αντίθετο. Δεν παίρνουμε τα χρήματα που πάνε σε ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο και επενδύουμε σε ταλέντα. Παίρνουμε τα κονδύλια αυτά από την ανάπτυξη για την έρευνα για το 2012 και το 2013. Αυτό λοιπόν είναι το αντίθετο από αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε. Δεν νομίζω λοιπόν ότι ακολουθούμε τους ε, ε, εμπειρογνώμονές μας, αλλά πριν τα Χριστούγεννα θα καταλήξουμε σε μια αντίθετη τελείως απόφαση. Ερωτήματα τώρα. Δεν με ικανοποίησε η απάντηση του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για το πώς θα πρέπει να έχει η νέα προσέγγιση της ε, τράπεζας για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο για την στρατηγική 2020. Μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε λίγα περισσότερα πράγματα. Ποια θα είναι η συνέπεια των, της στρατηγικής 2020 για τα project αυτά, τα project της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Επίσης, για την ευρωπαϊκή προσθεμένη αξία και τους δείκτες. Ένας δείκτης μείωσης του ε, του άνθρακα θα πρέπει να είναι δείκτης είναι μετρήσιμα τα αποτελέσματά του. Συνδέεται με τι πολιτικέ μα ή τέλο πάντων θα έπρεπε να συνδέεται με τι πολιτικέ τι περιβαλλοντικέ. Δεν θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα δείκτη τέτοιο κατά την άποψή σα. Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Αν δείτε το πρόγραμμα Εράσμους ή την διαβίου μάθηση ή τον ε, στόχο της, ε, των διαβριζονικών δικτύων ε, στην Ήπεθρο. Φυσικά υπάρχει προστιθέμενη αξία. Ίσως να υπάρχουν και το ε, μίσο όπου υπάρχει μεγαλύτερη προσθέμενη αξία και αν μπορείτε μας λέτε εσείς. Και επίσης πρέπει να τονίσω και πάλι ότι εάν μιλούμε για τους μεγάλους στόχου, για το τι θα πρέπει να κάνουμε και ποιε θα πρέπει να είναι, θα πρέπει να είναι οι μελλοντικέ επενδύσεις μας, αυτό που συνειδητοποιώ είναι ότι ε, αναρωτιέστε, αμφισβητείτε όλε αυτέ τι μεγάλε ιδέε κατά πόσο είναι μετρήσιμε. Ίσως να είναι ένα σύμπτωμα αυτό, γιατί αν είσαστε τόσο σκεπτικοί για τις μεγάλες αυτές ιδέες και πώς μπορούν αυτές να συνδεθούν με το ευρωπαϊκό, ε, το ευρωπαϊκό επίπεδο και το εθνικό επίπεδο, Νομίζω ότι αυτή είναι η, ε, ε, η προσέγγιση των του Συμβουλίου, ε, να γίνονται δηλαδή περισσότερες δραστηριότητες διμερός και να μην ακολουθήσουμε αυτή τη γενική προσέγγιση. Θα ήθελα να μου το αιτιολογήσετε αυτό. Ευχαριστώ. Η Μέρη έχει το λόγο. Thank you very much, Chair. Uh, Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που απουσίασα χθε. Χαίρομαι που ήρθα και έφτασα και σήμερα λόγω του τσικονοφύλλας χθε στην Ιρλανδία. Γενικά το κλίμα είναι παγωμένο και για πολλούς λόγους. Όσοι εισηγήτρια για τα γεωργικά για του χρόνου θα με ενδιέφερε ε, η άποψη της εκπροσώπου του ελεγκτικού συνεδρίου για τη γεωργία. Από ό,τι νομίζω, όπως είπατε και εσείς σωστά, λάβαμε μια απόφαση. Την απόφαση να έχουμε μια κοινή γεωργική πολιτική. Αυτό δεν έχει αλλάξει η συνθήκη. Το ζήτημα τώρα του προπολογισμού δεν κατάλαβα καλά Ίσως θα μπορούσατε να το διευκρινίσετε. Είπατε ότι είναι γενναιόδωρος ο προϋπολογισμός, αλλά νομίζω ότι αμφισβητήσατε την εφαρμογή του. Κατά την άποψή μου, γενναιόδωρο δεν είναι κάτι που χαρακτηρίζει την κυνηγιορική πολιτική. Το ζήτημα της ασφάλειας των τροφίμων που ανέφερε ένας άλλος ομιλητής ήταν κάτι που ε, με ικανοποίησε, που ετέθη. Νομίζω ότι αντιμετωπίζουμε σοβαρές προκλήσεις ό,τι αφορά τους φυσικούς πόρους, περιβαλλοντική προστασία, ασφάλεια τροφίμων, παραγωγή τροφίμων. Αν δούμε όλα αυτά από οικονομικής πλευράς, χρήμα, είπε ο εισηγητής, τι μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με την ε, λιγότερο, σε σχέση με τον προπολογισμό. Εγώ θα έλεγα όχι λιγότερο, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα με τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιε είναι οι προτεραιότητέ μα. Ε, φοβούμε ότι τα τρόφιμα, η ασφάλεια των τρόφιμων, παρότι μεν συζητούνται ω προτεραιότητα, δεν έχουν ουσιαστικά ληφθεί υπόψη επαρκώς. Όταν κάποιος ε, έχει το στομάχι του γεμάτο, ε, ίσως να μην καταλαβαίνει ποια είναι τα ζητήματα με την ασφάλεια των τροφίμων. Έχουμε και τους προπολογισμού αναπτυξιακής βοήθειας. Επειδή είμαστε έτσι χορτασμένοι, ε, ίσως αυτό μας ε, κάνει λίγο να κλείνουμε τα μάτια και να μειώνουμε τους προπολογισμού και να αλλάζουμε την ε, εστίαση και το επικεντρό μας. Άρα το ερώτημα που απευθύνω στο πάνελ και ουσιαστικά είναι μια ανησυχία μου, είναι μας φοβίζει να έχουμε προπολογισμό για άλλες προτεραιότητες, γι' αυτό διαβαθμίζουμε έτσι τον προπολογισμό το γεωργικό. Και σε ό,τι αφορά τη χείριση των φυσικών πόρων, εκ με την ασφάλεια των τροφίμων, για τους Ευρωπαίους πολίτες μπορούμε να το εξασφαλίσουμε και μπορούμε βέβαια να δούμε και τις γενικότερες ανησυχίες ασφάλειας των τροφίμων εκτός από τη στόχευση αυτή μέσω του προπολογισμού μπορεί να βρεθεί ένας καλύτερος τρόπος. Έχω μελετήσει τα ε, μοντέλα. Παραδείγματος χάρη θέλουμε ένα νεοζηλανδικό μοντέλο για την Ήπεθρο και το σύστημα παραγωγής γεωργικής στην Ευρώπη. Είναι προκλήσεις αυτές. Πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά ε, αν θέλουμε να κάνουμε το σωστό. Και για τον προπολογισμό και για τη γεωργική πολιτική που είναι κοινή πολιτική αλλά και για την ευρύτερη ευρωπαϊκή κοινωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, μπήκα και εγώ στον ε, κατάλογο των ομιλητών. Χωρίς αμφιβολία την πιο ακραία θέση μας την ανέφερε η εκπρόσωπος των, ε, ε, των, του ελεκτικού συναδρίου λέγοντας ότι συνοθείτε στα σημαντικά. Και τα σημαντικά ε, εκτός από την ε, γεωργία μας είναι και η, η πολιτική συνοχής, η έρευνα αλλά πολιτική συνοχής για τους φτωχότερους των φτωχών και ταυτόχρονα συγκέντρωση εσωτερική των, ε, εντός των φτωχών χωρών για θέματα ε, αναδιάρθρωσης υποδομών κτλ. Ώστε να μπορέσουν να φτάσουν τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα υπόλοιπα, αν ακολουθήσουμε αυτή την αρχή ε, της συγκέντρωσης, όλα τα υπόλοιπα θα μπουν στην διαδικασία της επικουρικότητας. Οπότε όλα όσα κάνουμε, όσα θέλουμε να εφαρμόσουμε, όσα θέλουμε να επιτύχουμε με τους στόχους για το 2020 θα πρέπει να τα αναλάβουν τα κράτη-μέλη, να τα εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη. Αλλά αυτό θα σήμαινε ότι από τα κράτη-μέλη και από τους εθνικούς προπολογισμούς θα πήγαιναν επιδοτήσεις στις περιφέρειες. Και όταν λέω επιδοτήσεις κλείνω γιατί οι επιδοτήσεις απαγορεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση επί της αρχής. Οπότε χρειάζεται η έγκριση των αρχών ανταγωνιστικότητας, της Κομισιόν για επιδοτήσεις. Νομίζω λοιπόν ότι την νομική τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να την αλλάξουμε ώστε να μπει να λάβει τον ρόλο που της ε, αρμόζει αυτή τη στιγμή η επικουρικότητα, έτσι όπως το προτείνετε κι εσείς με την αρχή της συγκέντρωσης. Το έχετε σκεφτεί αυτό ή απλώς λέτε οι περιφέρειες θα πρέπει να, εφαρμόσουν κι αυτές την ε, ε, αρχή της επικουρικότητας και με τις δικές τους δυνάμεις μετά να ακολουθήσουν και να εφαρμόσουν τις διάφορες αρχές. Ούτως ή άλλως λέμε παντού ότι θα υπάρξουν μειωμένοι, κομμένοι προπολογισμοί. Οπότε αυτή η αρχή θα πρέπει να ισχύει από πάνω μέχρι κάτω ή θέλουμε να αλλάξουμε το δίκαιο που αφορά τις επιδοτήσεις ώστε να αλλάξουμε την κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2020 θα εφαρμοστεί με βοήθεια των κρατών μελών και μόνο εάν μπορέσουμε να δώσουμε κίνητρα στα κρατημέλη από, την, από τον προπολογισμό. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Εσείς πώς ακριβώς το έχετε σκεφτεί αυτό. Ευχαριστώ Γιούτα. Έχω και εγώ κάποια σχόλια και ένα βασικό ερώτημα. Νομίζω ότι η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία σημαίνει ότι το παιχνίδι που παίζουμε δεν είναι ένα παιχνίδι μηδενικού ποσού, αλλά είναι μια κατάσταση όπου βγαίνουν όλοι κερδισμένοι. Ότι δηλαδή κάτι καταφέρνουμε παραπάνω στο ευρωπαϊκό από ότι στο εθνικό επίπεδο. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ένα πιο μακρόπνο όραμα και μια ε, μακροπρόθεσμη σκέψη, κάτι που δεν είναι τόσο ορατό λόγω της κρίσης, λόγω των εγχώριων πολιτικών πιέσεων σε διάφορες χώρες. Χρειάζεται πάντως μια σκέψη η οποία θα υπερβαίνει απλά τα ζητήματα των εσόδων, ε, της συμμετοχής και της ισορροπίας αυτών των δύο. Νομίζω ότι είναι κάτι ε, που αναφέρατε ορισμένοι από εσάς ε, πολύ σημαντικό. Δηλαδή τα συγκεκριμένα παραδείγματα, η εφαρμογή, η εκτέλεση, ότι αυτό έχει σημασία αυτό που ο κύριος ε, Κράγενκουρ είπατε ότι τα πραγματικά καλά έργα, προγράμματα είναι αυτά τα οποία είναι καταλυτικά, αυτά που έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα, είναι αυτός ο μακροοικονομικός μηχανισμός και αύριο έχουμε μια ακρόαση για το θέμα αυτό. Η εντύπωση που έχω αποκομίσει είναι ότι αρχικά τα πράγματα και στο Συμβούλιο ήταν πάρα πολύ καλά, τώρα όμως και επειδή υποτίθεται ότι θα ήταν ένα ε, κονδύλι το οποίο θα επανερχόταν, θα επέστρεφε στα κράτη-μέλη, τώρα δεν ξέρουμε ακριβώς λόγω της, ε, του χρονικού ορίζοντα πώς θα εξελιχθεί. Υποτίθεται ότι θα ε, υπήρχαν τεράστιες επενδύσεις από τις εμπορικές τράπεζες, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική από ό,τι φαίνεται. Φοβούμαι επίσης ότι ο στόχος ήταν να προσεγγιστούν πελάτες που δεν ήταν μέχρι τότε για τη σύναψη δανείων. Και μάλλον τώρα η κατεύθυνση είναι διαφορετική. Δεν απευθυνόμαστε πια σε αυτά τα άτομα. Άρα δεν έχουμε εκπλήρωση του στόχου ανάπτυξη για όλους τα 2020, αλλά προσεγγίζονται πια οι δύσκολοι πελάτες, θα έλεγα. Ε, τέλος πάντων, αυτή είναι η εντύπωσή μου. Νομίζω ότι είναι πράγματι πολύ σημαντικά τα συγκεκριμένα παραδείγματα. Τέρο κύριο Μπέρτε ε, και η κυρία Μπαρμπιέ Γκουσάρ το ανέφερε. Κυρία Μπαρμπιέ Γκουσάρ, νομίζω ότι επεξεργάζεται μια μελέτη για τη σχέση μεταξύ κρατικών προεπολογισμών και ευρωπαϊκού προεπολογισμού. Νομίζω ότι θα ήταν πιο χρήσιμο να ακούσουμε πιο συγκεκριμένα παραδείγματα. Γιατί για να πείσουμε τα κρατημέλη και το Συμβούλιο για την πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία που υπερβαίνει απλά τα έσοδα, ε, που υπερβαίνει απλά τις εθνικές συμμετοχές, για να το κάνουμε αυτό θέλουμε καλά παραδείγματα. Δεν έχουμε ακόμη τόσο καλά πιστικά παραδείγματα. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω από εσάς παραδείγματα τα οποία θα μπορούσαμε και εμεί να αξιοποιήσουμε για να πείσουμε τα κρατημέλη και το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Θα μπορούσατε να κάνετε μια αξιολόγηση, ώστε να δούμε σε ποιο βαθμό αυτό το οποίο βλέπουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποτέλεσμα του ευρωπαϊκού προπολογισμού που είναι 1% ή είναι αποτέλεσμα το ότι είμαστε όλοι μαζί και έχουμε μια ενιαία αγορά. Όλοι βέβαια αποκομίζουμε όφελος, αλλά σε ποιο βαθμό. Γιατί η ανάλυση αυτή θα μας επιτρέψει να δούμε κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Να δούμε με νέο μάτι το προπολογισμό. Όπως δείχνουν σωματικές επιστημονικές μελέτες, τα χρήματα τα οποία δίδονται στους δικαιούχους αποφέρουν πραγματικό όφελος. Αλλά βέβαια μπορεί κανείς να δει διαφορετικά τα πράγματα. Μπορεί κανείς ε, να σκεφτεί αυτή τη ε, δημοσιονομική φιλοσοφία και σε αυτό το πλαίσιο είναι πολύ σημαντική η συζήτηση που έχουμε σήμερα εδώ. Πρέπει να δούμε ποια είναι η συσχέτιση μεταξύ προϋπολογισμών και οικονομικής κατάστασης ε, σε επίπεδο ένωσης. Και πρέπει να δούμε και τι λέει και η έκθεση για την ενιαία αγορά που λέει ότι πρέπει να υπάρξει περαιτέρω εμβάθυνση. Άρα θα πρέπει να δούμε όλες τις συσχετήσεις πολιτικές, δημοσιονομικές, φορολογικές. Μιλήσατε, κυρία Μπαρδιέ Γκοσά, για την συγκέντρωση των οικονομικών δυνατοτήτων, χρηματοπιστωτικών δυνατοτήτων. Εγώ έχω κάποια εμπειρία στη συλλογή πόρων για την ε, επιστημονική έρευνα. Θεωρείτε ότι έτσι θα αξιοποιήσουμε καλύτερα τους πόρους. Θεωρείτε ότι τα αποτελέσματα είναι καλύτερα. Πιστεύετε ότι αυτό θα γίνει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν όλα μπουν σε ένα κοινό κορβανά. Για παράδειγμα, στο δικό μου πανεπιστήμιο υπάρχουν πολλοί φοιτητέ ε, οι οποίοι κάνουν μια περίοδο άσκηση και κάποιοι από αυτού ε, δέχονται πρόταση σε μια θέση εργασία. Αν ένα άτομο, παραμείνει κάποιος, θα μπορούσαμε ίσως να κάνουμε κάποιες άλλες επενδύσεις, να χρηματοδοτήσουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, θα μπορούσε ένα πανεπιστήμιο να ζητήσει να έρθει κάποιος από την Αλοδαπή για περίοδο άσκησης ε, για ένα στάζ εδώ. Α συνενωθούν οι πόροι το πανεπιστημίων. Τώρα, σε ό,τι αφορά άλλα προγράμματα για τη Βαλτική, για το Δούναβη κτλ. μπορούμε να κάνουμε μια διαφοροποίηση των προγραμμάτων αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα πρέπει να δει κανείς ποιος είναι ο βαθμός διαφοροποίησης αυτή τη στιγμή και αν μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο ή αν μπορούμε να επεκτείνουμε τα προγράμματα σε φτωχότερε χώρες που έχουν μεγάλες ανάγκες. Και έρχομαι σε ένα άλλο ερώτημα. Τα ταμεία τα οποία θα πρέπει να διατεθούν για τη δημιουργία μιας ε, δύναμης παρέμβασης στο εξωτερικό. δυνάμεις ε, γρήγορης ε, ταχείας επέμβασης σε περίπτωση φυσική καταστροφής κτλ. Αυτό ε, υποτίθεται θα ήταν μια ιδιαίτερη αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέτοιου είδου δράσεις θα μπορούσαν να έχουν και θετικό αντίκτυπο. Πολύ πιο θετικό από το έργο το οποίο κάνουν οι χιλιάδες ευρωϊπάλληλοι. Ολοκληρώνοντας, Πιστεύετε ότι έχουμε μια καλή ανάλυση των αποτελεσμάτων έτσι αναλυτικά για να μπορέσουμε να δούμε καλύτερα προς το μέλλον σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό και σε ποιο βαθμό θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν οι εξωτερικοί και εσωτερικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Äh, Ευχαριστώ. Ο Μισελ Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Με καταπλήσει που στη συζήτηση αυτή για την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία οι διάφοροι παρεμβαίνοντες δεν τόνισαν περισσότερο την τον χαρακτηρισμό των κατηγοριών των δαπανών. Παρέμβαση εκτός μικροφώνου. Χωρίς να μιλήσουν και για τα εργαλεία δημοσιονομικής παρέμβασης ε, στον Έρασμο, στην ΚΑΠ, ο προϋπολογισμός παρεμβαίνει άμεσα, αλλά σε μια πολιτική που έχει να κάνει πιο πολύ με τις επενδύσεις, σκέφτομαι τώρα το περιβάλλον, όταν θέλουμε να επιδράσουμε στο ύδατα. Χρειαζόμαστε ε, επίσης οι μεταφορές, η ενέργεια, ε, ο τουρισμός, τα εμπορεύματα. Μιλούμε για μια υποδομή που πρέπει να διαρκέσει 30, 40, 50 χρόνια. Πρέπει λοιπόν να εξακολουθήσουμε να δρούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο με μόνο εργαλείο τη δημοσιονομική παρέμβαση όπως ξέρουμε μέχρι σήμερα. Θα αποκτήσουμε μια προστιθέμενη αξία καλύτερη εάν αφιερώσουμε ένα μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση των μεγάλων ευρωπαϊκών υποδομών που μπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη και το ΑΕΠ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Οι δικές μου σκέψεις, οι ερωτήσεις πιο πολύ έχουν να κάνουν με την παρέμβαση της ε, κυρίας, της κυρίας από το ελεκτικό συνέδριο η οποία έλεγε ότι πιστεύει ότι πρέπει ο προϋπολογισμός και οι εργασίε στο πλαίσιο του προπολογισμού να, είναι πιο συγκεντρωμένε. Θα ήθελα να ακούσω τι λένε και οι άλλοι εισηγητέ. Θα πρέπει πράγματι να επικεντρωθούμε σε δύο, τρει, τέσσερι πολιτικέ ή καλό είναι να υπάρχει και κάποια διαφοροποίηση ώστε να μπορούμε να επηρεάσουμε σε διάφορου τομεί. Διότι λαμβάνοντα υπόψη ποιο είναι το μέγεθο του ευρωπαϊκού προπολογισμού, τελικά το σημαντικό που μας ενδιαφέρει είναι πώς μπορούμε εμείς να επηρεάσουμε τα πράγματα. Άλλη ερώτηση. Πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολιτικές που χρηματοδοτούνται από το προλογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που θα έπρεπε ίσως να τις, από, ε, να τις βγάλουμε από τον προπολογισμό γιατί δεν πληρούν τους στόχους ή μήπως αντίστοιχα υπάρχουν αντίθετα μάλλον πολιτικές που πρέπει να συμπεριληφθούν, που δεν είναι τώρα μέλος στην κυρία τώρα Μπαρμπιέ Γκοσάρη, η οποία έχει κάνει νομίζω μία μελέτη για τους ίδιους πόρους, όπου διαρωτάται κατά πόσο πρέπει να αλλάξει κάτι ή να μείνουμε όπως έχουν τα πράγματα. Θα ήθελα να ακούσω τι λέει η έκθεση αυτή, ποια είναι τα πορίσματά της, αλλά θα ήθελα να ακούσω και την άποψη των εισηγητών, των υπόλοιπων μελών του πάνελ και για τον προπολογισμό όσο έχει και για το κατά πόσο θα είχαν να μας προτείνουν, εφόσον βέβαια αυτό είναι αναγκαίο, κάποιες αλλαγές. Ευχαριστώ. Ja, ähm, εγώ ευχαριστώ. Ίνια. Είναι ενδιαφέρον ότι ο εκπρόσωπο τη ε, Τράπεζα Επενδύσεων έχει επίση μια ακραία έτσι, προσέγγιση. Είπατε ότι θα πρέπει να, υπάρχουν, ε, να υπάρχει δανεισμό ο, το, για τον έλεγχο του προπολογισμού καμιά φορά έχουμε την εντύπωση ότι όντω μιλούμε α, ε, όχι για δανεισμό αλλά για κατασπατάληση. Η εμπειρία σας που έχετε από τα δημόσια ταμεία με την η μία ή την άλλη επιλογή θα μπορούσατε να, μας, ε, να τη μοιραστείτε μαζί σας. Τώρα για το μηχανισμό έχω ένα πρόβλημα για την ελληπή διαφάνεια. Ε, δεν βλέπουμε δηλαδή τι ακριβώς γίνεται και πού πάνε τα χρήματα. Θα ήταν λοιπόν απαραίτητο εάν ε, αναπτύξουμε τέτοιο μοντέλο, να δούμε πώς κυκλοφορεί το χρήμα τελικά και από πού κινείται προς τα πού. Επίσης, κάτι άλλο ενδιαφέρον που τέθηκε ήταν ένα ερώτημα. Πώς δηλαδή τα οικονομικώς αδύναμα μπορούν να ε, ε, προχωρήσουν με κάποια σημαντικά ε, οικονομικά κίνητρα. Η Ελλάδα, ας πούμε, εδώ και 30 χρόνια είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τώρα η κατάσταση είναι λυπηρή. Έχουν γίνει πολλά λάθη, αλλά τα πράγματα δεν μπορούν να συνεχίσουν όπως πήγαιναν. Ίσως λοιπόν αυτή την κρίση θα μπορούσαμε να τη δούμε σαν ευκαιρία και να τη χρησιμοποιήσουμε ως ευκαιρία. Αυτό που είναι κρίμα είναι ότι από τα κράτη-μέλη ποτέ δεν ζητούμε να, ε, ε να, να ε, στοχοθετήσουν καλύτερα την οικονομική τους πολιτική και τη φορολογική τους πολιτική με κίνητρα από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. τα κράτη-μέλη θα ήταν σκόπιμο να αλλάξουν τις οικονομικές τους πολιτικές και τις φορολογικές τους πολιτικές, να προβλέπεται ίσω αυτό μέσω του ευρωπαϊκού δικαίου. Και αν τα κράτη-μέλη που το κάνουν ε, να επιβραβεύονται, τα κράτη-μέλη που δεν το κάνουν, που δεν προχωρούν σε αναδιάρθρωση των πολιτικών του, οικονομικών και φορολογικών, να του κόβεται ας πούμε η επιδότηση, σε εισαγωγικά πάντα. Έχουμε περίπου 12 ε, ή 14 προγράμματα για τους νέους ε, και υπάρχει και ένα πάρα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον έγγραφο εργασία για την χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να λαμβάνουμε ε, συνεπείς αποφάσεις. Καλύτερα να παίρνουμε αποφάσεις για μικρή και λίγη χρηματοδότηση παρά να χρηματοδοτούμε γενικώ και μετά να μην μπορούμε να διορθώσουμε τα πράγματα. Αυτό που έκανε η Ιταλία την τελευταία ε, δημοσιονομική περίοδο, πώς θα το αποφύγουμε μια επόμενη φορά. 700.000 ε, προγράμματα χρηματοδοτήθηκαν και το, ο μέσο όρος χρηματοδότηση του καθενός ήταν 40.000 ε, ευρώ. Δηλαδή, σκεφτείτε πόσοι άνθρωποι πρέπει να τα οργανώσουν όλα αυτά, να τα ελέγξουν. και το χρήμα που κυκλοφόρησε ήταν τεράστια τα ποσά. Ε, πρέπει λοιπόν να αποφύγουμε να έχουμε τέτοιες ε, ακραίες ε, περιπτώσεις όπως αυτή της Ιταλίας, γιατί πραγματικά φοβάμαι ότι δεν πρόκειται αν συνεχίσουμε έτσι να επιτύχουμε τίποτε. Ωραία, καθόμαστε εδώ και τα συζητάμε, αλλά στο τέλος, αν δεν έχουμε μια σωστή νομική, ένα σωστό νομικό θεσμικό πλαίσιο, τότε δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Θα καταλήξουμε πάλι στην κατάσταση που είμαστε και σήμερα. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Uh, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και το μέλη του πάνελ για τις παρουσιάσεις. Έχω την αίσθηση μερικές φορές ότι αυτούς τους στόχους ε, της Ευρώπης το 2020 δεν τους παίρνουμε και τόσο σοβαρά. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δούμε Πώς θα αποφύγουμε μια κατάσταση που το 2020 θα πούμε «Ωραία ήταν οι στόχοι, αλλά τελικά δεν τους καταφέραμε». Δεν είδα στα μέλη του πάνελ να υπάρχει έτσι και μια συνέστηση της επίγουσας φύσης ε, των παρεμβάσεων που πρέπει να κάνουμε. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων αν μιλούμε για την εκπλήρωση αυτών των στόχων, ο σύνδεσμος μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού έχει ζωτική σημασία και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είναι ζωτικός. Καταρχήν, ένα σαφές ερώτημα είναι πώς θα διασφαλίσουμε σωστό βαθμό συνοχής μεταξύ των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, πολύ, σημαντική, φορέα ως φορέα χορήγησης δανείων, και από την άλλη πώς θα ικανοποιηθούν αυτά τα κριτήρια για την εκπλήρωση των στόχων του 2020 να αποφύγουμε το να κάνουμε πάλι λάθη στην Ευρώπη. Από την άλλη πλευρά, όταν κοιτούμε τις, δημοτικές και, τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Υπάρχουν πολιτικά ζητήματα. Πιστεύετε ότι υπάρχουν προγράμματα που τα επιδοτούμε αυτή τη στιγμή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με δημόσιες δαπάνες που έχουν τέτοιο βαθμό απόδοση που δεν έχει νόημα να τα κάνουμε με κρατικές δαπάνες. Θα ήταν καλύτερο να έχει γίνει με ιδιωτικέ επενδύσεις. Ο προπολογισμό μας είναι ισχνό. Μπορούμε λοιπόν να είμαστε πιο αποτελεσματικοί ε, αναθέτοντας τον ιδιωτικό τομέα να κάνει τις επενδύσεις που έχουν πολύ υψηλό βαθμό αποδόσεων. Ένα Κάτι ακόμα για την σύνδεση δημόσιο-ιδιωτικού. Μιλούμε για δεκαετίες, εντάξει. Αν δούμε όμως το πρόγραμμα Γαλιλαίο, και εκεί η πρόθεση ήταν ότι κάποια στιγμή θα μπουν μέσα οι ιδιωτικές επενδύσεις. Ωστόσο, μέχρι στιγμής στο Γαλιλαίο έχουμε εξ ολοκλήρου δημόσιες δαπάνες. Πώς θα μπουν οι ιδιωτικοί επενδυτές σε αυτά τα προγράμματα, ακόμα δεν μου έχει καταστεί σαφές αν δεν, είμαστε, αν δεν τα καταφέρουμε σε ένα πρόγραμμα όπως το Γαλιλαίο να επιτύχουμε τη σύζευξη δημόσιου και ιδιωτικού, τότε πώς περιμένουμε στο μέλλον να έχουμε τέτοιο μείγμα. Αν εντάξουμε πολλές δημόσιες επενδύσεις και στο τέλος το πρόγραμμα γίνει επικερδές και στο τέλος μόνο έρθουν μέσα οι ιδιώτες και τελικά εκείνοι αποκομίσουν όλα τα κέρδη, τότε δεν θα υπάρχει καμιά απόδοση για το δημόσιο. Γιατί αν ξεκινούμε βάζοντας όλα τα έξοδα εμείς από το δημόσιο τομέα και μόνο στο τέλος προσελκύσουμε τους ιδεώτες και αποκομίσουν εκείνοι όλα τα ωφέλη, τότε τι γίνεται. Νομίζω ότι αυτά τα θέματα πρέπει να επιληθούν. Διαφορετικά το 2020 θα πούμε πολύ ωραία ήταν όλα αυτά, αλλά για άλλη μια φορά δεν τα καταφέραμε. Χωσέ Μανουέλ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Μιλούμε για την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και για την αποτελεσματικότητα, αλλά πρέπει να γίνει λόγος και για αλληλεγγύη. Και ερωτώ, ε, το Ταμείο Αλληλεγγύης έχει προστιθέμενη αξία Όλα αυτά βασίζονται στην αρχή της αλληλεγγύης. Αυτή είναι η ουσία της ερώτησής μου. Η Ευρωπαϊκή Δράση για τη Στρατηγική 2020. Όλες αυτές οι δράσεις έχουν ως στόχο τη συγκεκριμενοποίηση των πέντε στόχων της στρατηγικής για την Ευρώπη το 2020. Ερωτώ, εάν δεν υπάρχει και εδώ μια ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Τι γίνεται, θα την έχουν εν τέλει, θα την προσφέρουν εν τέλει. Τι, να, μας να, να έχουμε κάποια παραδείγματα για τα προγράμματα που θα χρηματοδοτήσουμε στο επόμενο πολιετές χρηματοοικονομικό πλαίσιο, δημοσιονομικό πλαίσιο, ως συμπλήρωμα αυτού του πλαισίου. Τι μπορούμε να έχουμε. Ja, Ευχαριστώ. Δεν έχουμε άλλα ερωτήματα, οπότε να δώσουμε και πάλι το λόγο στο συντονιστή. Ευχαριστώ. Να κάνω και εγώ κάποια σχόλια και μετά θα δώσουμε το λόγο στους ομιλητές. Ένα από τα σημεία που προέκυψε από τις διάφορες ερωτήσεις δεν είναι μόνο το θέμα της προσθέμενης αξίας, αλλά και της ε, ε, και προτεραιοτήτων. Είμαστε σε μια πολύ περιοριστική περίοδο. Δεν μπορούμε να τα χρηματοδοτήσουμε όλα όσα θα θέλαμε. Οπότε πρέπει να αποφασίσουμε τι κριτήρια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να θέσουμε σωστά τις προτεραιότητες χρηματοδότησης. Βεβαίως θα πρέπει να έχουμε ως στόχο ότι όλα τα χρήματα που θα έχουν την προτεραιότητα θα έχουν και προσθεμένη αξία, αλλά πρέπει να πω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Πολλά πράγματα έχουν προστιθέμενη αξία. Πρέπει λοιπόν να θέσουμε σωστέ προτεραιότητε. Η Ευρωπαϊκή ε, ε, Πολιτική 2020 είναι η ευκαιρία μα για να θέσουμε προτεραιότητε στον προπολογισμό και μετά πρέπει να αναρωτηθούμε εάν όλα αυτά που λέμε όντω συμβάλλουν στην πολιτική για το 2020. Μερικέ φορέ, στι συζητήσει αυτέ που γίνονται ε, δείχνει, δείχνουν ότι ε, όλα, τα, όλα τα projects έχουν μια αλφα συμβολή στο 2020. Αλλά θα πρέπει να ρωτηθούμε αν αυτό είναι που θέλουμε να κάνουμε. Δεύτερον, για, τις, για τους ίδιους πόρους που αναφέρθηκαν. Να είναι σαφήτατα για το πώς θα λειτουργήσουν οι ίδιοι πόροι. Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ ιδίων πόρων ως μηχανισμός ε, εσόδων Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίων πόρων ως μέσω επίτευξης στόχων, ως πολιτικού εργαλείου δηλαδή. Μπορεί όντω να πρέπει να δούμε κατά πόσο χρειάζεται μεγαλύτερο εύρος εργαλείων για να επιτύχουμε τους στόχους του 2020. Αυτό που πρέπει λοιπόν να κάνουμε είναι να καθορίσουμε καταρχάς ποιες είναι οι καλύτερες πολιτικές που μπορούν να επιτύχουν τους στόχους του 2020 και μετά να συζητήσουμε τα εργαλεία. Ε, συνήθως το κάνουμε ανάποδα. Τρίτον, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ότι δεν αρκεί να κατανέμουμε ε, κονδύλια σε συγκεκριμένους τομείς που μπορεί να υποσχόνται προσθέμενη αξία. Αυτά τα χρήματα θα πρέπει όντως να είναι και αποτελεσματικά και ξέρουμε ότι σε πολλούς τομείς έχουν υπάρξει προβλήματα με, την, με τα αποτελέσματα. Οπότε δεν είναι, απλό το θέμα, δεν είναι το θέμα μόνο να έχουμε διαθέσιμα χρήματα. Το θέμα είναι να είναι σαφές και να υπάρχει τρόπος να ελέγξουμε ότι τα χρήματα αυτά θα επιτύχουν αυτά που πρέπει όντως να επιτύχουν. Και επειδή το είπα και στα εισαγωγικά μου σχόλια για την ε, βοήθεια των ε, πλέον αδυνάμων ε, οικονομιών της Ευρώπης, νομίζω ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα θα είναι ένας τρόπος για να βοηθήσουμε τέτοιες χώρες όπου υπάρχει ελάχιστη εσωτερική ζήτηση, ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε μεγάλης κλίμακας ε, προγράμματα υποδομών ε, διευρωπαϊκής ε, σημασίας, να ενισχύσουμε τη ζήτηση, την πρόσβαση στην προσφορά και πρέπει επίσης να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια αυτά για να ε, επενδύσουμε σε παράγοντες ανάπτυξης. Αυτούς δηλαδή που ζητά και η πολιτική 2020. Ειδικά σε χώρες όπου ο εσωτερικός τους, ο δικός τους προπολογισμό είναι αδύναμος και δεν μπορούν από μόνος τους να τα καταφέρουν. Ας πούμε, εκπαίδευση, καινοτομία. Ξέρουμε ότι ένας αριθμός χωρών ήδη αρχίζουν να κόβουν προγράμματα σε αυτούς τους τομείς λόγω των περιορισμών του προπολογισμού τους αντί να επενδύουν σε μελλοντική ανάπτυξη. Αυτά έτσι εισαγωγικά. Τέθηκαν αρκετά ερωτήματα για όλα τα μέλη του πάνελ. Να ξεκινήσουμε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να εξηγήσετε και εσείς το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και να απαντήσετε και στα υπόλοιπα ερωτήματα για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο μέλλον. <clears throat> Um, Ευχαριστώ. Πράγματι υπήρχαν αρκετά ερωτήματα αλλά νομίζω ότι μπορώ να τα συνοψίσω υπό πέντε θέματα. Πρώτον, ποιο τομέα παρέμβασης, ποιος ουσιαστικό τομέα για τη δραστηριότητα επί της οποίας έχει έλεγχο η ΕΤΕΠ και ποια είναι, η προτεραιότητα, ποια είναι η προτεραιότητά μας για τη στρατηγική 2020. Δεν το ανέφερα, πράγματι είναι πολύ σημαντικό. Δεν το ανέφερα γιατί το θεώρησα δεδομένο. Πάντα είναι λάθος να παίρνει κανείς κάτι ως δεδομένο. Όπως γνωρίζετε, μέτοχοί μας ε, είναι τα κράτη-μέλη και το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αυτό το οποίο θέτει τις προτεραιότητες και το οποίο απαρτίζεται από προσώπους ε, των κρατομελών και της Κομισιόν. Και πρέπει να σας πω ότι η τρέχουσα ανάλυση του εταιρικού μας σχεδίου για το μέλλον ε, έχει σαφώς ευθυγραμμιστεί πάνω στους στόχους της Στρατικής Ευρώπη 2020. Οι προτεραιότητες της τράπεζας είναι έξι επιχειρησιακές προτεραιότητες. Συνοχή, έρευνα και καινοτομία, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, περιβάλλον, ενέργεια και τη ευρωπαϊκά δίκτυα. Όλα αυτά μπορείτε να τα ομαδοποιήσετε πάρα πολύ εύκολα στους τρεις αυτούς τομείς ε, της εφιούς, της πράσινης και της ανάπτυξης για όλους. Νομίζω ότι όλοι είμαστε στην ίδια γραμμή και μας παρακολουθούν. Θέλουν να βλέπουν ότι είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Σε ό,τι αφορά τώρα την ερώτηση για τις μικροπιστώσεις και τα καλά παραδείγματα. Ερώτηση της κυρίας Γκέντς. Δεν θέλω να επισέλθω στο θέμα των μικροπιστώσεων, αλλά αυτό που είπατε ότι ε, πρέπει να έχει χαρακτήρα επιστροφή στα κράτη-μέλη, αυτό είναι σαφές ο ορισμός του ευρωπαϊκού προπολογισμού λέει ότι δεν θα πρέπει ένα μέσο να επιστραφεί πέραν της περίοδου δημοσιονομικής προοπτικής. Άρα αυτό σημαίνει ότι για πολύ μακροχρόνιες επενδύσεις υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει ακόμη επιληθεί. Τώρα το πώ θα επιληθεί δεν είναι δική μου δουλειά να το πω. Εμείς έχουμε αυτόν τον περιορισμό στην ε, τράπεζα, ότι αντιμετωπίζουμε κάποιες φορές αυτή τη δυσκολία με κάποια μέσα, με κάποιους μηχανισμούς. Ό,τι αφορά τώρα το καταλητικό αποτέλεσμα, τον καταλητικό ρόλο, πρέπει να σας πω ότι αυτή η πρωτοβουλία για τις μικροπιστώσει είναι εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αντιδιαστολή μετά εκτός, είναι ένα εντελώς καινούριο σύστημα. Και πρέπει να μάθουμε, ε, θα έλεγα στο κασίτι του κεφάλι κατά κάποιο τρόπο. Και έχουμε εταίρους οι οποίοι είναι έτοιμοι να συνεργαστούν μαζί μας και φαντάζομαι ότι και άλλοι θα ενθαρρυνθούν από τα αποτελέσματα τα οποία θα έχουμε να τους επιδείξουμε. Κάτι θέλει κάποιος να έχει ως αποτέλεσμα πριν προσχωρήσει, πριν ενταχθεί. Έτσι προσελκύουμε τους εταίρους. Υπάρχουν όμως καλά παραδείγματα ε, κάποιοι ίσως να γνωρίζετε το project Marguerite, Μαργαρίτα. Ένα equity fund για υποδομές, το οποίο έχουμε με έξι σημαντικούς ε, χρηματοπιστωτικούς φόρους ε, από τη Γαλλία, από την Ιταλία, από την Πολωνία, από την Ισπανία. Συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υποστηρίζουμε τις υποδομές ε, με επενδύσεις κεφαλαίων. Εκεί έχουμε καταλητικά αποτελέσματα. Υπάρχει ε, και άλλο πρόγραμμα όπως το Green for Growth. Αλλά δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες. Τώρα έρχομαι στην κυρία Γκρέσλε. Ελπίζω να μην είπα ότι είναι χάσιμο ε, χρημάτων ή επιδοτήσεις. Εγώ είπα ότι θα μπορούσε να είναι εάν δεν εφαρμοστεί σωστά η διάθεσή τους. Και αυτό είναι αλήθεια οι επιδοτήσει είναι και παραμένουν απαραίτητε. και κάθε φορά που στηρίζουν ε, δημόσιου στόχου και δεν έχουν μια τυπική επιστροφή, τυπική απόδοση και θα επανέλθω στον Καλλιλέο, θα είναι απαραίτητε αυτέ οι επιχορηγήσει. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ της εφαρμογής των ε, επιδοτήσεων όπου είναι αυτό απαραίτητο και του επιχείρηματος που εξέφρασα εγώ ότι αν δεν είναι βιώσιμη η επένδυση ως οικονομικό προϊόν τότε μπορεί να είναι περιτές διαφάνεια. Εγώ δεν συμφωνώ. Κάθε δικαιούχος επενδύσεων μέσω αυτού του μηχανισμού risk sharing, ε, του μερισμού κινδύνων, διαδημοσιεύεται στην ισοσελίδα και τίθεται προς έγκριση των διαφόρων φορέων της Κομισιόν στην προκειμένη περίπτωση. Ίσως απαιτείται καλύτερη ενημέρωση Πάντως θεωρώ ότι είναι ένα ιδιαίτερα διαφανές σύστημα, μια διαφανής προσέγγιση. Σε ό,τι αφορά τα PPPs, θα σας μιλήσω και για τα ομόλογα για δημόσια έργα. Όταν κάποιος προσπαθεί να ε, βάλει όλους τους κινδύνους στο ιδιωτικό τομέα, δεν θα τους ε, δεχθεί ο ιδιωτικός τομέας, εκτός αν υπάρχουν βέβαια επαρκή κέρδη για να εξορροπήσουν. Άρα σε αυτά τα PPPs, τις συμπράξεις ε, δημόσιο-ιδιωτικού τομέα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είπατε κάτι για τον Καλλιλέο. Το πρόγραμμα είναι ότι τα έσοδα είναι ακαθόριστα και άγνωστα αυτή τη στιγμή. κάποια στιγμή ίσως το ξαναδούμε και τότε και ίσως και ο ιδιωτικό τομέας θα μπορέσει να ενταχθεί. Αλλά στην αρχή νομίζω ότι χρειάζεται ένας δημόσιος στόχος για μια τέτοια επένδυση. Είναι τυπική περίπτωση. Για τα ομόλογα για δημόσια έργα, αυτό το οποίο συνέβη το εξής. Η αγορά ε, για, το δημόσιο, για τον ιδιωτικό τομέα, για τη χρηματοδότηση. Υπήρχε και πριν από την κρίση, αλλά η αγορά αυτή ουσιαστικά καταστράφηκε από την κρίση. Αυτή είναι η πραγματικότητα και υπάρχουν τεράστιες ρευστότητες. Υπάρχει ρευστότητα διαθέσιμη στους θεσμικούς επενδυτές, τα εξοδοτικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείε. Οι θεσμικοί επενδυτές έχουν χρήματα γιατί υπάρχουν ψηλά ποσοστά ε, αποταμίευσης, αλλά μπορούν να επενδύσουν μόνο σε ορισμένα εργαλεία και μέσα χαμηλού κινδύνου και μακράς ε, περίοδου ισχύω. Μακροπρόθεσμες υποδομές λοιπόν, για να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει μακροχρόνια πίστη υπό τη μορφή ομολόγων ή δανείων. Αυτό είναι και τα project loans για επέκταση, ουσιαστικά βελτίωση της πίστης. Δηλαδή υπάρχει μια πρώτη δόση, υπάρχει ένα ανώτατο όριο βέβαια, εκεί, ισοδύναμο σε ένα είδος κεφαλαίου, ώστε οι πρώτες όλες αν υπάρχουν να απορροφηθούν. Από το μερίδιο αυτό, τη δόση αυτή του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Και μετά υπάρχουν κάποια υπαγόμενα δάνεια, που είναι το δεύτερο, η δεύτερη δόση, το, το δεύτερο τμήμα που αν αυτά πληγούν από μια δεύτερη δέσμη δυσκολιών, το μεγάλο ποσό, που δεν μπορώ να σας βάλω ένα ποσοστό, εξαρτάται από το κάθε project, η χρηματοδότηση να μπορεί να παρασχεθεί στη συνέχεια από τον ιδιωτικό τομέα που μορφήν ομολόγων με αρκετά υψηλή ε, πίστη ώστε να μπορούν να επενδύσουν. Αυτό έκαναν και κάποιες ασφαλιστικές εταιρείε πριν την κρίση, αλλά εγκαταλείφθηκε λόγω της κρίσης. Και τώρα η διαφορά είναι ότι τέτοιου είδους ε, εγχειρήματα δεν θα γίνονται ε, εκτός ε, ισολογισμών, αλλά πάνω στον ισολογισμό, με τον ισολογισμό. Θα είναι διαφανής δηλαδή οι διαδικασίε αυτέ. Είναι τεχνικό το ζήτημα και δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειε, αλλά πιστεύουμε ότι η προσέγγιση αυτή πραγματικά μπορεί να βοηθήσει, μπορεί να κινητοποιήσει την ελκυστικότητα της χρηματοδότησης υποδομών από τον ιδιωτικό τομέα. Μιλάμε για μεταφορές, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες. Και επιμένω, γιατί τελικά αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι ότι αυτά τα ομόλογα θα εκδίδονται από τους εργολάβους, από τους κυρίους του έργου, όχι από την ΕΤΕΠ ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε από το πληθυσμό, ούτε από τίποτα. Το σχέδιο είναι αυτό το οποίο επενδύει. Οι εταιρείε που επενδύουν στο σχέδιο είναι αυτέ οι οποίε εκδίδουν τα ομόλογα. Εντάξει, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αλλιώ πέφτουμε σε μια άλλη κατηγορία. Ε, πολύ γνωστών πολιτικών θεμάτων. Thank you very much. Um, Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία μπαγδιεγκο Μπαγδιέγκο-Σάγα. Αναφέραστε στα... Είπατε κάποια γενικά σχόλια για το πού πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο, πού να εστιάσουμε λιγότερο. Θα ήθελα να επανέλθω στο επίκεντρο αυτής της προβληματικής στην ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία των ευρωπαϊκών δαπανών. Ποιο είναι το καλύτερο μερίδιο των χρηματικών ροών στα διάφορα επίπεδα, κοινοτικό, κρατικό, τοπική αυτοδιοίκηση. Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό θα έπρεπε να έχουμε μια συγκεκριμένη γνώση της κατανομής καθηκόντων μεταξύ των διαφόρων επιπέδων. Η πραγματικότητα πολύ απέχει από αυτό. Δεν έχουμε συγκεκριμένη γνώση. Ε, κάποτε είχαμε την πρωτοβουλία να κάνουμε μια στρατηγική ανάλυση για να μάθουμε ποιος κάνει τι στις διάφορους τομείς της πολιτικής. Ξεκινήσαμε κάποιες εργασίες, τις οποίες παρουσιάσαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που μας επιφύλαξε μια πολύ θερμή υποδοχή. Προσπαθήσαμε λοιπόν να δούμε ποια είναι αυτή η κατανομή των καθηκόντων. Ε, συνεχίζουμε να το κάνουμε αυτό για να μπορέσουμε να δούμε πού πραγματικά έγκυται η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Πρέπει να έχουμε λοιπόν μια σαφή άποψη του ποιος κάνει τι. Το παράδειγμα του έρασμος. Ο Υπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ε, ανέθεσε, μας ανέθεσε μια μελέτη για το πρόγραμμα Έρασμος για να δούμε τι παραπάνω, τι πρόσθετο παρέχει η Ευρώπη. Και ε, παρατηρήσαμε, όχι με μεγάλη έκπληξη, ότι από το σύνολο των πόρων που διοχετεύθηκε στην κινητικότητα των νέων στην Ευρώπη, το 70% ε, ε, χορηγήθηκε από την τοπική αυτοδιοίκηση. Το κονδύλιο του έρασμος είναι σχετικά χαμηλό. Δεν επιτρέπει σε έναν φοιτητή να ζήσει πραγματικά σε μια άλλη χώρα και γι' αυτό συχνά η τοπική αυτοδιοίκηση αυτοδιοίκηση προσθέτει ένα συμπλήρωμα που επιτρέπει στον φοιτητή να μπορέσει να ζήσει και να φοιτήσει σε μια άλλη χώρα. Ε, αυτό είναι τμήμα της κατανομής των πόρων. Λοιπόν, αυτό το 70% τι δείχνει. Δείχνει ότι πρέπει να έχουμε μια συγκεκριμένη εικόνα για το ποιος κάνει τι στους διάφορους τομείς δημόσιας παρέμβασης, μόνο που τα δεδομένα, τα ταστητικά στοιχεία που έρχονται μέσω της ε, Ευρωστάτ, που βασίζονται στα στοιχεία που διαβιβάζουν τα κράτη-μέλη, δεν είναι αρκετά συγκεκριμένα. Και έτσι λοιπόν ε, βλέπω πόσο επίγον και επιτακτικό είναι να γίνουμε πραγματικά επιχειρησιακοί και να, να κάνουμε πραγματιστικές προτάσεις, ρεαλιστικές προτάσεις. Για να το κάνουμε αυτό όμως πρέπει να έχουμε σαφή εικόνα του καταμερισμού καθηκόντων. Και εδώ έρχεται η αρχή της επικουρικότητας. Ε, όταν τα πράγματα μπορούν να εκτιληχθούν καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να αναλάβει το εκάστοτε δημόσιο καθήκον. Αλλά η λύση δεν είναι η πλήρη συγκέντρωση. Σκέφτομαι για παράδειγμα το θέμα των μεταφορών. Για τις μεταφορές ε, είναι ένα παράδειγμα ε, στο οποίο μπορούν να επιτευχθούν σημαντικές οικονομίες κλίμακας. Ένα τμήμα των ε, δαπανών παρέχεται κεντρικά, μόνο που οι μεταφορές δεν είναι μόνο υποδομή, είναι επίσης συντήρηση, είναι έρευνα και ανάπτυξη. Πρέπει να μπορέσουμε να, διακρίσουμε, να διακρίνουμε ποιοι τομεί πραγματικά παρέχουν αυτή την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Το ίδιο ισχύει και για τι ενεργειακέ υποδομέ για να, να, εντοπίσουμε τον τομέα που είναι πρόδειλη η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, να τον απομονώσουμε τον τομέα για κάθε πολιτική. Είτε μιλούμε για ενέργεια, είτε για μεταφορές, είτε για έρευνα και ανάπτυξη. Νομι... Ποιο ήταν το τελευταίο, η άμυνα, η άμυνα και η ασφάλεια. Και εκεί πρέπει πραγματικά να κάνουμε να είμαστε ακριβείς. Ακριβείς ως προς τις δαπάνες που δίνονται στις διάφορες πτυχές της ε, δημόσιας πολιτικής. Η αλήθεια είναι όμως ότι η πρώτη ύλη μας είναι η στατιστική. Αλλά δεν είναι ε, αυτονόητο ότι υπάρχουν τόσο συγκεκριμένα στοιχεία στατιστικά. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να, μας ε, να διαβιβάζουν γενικά πιο συγκεκριμένα στοιχεία για τη σύνθεση του προϋπολογισμού, για τις εθνικές πραγματικότητες για τις προτιμήσεις έτσι ώστε το ευρωπαϊκό επίπεδο να μπορέσει ε, πραγματικά να βασιστεί στις πιο σωστές πληροφορίες ώστε να προτείνει λύσεις οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις εθνικές ιδιαιτερότητες. Το να έχουμε λοιπόν συγκεκριμένες πληροφορίες για τις τομείς της δημόσιας πολιτικής είναι ανικαία προϋπόθεση ώστε να μπορέσουμε κάποια στιγμή να προτείνουμε πρακτικές και επιχειρησιακές λύσεις. Μεταξύ των τομέων που σας παρουσίασα, η οπτική μας είναι να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας. Ας δούμε λοιπόν πώς θα παροτρύνουμε τα κράτη-μέλη να κάνουν περισσότερα πράγματα. Ε, το πρώτο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους δείξουμε ότι με τη σωστή παρέμβαση ο καθένας μπορεί να κάνει οικονομίες κλίμακος. Και επομένως, ε, όσο πιο πολλές ε, χώρες συμμετέχουν, τόσο περισσότερο το κόστος διαμοιράζεται και επιτυγχάνονται αυτές οι οικονομίες κλίμακας. Αυτό όμως που πρέπει πραγματικά να διακρίνουμε είναι οι υποτομείς της ε, δημόσιας πολιτικής όπου μπορούμε να προσφέρουμε αυτήν την προστιθέμενη αξία και σε αυτό έγκυται και όλος ο κίνδυνος. Αυτή την ικανότητα πραγματικά να απομονώνουμε εκείνους τους τομείς όπου είναι πιο έντονη και ισχυρή η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Μιλήσαμε βέβαια για αυτή την οικονομία κλίμακος, υπάρχει όμως και τα εξωτερικά οικονομικά στοιχεία, τα externalities, υπάρχουν ε, τα θέματα της διασυνοριακής ε, συμμετοχή τα θέματα της διακυβέρνησης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο. Πραγματικά όμως, για να είναι κανείς επιχειρησιακός, αποδοτικός, πρέπει να μπορεί να είναι ακριβής. Ε, για παράδειγμα, στην άμυνα έχουμε τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Έγινε μία μελέτη για τις δαπάνες που είχαν χαρακτηριστεί ως μη κοινοτικέ αλλά ευρωπαϊκές. Στον τομέα έρευνα και ανάπτυξη αλλά και στον τομέα της άμυνας υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη που ήδη συνεργάζονται γιατί έχουν συνειδητοποιήσει τις οικονομίες κλίμακος που επιτυγχάνονται. Πρέπει πραγματικά τώρα να κάνουμε αυτή την εργασία ακριβίας και να δούμε ε, πού είναι εκεί που μπορούμε να έχουμε πιο έντονη προστιθέμενη αξία. Πρέπει λοιπόν να μπορούμε να γνωρίσουμε σε επίπεδο μεγάλης ακρίβειας τον προϋπολο... τους εθνικούς προϋπολογισμούς με τις υποδιαιρέσεις τους. Υπήρχαν και κάποια ερωτήματα για εσάς, για την ακραία σας ε, προσέγγιση. Να προσθέσω όμως και εγώ κάτι. Όταν ε, κάνατε τα σας σχόλια, ε, ήταν σαν να είπατε ότι η Γεωργία έχει προστιθέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ούτως ή άλλως ρυθμίζεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε αναρωτιέμαι Ε, ενσυνείδητα εξαιρέσατε τη γεωργία από την ε, δραστική αυτή προσέγγιση που ακολουθήσατε. Ευχαριστώ. Όντως, θα ξεκινήσω με την ε, γεωργία και θα ξεκινήσω απαντώντας στο δικό σας ερώτημα. Η γεωργία είναι λίγο διαφορετικός τομέας όταν μιλούμε για την προστιθέμενη αξία γιατί ουσιαστικά δεν ε, ψάχνουμε να βρούμε προστιθέμενη αξία γιατί έχει εκχωρηθεί από τον, Ευρωπαϊ... από τον εθνικό προπολογισμό στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Οπότε οι διάφορες γεωργικές πολιτικές των διαφόρων κρατών μελών δεν έχουν στρεβλωτικές επιπτώσεις στον, ε, στην ευρωπαϊκό προπολογισμό γιατί μιλούμε για κοινή αγορά. Είναι λοιπόν μια κοινή πολιτική. Οπότε ούτως ή άλλως προσθέτει αξία η γεωργία, ο τομέας γεωργίας. Τώρα, για την ε, ασφάλεια τροφίμων. Ε, ε, στην ομιλία μου στην αρχή έκανα μια, ένα παραλληλισμό για την ενίσχυση των α, α, τομέων αυτών ώστε να ενισχυθεί η ζήτηση, να, υπάρξουν, να υπάρξει εξορόψη των ανισορροπιών Ούτως ή άλλως τώρα έχουμε σχηδείς στόχους. Και για την ε, γενεοδορία έχω δει κάποια παραδείγματα όπου όντω υπάρχει χώρος για βελτίωση το Κοινοβούλιο προσπαθεί με το δικό του τρόπο να αντιμετωπίσει τα προβλήματα, είτε μιλούμε για μεγάλους παραγωγούς, είτε μιλούμε για παγκόσμιες ε, εταιρείες γεωργικές οι οποίες ε, θέλουν να εξασφαλίσουν ε, κάποια εχέγγυα, ώστε να μην έχουμε μόνο γη και τεχνολογία, αλλά να έχουμε και ανθρώπινο δυναμικό, γιατί αυτό είναι που μας εξασφαλίζει χρειάζονται, είτε είναι μεγάλη η παραγωγή είτε είναι μικρή παραγωγή. Χρειάζεται ανθρώπινο δυναμικό για να καλλιεργηθεί η γη που θα παραμείνουν εκεί επί τόπου για να υπάρξει παραγωγή η οποία παραγωγή έρχεται από διάφορες, ε, από διάφορες περιφέρειες της ε, Ευρώπης ή των χωρών. Το δηλαδή το εύρος και ο περιορισμός ε, είναι ένα θέμα, ναι, αυτό θα πρέπει να το, να το δούμε. Όπως στην, ενέργεια, στην παραγωγή ενέργειας έχουμε την ε, δυνατότητα παραγωγής και έχουμε και την ενέργεια. Οπότε αποσυνδέουμε. Τώρα πώς θα αναλύσουμε τις συνέπειες αυτών των δράσεων, δηλαδή ποιος είναι ο στόχος των τοπικών κυβερνήσεων που δημιουργούν οι κοινοτικές εταιρείες, και παίρνουν υποστήριξη για την ε, γη που έχουν για την ε, χρηματοδότηση ε, των, της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ούτως ή άλλως αυτό δεν έχει να κάνει με την γεωργία και δεν χρειάζεται να έχει να κάνει με τη γεωργία. Και το λέει και η Κομισιόν αυτό. Η γη διατηρείται σε μια καλή κατάσταση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αλλά με το ανθρώπινο δυναμικό και την τεχνολογία τι γίνεται δεν ξέρω μήπως είμαστε πολύ ε, γενναιόδοροι προς τις εταιρείε που δεν έχουν καμία σχέση με τη γεωργία. Επίσης, η διασταυρώμενη συμμόρφωση, η πολλαπλή συμμόρφωση. Εάν ε, έχετε ε, αγροτικές δραστηριότητες συμμορφούμενες προς το περιβάλλον, όλα καλά. Μιλούμε δηλαδή για πολύ μικρά ποσοστά, 1%, 2%, 5%, οπότε δεν έχουν επιπτώσεις στην ε, πολλαπλή συμμόρφωση. Οπότε μπορούμε να δεχτούμε την πολλαπλή συμμόρφωση. Αυτά νομίζω για τη Γεωργία. Α, και ένα ακόμη. Ίσως να είναι πολύ ιδεαλιστικό βέβαια αυτό για το δικό σας προπολογισμό, αλλά οι αγορές για γεωργικά προϊόντα δεν μειώνουν τις ε, τιμές, πολλές φορές αυξάνουν τις ε, τιμές και καλό θα ήταν να ε, δημιουργήσουμε ε, έτσι μια δυνατότητα ενίσχυσης. Όταν ας πούμε αυξάνεται η τιμή ενισχύεται η ενίσχυση. Ενισχύεται η επιδότηση, συγγνώμη. Τώρα για τις υποδομές και τα σχετικά προγράμματα και πώς αυτά μπορούν να συνδεθούν με τις δαπάνες για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Χρειαζόμαστε ενέργεια, ηλιακή, υδροελεκτρική, χρειαζόμαστε δρόμους, χρειαζόμαστε μεταφορές, χρειαζόμαστε καθαρούς ποταμούς. Όλα αυτά γίνονται στα πλαίσια της, ε, της πολιτικής συνοχής και είναι υπερεθνικοί οι στόχοι που έχουν τεθεί. Οπότε θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτά τα προγράμματα θα τα διαχειριζόμαστε σε κεντρικό επίπεδο και θα θεωρούνται προγράμματα άμεσης διαχείρισης. Τώρα, το catching up. Έχουμε περιφέρειες πλούσια κρατημέλη που πρέπει να έρθουν να προχωρήσουν και υπάρχουν και κάποια άλλα κρατημέλη τα οποία είναι πιο φτωχά και είναι λίγο πιο πίσω στην σειρά. Μια χώρα όμως που έχει μικρό μερίδιο, που παίρνει μικρό μερίδιο από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό μπορεί να έχει τον ελεκτικό μηχανισμό, τον, την ε, ενδιάμεση αρχή, την ε, ε, διαχειριστική αρχή. Γιατί το δέχεται. Υπάρχει μεγάλο διοικητικό άχθος και μπορεί να τύχει και μεγάλη κριτική και από το Κοινοβούλιο και από το Ελεκτικό Συνέδριο. Αξίζει τον κόπο να το κάνει. Δηλαδή, αν δείτε το κόστο και την ωφέλεια, ίσω καμιά φορά να μην είναι ε, σκόπιμο να δαπανηθούν αυτά τα χρήματα. Για τα φτωχά τώρα κρατημέλη, και το κατά πόσο αυτά μπορούν ακόμη να χρησιμοποιούν αυτή την αρχιτεκτονική ή την οικονομική που προβλέπεται από, το, κεντρικά, από την κεντρική διοίκηση. Να χρησιμοποιείτε τα, ε, τα χρήματα της, ε, του ευρωπαϊκού προπολογισμού μέσω των δικών σας συστημάτων εφαρμογής. Έχουμε κάποιου κανόνες που είναι οι βασικοί κανόνες που διέπουν την ε, σωστή χρηστή διαχείριση των, ε, των ε, κονδυλίων για τη συνοχή και τα οποία είναι πάνω κάτω λίγο πολύ εναρμονισμένα. αυτοί οι κανόνες είναι παρόμοιοι σε διάφορα κράτη-μέλη με τους Ευρωπαϊκού. Οπότε γιατί δεν καθόμαστε μαζί με ένα κράτος μέλος που πρόκειται να λάβει αυτά τα χρήματα για να ανακάμψει από την πολιτική συνοχή και να πούμε θέλουμε συγκεκριμένα μέτρα, περίληψη των νέων ε, ανθρώπων, από, λιγότερο, από θέλουμε λιγότερη εγκληματικότητα σε αυτέ τι ε, περιοχέ και συμφωνούμε για στόχου. Οπότε δίνονται τα χρήματα στα, ε, στα κρατημέλη. Ένα, για να σας πω ένα παράδειγμα. Ένας ε, δάσκαλος από μια φτωχή περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μου είπε «Μπορώ να κάνω τρία σεμινάρια το χρόνο στην περιφέρειά μας για να αναλύσω το πρόβλημα. Γιατί, α πούμε, τα παιδιά δεν πάνε σε μαθήματα γυμναστική, γιατί δεν πάνε σε μαθήματα μουσική, γιατί είναι στου δρόμου και γιατί υπάρχει εγκληματικότητα. Και γιατί αυτά τα παιδιά σταματάνε το σχολείο μπορώ να κάνω αυτά τα σεμινάρια και όλα είναι ωραία και νόμιμα, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν μέτρα αυστηρότητας τώρα. Ακόμη όμως και πριν ο προπολογισμό μας δεν ήταν τόσο μεγάλος ώστε να υπάρχει άμεση ενίσχυση αυτών των μαθητών για τέτοιου είδους ε, ε, μαθήματα. Η Ευρωπαϊκή, ο Ευρωπαϊκός προπολογισμό δεν μπορεί να μας δώσει ε, την, τέτοια υποστήριξη. Όχι, δεν μπορούμε ευρωπαϊκά να στηρίξουμε τέτοιου είδους δράσεις. Αν είσαστε έξυπνοι μπορεί να πείτε ναι θα κάνουμε μια πιλωτική ανάλυση, ένα τέτοιο πρόγραμμα και με κάποιο τρόπο θα βρείτε ένα παραθυράκι. Γιατί όμω να συμβαίνει όλο αυτό. Δεν θα ήταν πολύ πιο απλά τα πράγματα αν είχαμε συγκεκριμένου στόχου για, για κράτη-μέλη, για περιφέρειες και να δίδονται κατευθείαν τα χρήματα. Γιατί όχι. Η λογοδοσία παραμένει. Αλλά τουλάχιστον μπορούμε να ελέγξουμε του στόχου. Και κατά πάσα πιθανότητα χρειάζεται και μια καταρχητική ημερομηνία. Να πούμε, ναι, ωραία, έχετε, έχετε δίκιο, έχετε κάποιες δημοσιονομικές προπτικές, δύο-τρεις ας πούμε, για να, για να ανακάμψετε. Αν δεν τα καταφέρετε, λυπούμεθα. Δίνουμε δηλαδή ένα χρονικό περιθώριο. Είναι διαφορετικό, είναι πολύ ιδεολογικό αυτό που σας λέω. Αλλά ξέρω ότι αυτό το κοινοβούλιο ήταν ε, πολύ, ε, δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένο με την ε, μεικτή διαχείριση. Γιατί μιλούμε για, για κόστος ε, ε, και καθυστερήσεις, για κόστος ελέγχου, για κόστος εφαρμογή για καθυστερήσει σε όλο αυτό το σύστημα. Ναι, προφανώς. Το έχω σκεφτεί λοιπόν. Επίσης, τα χρήματα από την ε, συνοχή δεν είναι πολύ ευέλικτα για να λάβουν υπόψη και τι μακροοικονομικές πτυχές. Πρόσφατα μίλησα με συναδέλφου από την Γενική Διεύθυνση ε, Ρίτζο και, είπαν, και μου είπαν ότι όντω έχει δημιουργηθεί πληθωρισμό στα κρατημέλη. Ειδικά στα χαμηλά εισοδήματα που έχουν ε, όμως μια αγορά εργασίας η οποία έχει μια δυνατότητα ανάπτυξης 3-4%. Αλλά πρέπει να αυτό να γίνει τώρα, δεν μπορεί να μπει μετά, αργότερα, μέσα στον, σε αυτόν τον κύκλο, γιατί χάνεται το τρένο. Και μετά δεν μπορούμε να μιλάμε για αποπληθωρισμό. Υπάρχουν και τα κριτήρια του Μάστριχτ πρέπει να είμαστε σε, ε, σε συγκεκριμένα όρια για το έλλειμμα, για το χρέος. Τι γίνεται τώρα όμως, πρέπει να αγγίθουμε τη συγχρηματοδότηση. Ξεπεράσατε δηλαδή εσείς από μόνοι σας τους προπολογισμού σας και τις δαπάνες. Έχετε ένα εξαιρετικό εργαλείο για να φροντίσετε ας πούμε τους ηλικιωμένους που δεν το έχει ξαναδεί καμιά χώρα αλλά δεν υπάρχει το, το προσωπικό για να φροντίσει αυτούς τους ανθρώπους γιατί το, ο μισθό του κόπηκε σε τέτοιο βαθμό από το Υπουργείο Εσωτερικών και Κοινωνική Πρόνοια που έφυγαν οι άνθρωποι αυτοί από τη χώρα αυτή και πήγανε κάπου αλλού να βρουν δουλειά. Επίση, ένα ερώτημα για το αν κάποιοι τομεί πολιτική μπορούν να αφαιρεθούν. Το θέμα είναι πού πρέπει να διαχειριστούμε και πού πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένα projects. Πολλές, ε, υπάρχουν πολλοί τομείς ε, εκπαίδευση, ηθαγένεια, πολιτισμός μπορούν να τύχουν τέτοιας ε, χρηματοδότησης. Ας πούμε μπορούν να δοθούν πολύ ε, μικρές δόσεις. Υπάρχει λοιπόν περιθώριο εδώ για δράση. Επίσης το, το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση και τη αλληλεγγύη για τα κρατη που αντιμετωπίζουν φυσικές καταστροφές. Η ασφάλεια είναι το θέμα εδώ και δεν χρειάζεται να είναι τμήμα του προπολογισμού. Αν δεν είμαστε ε, ικανοποιημένοι από την, ε, από την αγορά ασφάλειας, ε, των ασφαλιών, ωραία. Αλλά γιατί να συνεχίσουμε να διατηρούμε ένα σύστημα το οποίο δεν λειτουργεί, εμένα με ξεπερνάει, δεν το καταλαβαίνω. Για την έρευνα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα χρήματα θα πρέπει να είναι ελεύθερα, να ρέουν. Και εδώ πάλι τίθεται το ερώτημα, έκαναν αυτό που πρέπει να κάνουν. Να έχουμε ένα σύστημα επιδοτήσεων που βλέπουμε μέσω κάποιων κριτηρίων τα αποτελέσματα. Που πάνε στους ερευνητικούς οργανισμούς. ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε περιθώριο και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στα πανεπιστήμια να έχουν τη δυνατότητα του opt-in. Και κάτι τελευταίο για τις ε, ε συμπράξεις ιδιωτικού και, ε, και δημοσίου τομέα, για τον Γαλιλαίο. Ο Γαλιλαίο δεν ήταν εμπορεύσιμος στη φάση που ήταν όταν προτάθηκε να τεθεί σε εφαρμογή. Ε, υπήρξε μια πρόταση να αναλυθεί από μια ε, ιδιωτική εταιρεία. Και μόνο αναλύοντας λίγο καλύτερα πού ακριβώς πρέπει να απευθυνθεί αυτή η εταιρική σχέση μπορεί να προκύψει για η κατάσταση όπου για ένα τομέα της, ε, για ένα κομμάτι της επένδυσής σας μπορεί μια ιδιωτική εταιρεία να αναλάβει. Ο Γαλιλαίο νομίζω ότι θα πρέπει εδώ να θεωρηθεί ως ένα αρνητικό παράδειγμα. Χρειάζεται περισσότερη ε, ανάλυση για το πότε και ποια χρονική στιγμή μπορούμε να ξεκινήσουμε μια εταιρική σχέση ιδιωτικού και δημοσίου. Άντρες είδα ότι ένευε καταφατικά σε κάποια από τα σχόλια. Ναι, πράγματι. Πρώτα απ' όλα να το πω ότι συμφωνώ 100% με τα φανταστικά παραδείγματα που ανέφερε. Αυτό ακριβώ ενώσα και εγώ όταν μίλησα πριν. Απεσιόδοξος είμαι μόνο υπό την εξή έννοια. Η οικονομική θεωρία μπορεί να ε, αποφασίσει για το πώ θα προγραμματιστεί ο προπολογισμό Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρουμε πάντως πώς μπορεί να γίνει να υπάρχει αποτελεσματικότητα. Δεν ξέρω τώρα ποιο είναι το πασιστό, νομίζω ίσως είναι το 70% ε, που έχουμε τα πρακτικά, την πρακτική εφαρμογή. Είμαι αισιόδοξο και γιατί υπάρχει η πρακτική εμπειρία. Συμφωνώ επίσης για τη ε, διαβίου μάθηση, δίκτία δίκτυα, έρασμος, επενδύσεις στη συνοχή, ή στην προστασία του περιβάλλοντος, ε, επενδύσεις στην ε, προστασία των τροφίμων, στην ασφάλεια των τροφίμων και στην κοινή γεωργική πολιτική κτλ. Ε, στην Ουγγαρία έχουμε πάρα πολύ καλά παραδείγματα. Πριν από κάποιους μήνες πήγα σε μια γεωργική εκμετάλλευση που ίσως να είναι πιο σύγχρονη από οποιαδήποτε αμερικανική αντίστοιχη. Έχουμε δει επίσης ε, πολλές επενδύσεις σε αυτοκινητόδρομους και σε άλλα στοιχεία. Επίσης μοκλέψαμε πάρα πολλές ιδιωτικές επενδύσεις σε τομείς που ε, ήταν υποβαθμισμένοι κατά το παρελθόν. Άρα πραγματικά είμαι αισιόδοξο. υπό αυτήν την έννοια. Αλλά τονίζω ότι είναι πολύ σημαντική πρακτική εφαρμογή ο Φάμπιαν μας ε, είπε να πούμε προτεραιότητες, ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Δική μου προτεραιότητα, μάλλον τρεις θα αναφέρω. Πρώτον, χρειάζεται πολιτική βούληση για να τα καταφέρουμε καλύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό νομίζω είναι η σημαντικότερη προτεραιότητα, κατ' εμέ τουλάχιστον. Δεύτερη προτεραιότητα. Πρακτική αποτελεσματικότητα. Θεωρώ ότι είναι το βασικό στοιχείο. Δηλαδή, διαρθρωτικές αλλαγές προς ευφυή, βιώσιμη ανάπτυξη για όλους για να υποστηριχθούν οι στόχοι της στρατηγικής 2020 και θα πρέπει να συμπεριληφθούν όλα τα στοιχεία των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη προτεραιότητα, η αύξηση του μεριδίου όλων των πόρων. Νομίζω ότι αυτό χρειάζεται. Ένας πιο ευέλικτος ε, προϋπολογισμός ε, με βιώσιμα κεφάλαια. Και βέβαια σίγουρα νομίζω ότι πρέπει να αναδιαρθρωθεί ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Λέω συντονιστής, δυστυχώς μας τελειώνει ο χρόνος. Ακούστηκαν πολλά ενδιαφέροντα ερωτήματα στο πάνελ αυτό. Ετέθησαν ενδιαφέροντα ζητήματα. Ίσως να μην δώσαμε τόσες απαντήσεις όσες ε, θα θέλατε. Και γι' αυτό ε, δύο λόγοι ε, είναι οι βασικοί. Πρώτα απ' όλα γιατί νομίζω ότι τελικά εναπόκειται στις πολιτικές διαδικασίες. Αυτή η διαδικασία είναι που θα ιεραρχήσει τις προτεραιότητες. Δεν είναι δουλειά των οικονομολόγων. Εμείς δεν παίρνουμε τέτοιες αποφάσεις, μπορούμε ίσως να σας ε, μεταφέρουμε τις σκέψεις μας για το τι θεωρούμε πιο πολύτιμο, για το τι θεωρούμε ότι μπορεί να λειτουργήσει πιο καλά ως εργαλείο, αλλά τελικά είναι πολιτική η απόφαση της ιεράρχησης των προτεραιοτήτων του προπολογισμού και του καθορισμού των στόχων που εσείς, τα κράτη-μέλη, οι πολιτικοί θέλουν να υπάρξουν. Δεύτερος λόγος, συχνά στη συζήτηση που κάνουμε τα μέσα και, τα, και οι στόχοι συγχέονται μεταξύ τους. Και νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Πρώτον, να καθορίζουμε τους στόχους μας, τι θέλουμε και δεύτερον, να αποφασίζουμε ποια μέσα, ποια εργαλεία πολιτικής μπορούν να φέρουν τα πιο επιθυμητά αποτελέσματα σε περιφερειακό, εθνικό επίπεδο. Πολλές φορές πρώτα συζητάμε τα μέσα και τις διαδικασίες, ίσως αποκλειστικά και μόνο αυτά και δεν έχουμε συζήτηση για τους επιδιωκόμενους στόχους ή αυτή η συζήτηση έρχεται σε μεταγενέστερο στάδιο. Νομίζω όμως ότι και πάλι οι πολιτικοί είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να αποφασίσουν πρώτα απ' όλα για του στόχους και έπειτα εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε λέγοντα πώ μπορούν να επιτευχθούν αυτοί. Με αυτές, τις, κουβέντε σα ε, σας δίνω πάλι την Προεδρία, αλλά να ευχαριστήσω πρώτα όλα τα μέλη του πάνελ για τις πολύ ενδιαφέρουσες ε, παρεμβάσεις τους ε, που μας έδωσαν ε, λαβή για συζήτηση και σίγουρα κάποιες από αυτές ήταν ε, και αντικρόμες μεταξύ τους. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και εγώ όλους τους εμπειρογνώμονες που ήρθαν σήμερα και χτες. Όλους όσους είναι εδώ, τα καταληκτικά μου σχόλια είναι τα εξής. Μόνο Το μόνο σημαντικό είναι ότι αυτό που, λένε, αυτό που είπε μάλλον η εκπρόσωπος από το ε, συνέδριο είναι ελκυστικό γιατί είμαστε Ευρωπαίοι βουλευτές, ευρωβουλευτές που προσπαθούμε πολλές φορές να πείσουμε τους εθνικούς βουλευτές, τις κυβερνήσεις και ξέρετε πόσο δύσκολο είναι αυτό πολλές φορές. Εγώ ευχαρίστως θα προέβλεπα σε κράτη-μέλη πώς θα κάνουν, πώς θα διαμορφώσουν τις δομές τους, τις υποδομές τους για να επιτύχουν τους στόχους που θέτουμε, για να, πώς θα οργανωθούν και τι θα γίνει. Πώς δηλαδή μπορούν κάποια πράγματα να τα εφαρμόσουν. Αλλά η κοινοτική προσέγγιση είναι η προσέγγιση του Κοινοβουλίου προφανώς, αλλά ε, στο να είμαστε τόσο κοντά στο να τα καταφέρουμε, δεν έχουμε φτάσει ακόμα. Κάτι άλλο τώρα, ότι η, η τελειότητα σε ένα τέτοιο μακρόπνο σχέδιο δεν είναι εφικτή, το προσυπογράφω. Προσπαθήσαμε να είμαστε τέλειοι με, την, ε, με το χρηματοοικονομικό μας πρόγραμμα, κάναμε ό,τι μπορούσαμε στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, αλλά όπως είδαμε ε, δεν ήμασταν καθόλου κοντά στην τελειότητα. Έπρεπε να ξαναοργανώσουμε τα σχέδιά μας, έπρεπε να αλλάξουμε τα πράγματα. Οπότε Πρέπει να εκπονήσουμε νέε κατευθυντήρε γραμμές, να βρούμε νέα σχέδια, να κάνουμε μια αξιολόγηση που να αξίζει να λέγεται αξιολόγηση, να έχουμε συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία θα συμφωνήσουμε μεταξύ μας. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι δεν είδαμε μόνο τις δομές της ε, του οίκου μας, πώς δηλαδή θέλουμε να, είπα, να είναι οι επόμενες ε, ε, εσωτερικές, ε, δημοσιομικές προοπτικές, αλλά είδαμε και τον ιστορικό μας κανονισμό. Να δούμε δηλαδή πώς, τι γίνεται με το πρόγραμμα δαπανών μας, τι γίνεται με τους κανόνες που έχουμε για το πρόγραμμα δαπανών και τι κάνουμε όταν θέλουμε να ενσωματώσουμε αυτά τα rewarding funds όπως λέγονται και πώς μπορούμε να αλλάξουμε τους, καταλό... τους ε, κανόνες μας. Αλλά επίσης πρέπει να δούμε πόσο ψηλά, πόσο μεγάλη ευελιξία θέλουμε να έχουμε, όπως ας πούμε σε αυτό, αυτό που συμβαίνει στην ε, Γεωργία, στον τομέα της Γεωργίας. Τι γίνεται, όπως το είπε και η κυρία Λάιτ, τι γίνεται όταν πέφτουν οι τιμές για το γάλα. Δεν θα έπρεπε να ενισχύσουμε τους ε, γαλακτοπαραγωγούς. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κανέναν κανόνα που να το επιτρέπει αυτό. Και αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε. Ξέρω ότι έχουμε το ταμείο, αλλά... Σχόλια εκτός μικροφώνου από τον κύριο Μπέγκε. αν θέλουμε να, πρέπει, αν θέλουμε να προχωρήσουμε, πρέπει να σκεφτούμε και εκτός των δημοσιονομικών προοπτικών. Επίσης, σαφές ήταν ότι χωρίς τον προπολογισμό τον ευρωπαϊκό δεν θα επιτυχάναμε τους στόχους που έχουμε για το 2020. Ναι, είναι μικρός ο προπολογισμό του, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1% δηλαδή του ΑΕΠ, αλλά δεν είναι συμβολικός. Η Ευρώπη πρέπει να δώσει την κατεύθυνση και τα κράτη-μέλη πρέπει να ακολουθήσουν. Οπότε πάλι είμαστε στην κοινοτική μέθοδο και είμαστε πάλι στο πεδίο του τι κάνουμε εμείς ως ευρωβουλευτές. Και το τελευταίο είναι ότι ε, επί τη βάση των ε, ε, εγγράφων στοχασμού είναι ότι προκύπτει ότι πρέπει να υπάρξει μια συγκεκριμένη προσέγγιση. είπαμε για το έξυπνο, για, το, για, το, βιώσιμο και για το συμπεριληπτικό. Ε, δεν μπορούμε όμως αυτά να τα διαχωρίσουμε, πρέπει να τα δούμε από κοινού. Έχουμε δηλαδή έναν, αν, ένα, αν έχουμε ένα στόχο που προχωράει σε μια, άλλη, σε μια πολιτική, δεν σημαίνει ότι ξεχνάμε όλους τους υπόλοιπους. Τα βλέπουμε όλα μαζί. Νομίζω ότι Α, ναι, ναι. Ε, είδα την ώρα και ε, δεν, ε, δεν είδα καθόλου το Σαλβαδόρ. Αντί να... έπρεπε να μιλήσει πριν από μένα βέβαια. Γιατί πρέπει και ο εισηγητής να κάνει τα σχολιά του. Σαλβαδόρ, λυπάμαι, το κάνουμε λίγο ανάποδα τώρα. Ε, εγώ ε, ανέφερα τα συμπεράσματα, εν πάση περιπτώσει αυτά ήταν τα δικά μου τα συμπεράσματα, τώρα μπορείς να πεις και εσύ τα δικά σου συμπεράσματα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. αλλά θα μπορούσαν να είναι συμπεράσματα ε, τα δικά σας. Εγώ δύο λεπτά έχω στη διάθεσή μου, μπορώ να είμαι πολύ πιο σύντομος. Θέλω να ευχαριστήσω τις δύο ε, ομάδες, τα δύο πάνελ που μίλησαν για τόσο σημαντικά ζητήματα. Κάποια ευθυγραμμίζονται, ευθυγραμμίζονται με τα έγγραφα προβληματισμού που έχουμε υποβάλει, κάποια όχι. Απλά εγώ, σε σχέση με το πρώτο πάνελ, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι γενικό, δηλαδή η οικονομική κρίση πρέπει να ενισχύσει την πολιτική συνοχής, διότι είναι σαφές ε, ότι Υπάρχει ένα χάσμα σε ό,τι αφορά τη σύγκληση μεταξύ των κρατών μελών, το οποίο αντί να μειώνεται, αυξάνεται, επειδή βρισκόμαστε εν καιρό Αυτή είναι η πρώτη από τις ανησυχίε. Και εν συνεχεία είναι ότι οι εισηγητέ θεωρούν ότι η πολιτική συνοχή θα έπρεπε να εννοηθεί ως οριζόντιο εργαλείο. Ότι η πολιτική συνοχή ε, θα πρέπει να τροποποιηθεί σημαντικά ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει ε, ή τέλος πάντων να επιτύχει τους στόχους της ε, στρατηγικής Ευρώπη 2020 και δεν τους φαίνεται ιδιαίτερα ελκυστική ιδέα υποδιέρεσης των ε, υφισταμένων κατηγοριών σε συνάρτηση με τα διαφορετικά είδη ανάπτυξη. Κάποιοι μάλιστα αυτά τα τρία είδη τα ονόμασαν σλόγγαν. Τέλο πάντων, εγώ θεωρώ ότι είναι κάτι πιο βαθύ από σλόγγαν, αλλά λαμβάνω υπόψη τι παρατηρήσει σα. Είναι σαφές ότι το επίπεδο διακυβέρνησης στα διάφορα επίπεδα το οποίο προβληματίζει ε, τους διάφορους πανελίστες όπως και εμάς άλλωστε. Συμφωνούμε απόλυτα με τις έννοιες ε, περί προϋποθέσεων ε, και προσανατολισμού της πολιτικής συνοχής αποτελέσματα, ενώ σε ό,τι αφορά τη διάρκεια και τη δομή, εμείς οι εισηγητές της Επιτροπής ΣΟΥΡ έχουμε αυτό το πρόβλημα, ότι τελικά πρέπει να προτείνουμε μία δομή στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. Και από ό,τι φαίνεται μάλλον είμαστε περισσότερο υπέρ μιας πολύ πιο περιοριστικής πρότασης σε σχέση με την αρχική που ήταν η πρόταση υποδιέρεσης των κατηγοριών με βάση την ε, κατανομή της στρατηγικής 2020. Γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν επαρκείς πόρη στον κοινωτικό προϋπολογισμό για την εφαρμογή μιας τόσο φιλόδοξης στρατηγικής και αυτό το οποίο με εκπλήσει είναι ότι με εξαίρεση τον τελευταίο μιλητή του τελευταίου πάνελ κανείς δεν αναφέρθηκε στην ευελιξία, στο ζήτημα της ευελιξίας που για το κοινοβούλιο ε, έχει πρωταρχική σημασία αν θέλουμε να έχουμε δημοσιονομικές προοπτικές που θα είναι προσαρμοσμένες ανα πάσα στιγμή στην πραγματικότητα. Σε ό,τι αφορά τώρα το δεύτερο πάνελ για την ευρωπαϊκή προστεθέμενη αξία. Ξέρετε ότι ήδη έχουμε εκπονήσει ένα έγγραφο προβληματισμού και μετά και ένα έγγραφο εργασίας το οποίο περιλαμβάνει και τις περισσότερες από τις υποδείξεις των εμπειρογνωμόνων. Ευτυχώς. Φυσικά και θα λάβουμε υπόψη αυτό που, αυτά που είπαν και στα συμπεράσματα της έκθεσης. Πάντως κάποιες από τις ε, απόψεις και ερωτήσεις Νομίζω ότι αν τις περιλάβω στα καταληκτικά συμπεράσματα της έκθεσής μου, ε, θα μου τις στήσουν ε, μπαίνοντα στο κοινοβούλιο κάποιοι συνάδελφοι. Ε, τι κίνητρο θα έχουν τα κράτη-μέλη όταν έχουμε μια τόσο σοβαρή δημοσιονομική κρίση για να συνεισφέρουν πόρους στο κοινοτικό προπολογισμό όταν τα θύματα, τα βασικά θα είναι η κοινή γεωργική πολιτική και πολιτική συνοχής. Βέβαια, όπως και να έχει, εμείς ε, συμφωνούμε με τα κόνσεπτ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και φυσικά κάθε πρόταση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τις νέες πηγές χρηματοδότησης που προτείνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και βέβαια θα πρέπει να υπάρξει συγκέντρωση. Συγκέντρωση των πόρων στις πολιτικές εκείνε που δίνουν μεγαλύτερη προσθέμενη αξία. Και αυτή η μεγαλύτερη προσθέμενη αξία πρέπει να εννοηθεί όχι μόνο με αυστηροοικονομική έννοια, αυστηρά οικονομική έννοια, αλλά ε, θα πρέπει να εφαρμοστεί η αρχή της προστιθέμενης αξίας σε όλες τις πολιτικές. Και ίσως με μείωση στόχων, με μείωση έργων. Έχουμε τους πέντε στόχους της στρατηγικής 2020. Δεν είναι φυσιολογικό ένα κράτος μέλλον να έχει 700.000 σχέδια ή όπως λένε οι Financial Times μόνο το 10% όλων των διαρθρωτικών πόρων αυτής της περίοδου προγραμματισμού τελικά να μην έχει ακόμη καταβληθεί είναι προφανέ ότι πρέπει να γίνουν κάποιε μεταρρυθμίσει. γι' αυτό θα στηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε ό,τι αφορά το σχέδιο μεταρρύθμιση τη κοινή γεωργική πολιτική όσο και σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση τη πολιτική συνοχή. Θέλω να ευχαριστήσω τους ε, ομιλητέ των πάνελ, γιατί πραγματικά οι παρεμβάσει του νομίζω ότι θα κάνουν το έγγραφό μα πολύ πιο ρεαλιστικό και προσγειωμένο στην πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Ε, ε, Εγώ ευχαριστώ, Σαλβαδόρ. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που ήταν εδώ δύο μέρες σήμερα, που άκουσαν με ενδιαφέρον όσα είπαν οι εμπειρογνώμονές μας. Ευχαριστώ και όλους όσους υπηρεσιακά έπρεπε να είναι εδώ ή από ενδιαφέρον έφτασαν εδώ και που κράτησαν σημειώσεις. Ευχαριστώ και όλους τους εμπειρογνώμονές μας. Καλή σας όρεξη!